Συνάδελφοι, έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Espen Barth Aid, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Νορβηγίας, σχετικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον Απότατο Βορρά. Μέρο τη Επιτροπή μα. να καλωσορίσω τον Υπουργό και τον κύριο Γκάλαγκερ, ο οποίος είναι μέλος της, ε, είναι πρόεδρος της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κύριε Υπουργέ, πριν από κάποιο διάστημα με τον κύριο Στόρ, τον προκάτοχό σα, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Για θέματα που μα απασχολούν και εσά και εμά. Τι διμερεί μα σχέσει, τι εξελίξει στην Μέση Ανατολή και τον απότατο Βορρά. Για να αναφέρω μόνον ορισμένα σημεία. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μας περιουσιάσετε σύντομα τις, τις δικές σας απόψεις για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας και τα θέματα που μόλις ανέφερα. Σας δίνω αμέσως τον λόγο. Thank you. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Προβέρα. Και καταρχάς επιτρέψτε με να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίδεται να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και προοπτικές μαζί για τα τρία θέματα που αναφέρατε, την κατάσταση Μέση Ανατολή μετά τη χθεσινή συνεδρίαση στην Επιτροπή Ad Hoc, η Επιτροπή Δωρετών για την Παλαιστινική Αρχή, ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωση και την Αρκτική. Με αυτή τη σειρά ε, θα το κάνω γιατί ίσως το πιο επίκαιρο ήταν η χτεσινή μα συνεδρίαση εδώ στι Βρυξέλλε. Όπω θα θυμάστε από πέρυσι όσοι ήσασταν παρόντες, η Νορβηγία προεδρεύει ε, στην Επιτροπή που συντονίζει την διεθνή υποστήριξη για του παλαιστινίου και τη διαδικασία ε, ATLC, Ad Hoc Liaison Committee λέγεται, ε, Ad Hoc βέβαια για τα τελευταία 20 χρόνια για τη σύσταση του Παλαιστινιακού κράτους, πάρα πολύ εύστοχος ο τίτλος. Στόχος της Επιτροπής Δωρητών ήταν να υποστηριχθεί η ε, πολιτική διευθέτηση του Παλαιστινιακού να δημιουργηθούν δύο έτη. Ε, το 1993 ε, είχε ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία πριν από 20 έτη. Η ιδέα ήταν και παραμένει πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εφόσον περιμένουμε την πολιτική λύση, τα μεγάλα θέματα της διαπραγματεύσης, δηλαδή με ποιο τρόπο το Ισραήλ και η Παλαιστίνη μπορούν να συμβιώνουν ε, δημοκρατικά, ειρηνικά, ανεξάρτητα δύο ανεξάρτητα κράτη που να συμβιώνουν πλάι-πλάι. Αρχίσαμε να ε, βοηθούμε στη σύσταση των θεσμών στην Παλαιστίνη, από κάτω προς τα πάνω. Αυτό ήταν ο στόχος της Επιτροπής. Η Νορβηγία όλη αυτή την περίοδο είναι πρόεδρος μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες ως συμπροέδρους και είπα ότι εκπρόσωπος η κυρία Κάθριν Άστον εχθές ε, υποδέχτηκε τη ε, συνεδρίαση και μέλη εκεί είναι ε, τα ενεχόμενα μέρη βεβαίως, η Παλαιστινιακή Αρχή, ο κύριος Σαλάμ Φαγιάτ, πρωθυπουργός στο Ισραήλ και όλοι οι δωρητές που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή καθ' αυτή, αλλά και κράτη-μέλη της, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, και διάφορες αραβικές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, άλλα κράτη του Περσικού κόλπου κλπ. Είναι μια ευρεία λοιπόν διεθνή συμμαχία κρατών που εργάζεται προς την υποστήριξη και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, το 2011, ακριβώς πριν από δύο χρόνια περίπου, επετεύχθη συμφωνία στην Επιτροπή αυτή και οι δωρητέ συμφώνησαν, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, τα ενεχόμενα μέρη και ο ΙΕ, που έλεγαν ότι οι Παλαιστινιακοί θεσμοί είχαν οριμάσει αρκετά ω θεσμοί ε, και ήταν συμβατοί με ένα ε, κράτος σε εύρυθμη λειτουργία. Βέβαια, ενώ λοιπόν δεν υπάρχει κράτος, υπήρχαν θεσμοί κρατικοί που είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν μια κρατική υπόσταση. Ε, υπήρξε λοιπόν μια αισιοδοξία ότι αυτή η δουλειά τελείωσε και τώρα αυτό που χρειαζόταν να ολοκληρωθεί πλέον η πολιτική διαδικασία και όχι η διαδικασία γέννηση των θεσμών. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχει οδηγηθεί σε αποτελμάτωση εκ τότε η πολιτική αυτή ατραπός και είναι μικρή η εργασία ε, σε πολιτικό επίπεδο για τα μεγάλα θέματα. Ταυτόχρονα βλέπουμε και κάποιες εξελίξεις οι οποίες υπονόμευσαν τη ζωτικότητα και τη βιωσιμότητα της ε, διαδικασία του Παλαιστινιακού κράτου. Το ένα είναι μια αυξανόμενη κόποση των δωρητών όσο και αμφισβήτηση για το κατά πόσο έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία εφόσον δεν υπάρχει η πολιτική πρόοδος. Το δεύτερο ίσως είδος προβλημάτων είναι όλοι οι περιορισμοί που ε, συνεχίζει να επιβάλλει η ε, Ισραηλινή κατοχή σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στην ε, ε, περιοχή C, όπως είναι γνωστά στη Δυτική Όχθη τα κατεχόμενα, ε, η σύνδεση Δυτικής Όχθης με τη Γάζα, εξαγωγές Παλαιστινιακών προϊόντων ε, προς τον υπόλοιπο κόσμο και στην κανονική του συναλλαγή με το Ισραήλ και μια σειρά άλλων περιορισμών πολλών που υπονομεύουν αυτό που κανονικά θα ήταν η φυσιολογική ανάπτυξη της Παλαιστινιακής οικονομίας και μεγέθυνση. Πριν από λίγα χρόνια η Παλαιστινιακή οικονομία ε, αυξανόταν εντυπωσιακά. Αυτό τώρα έχει κάπως καθίσει Κάποια στιγμή φάνηκε ότι μπορεί να μην είχαν και ανάγκη από τους δωρητές οικονομικοί. Τώρα αυξάνεται η εξάρτησή τους. Ο, ο Πρωθυπουργός Φαγιάντ λέει ξεκάθαρα ότι εκείνος θέλει να φτιάξει κράτος, το οποίο να είναι όσο γίνεται ανεξάρτητο και από την ανεξάρτητη και τη διεθνή συγγνώμη, βοήθεια. Αλλά ακόμα αυτό δεν συμβαίνει. Είναι οξία λοιπόν η οικονομική κρίση ε, στα παλαισθηνιακά εδάφη. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη αυτή η ανάγκη. Τι σημαίνει αυτό. Ε, μετά την έραξη φέτος της σχολικής χρονιάς, έχουν χάσει τα παιδιά 36 ημέρες μαθήματος, γιατί δεν πληρώνονται οι δάσκαλοι και απεργούν, υπάρχουν προβλήματα οικονομικά στο εσωτερικό πλέον ε, της Παλαιστινιακής Αρχής. Εξαιτίας ε, της υπολοιπόμενης ε, οικονομικής βοήθειας. Και επίσης η Ισραηλινή κυβέρνηση ήταν πολύ ε, αργή και εμπόδισε την επιστροφή των εσόδων ε, ε, από δασμούς και φόρους από τα παλαιστινικά προϊόντα. Αυτά τα χρήματα ανήκουν στους Παλαιστινίους, δεν ανήκουν στους Ισραηλινούς. Θα πρέπει να τους επιστραφούν, πράγμα που δεν συμβαίνει. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση με την αίσθηση ότι υπάρχει μια οξία ε, χρηματοοικονομική κρίση. Βέβαια με τη στενή έννοια επέτυχε η συνεδρίαση, βρήκαμε και άλλα κονδύλια, ο προπολογισμό φαίνεται να είναι καλύτερο από ό,τι είχε υπολογιστεί πριν ε, τη συνεδρίαση και σε μεγάλο βαθμό θα είμαστε σε θέση μάλλον να καλύψουμε το έλλειμμα του Παλαιστινιακού προπολογισμού. Δηλαδή θα επιβιώσουν για μερικούς μήνε ακόμα. Αυτά είναι τα καλά νέα. Αλλά τα δυσάρεστα και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ποια είναι. Ταυτόχρονα υπάρχει πολύ μεγάλη αίσθηση ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση για πολλά χρόνια ακόμα, εάν δεν υπάρχει πολιτική διαδικασία που να επιστρέψει. Γιατί ε, ουσιαστικά ε, συνεχώς αναβάλουμε την πραγματική λύση του προβλήματος, αν εξακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Και ε, ο κίνδυνος ποιος είναι. Είτε κατάρρευση προς το εσωτερικό, είτε πολιτική αναταραχή στους Παλαιστινίου. Ε, και τελικά ε, μπορεί να εκδιώξουν ε, τον πρόεδρο Αμπάς, τον πρωθυπουργό Φαγιάτ και να αναλάβουν ακραίες ακραίε αυξηθεί και άλλο η κόπος των δωρητών, οπότε κάποια στιγμή θα κλείσουν τη στρόφιγγα. Λοιπόν, συμπέρασμα... Και χαίρομαι που συμφωνήσαμε σε αυτό. Στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη θα συγκαλέσουμε σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη συνεδρίαση και θα δούμε αν έχει νόημα αυτή η διαδικασία ολόκληρη ή μήπως χρειάζεται αναθεώρηση συλλήβδινή στρατηγική. Ο πρόεδρος Ομπάμα και ο υπουργό Εξωτερικών και Αεριομόλογος μου είναι τώρα στη Μέση Ανατολή. Ε, υπάρχει κάποια αμυδρή ελπίδα ότι κάτι μπορεί να ε, αναζωογονηθεί, αλλά δεν είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά ε, ε, και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ήθελετε να σας πω και για τα υπόλοιπα θέματα. Να αναφερθώ λίγο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα αυτή της κυβέρνησής μου και βεβαίως εδώ και χρόνια, αλλά τώρα ε, δίνουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό, διότι μας προβλημάτισε σοβαρά και εμάς, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα, αλλά και το Συμβούλιο, αυτή η σχέση. Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η παρούσα μορφή. Νομίζω θα ήταν σωστό να πούμε ότι εκατέρωθεν συμφωνούμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, ΕΟΧ, και η συμφωνία του υλοποιεί αυτά που υποτίθεται ότι θα υλοποιούσε Υπάρχουν βέβαια κάποιες προσαρμογές που γίνονται αυτόν τον καιρό. διαρκή. Ξέρετε αυτή η διαδικασία είναι δυναμική. Είναι πολύ ευρύτερη ε, από ό,τι στο παρελθόν, πάντως αποδίδει. Η Νορβηγία, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι το πιο συνδεδεμένο μη μέλος. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος που να είναι ε, τόσο πολύ κοντά στο να είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Νορβηγία, χωρίς να είναι μέλος. Συμμετέχουμε στην εσωτερική αγορά μέσω του ΕΟΧ παντού, εκτός από την Αλία και την ε, Γεωργία που έχουμε άλλες συμφωνίες. Είμαστε μέλη του Σέγγεν. Δηλαδή, αν έρχεστε από το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλετε διαβατήριο για να πάτε στην Νορβηγία, γιατί μπαίνετε στη ζώνη Σέγγεν, όχι γιατί έρχεστε στην Νορβηγία. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Και επίσης, συμμετέχουμε στην ε, ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και άμυνας στην ΕΠΑΑ και σε άλλες προσπάθειες. Η συμφωνία για το ΝΕΟΧ είναι ευρύτερη ε, μακράν όλων των υπολείπων που έχει συνάψει ποτέ η Νορβηγία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, είναι και η Ισλανδία και το Λίχτενστάιν σε αυτή ε, τη ζώνη. 30 χρόνια είναι στο ΝΕΟΧ, ε, προσεχώς 31 με την Κροατία και βεβαίως διαπραγματευόμαστε την ένταξή της στο ΝΕΟΧ. Και ε, βεβαίως που καλωσορίζουμε αυτή την εξέλιξη όπως και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να σας πω, μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά, διότι ε, θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολλά ωφέλη και ευεργετήματα να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Αλλά μάλιστα είναι διπλής κατεύθυνση αυτός ο δρόμος, είναι αμοιβαίο το όφελος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κάτω-κάτω η Νορβηγία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος ε, της Ένωσης και ε, επενδυτής το 2% στην Ευρώπη ε, κατέχεται ε, το μετοχών από τη το κράτος της Νορβηγίας. Έχουμε ένα μεγάλο επενδυτικό ταμείο, εξάγουμε ενέργεια, ιδιαίτερα φυσικό αέριο. Και είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο με τη Ρωσία και την Αλγερία, τους δύο άλλους μεγάλους εταίρους εξαγωγής ε, φυσικού αερίου και ευρέως συμμετέχουμε στη συζήτηση για την ενέργεια στην Ευρώπη και θέλουμε να διαδραματίσουμε ρόλο, να είμαστε φίλος, εταίρος και γενικότερα πρωταγωνιστής στις μελλοντικέ αγορές της ενεργειακές στην Ευρώπη. Και επίσης ε, προσπαθούμε να επιδείξουμε και αλληλεγγύη με την παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη. Ε, αυξάνουμε τις δωρεές ε, του ΕΟΧ, τι είναι αυτό, αυτό είναι χρήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως στα πιο νέα αλλά και σε παλαιότερα, ε, σαν να πληρώναμε, πούμε, μια κρατική συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος με ένα αρκετό ποσό και στη χώρα μας υπάρχει συνένεση γι' αυτό και υποστήριξη παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε μέλη. Είναι ευρεία η άποψη ότι οικονομικά θα πρέπει να συνεισφέρουμε στην Ευρώπη και μάλλον είναι αυξανόμενη η τάση υποστήριξης. Επίσης, ε, μέσω του Διεθνέους ε, Νομισματικού Ταμείου συμμετέχουμε με δάνεια της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, τι εννοώ εδώ λοιπόν λέγοντας όλα αυτά ότι ελπίζω να μας ε, βλέπετε ως ε, στενό και σημαντικό εταίρο σας στην ευρωπαϊκή υπόθεση. Εγώ το 1994 υπερψήφισα να, την ένταξη, έχασε τον ναι με μικρή διαφορά, εν πάση περιπτώσει το όχι πέρασε. Αλλά περισσότεροι θεωρούμε τώρα στην Ορβηγία ότι ε, το επόμενο βήμα, το αμέσως μετά την ιδιότητα μέλους, είναι ο ΕΟΧ. Και πολλοί που δεν ήθελαν να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρονται που είμαστε στον ΕΟΧ, γιατί αυτό μας αποτρέπει από το να γίνουμε μέλη. Ε, ένα είναι το πρόβλημα, το έλλειμμα, είναι το δημοκρατικό λεγόμενο έλλειμμα, διότι δεν συμμετέχουμε εδώ, στο παρόν κοινοβούλιο, δεν παίρνουμε αποφάσεις. Ούτε εκπροσωπούμαστε στο Συμβούλιο, ούτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ορισμένοι από εμά θεωρούμε ότι τόσο πολλοί που είμαστε σωματωμένοι και ενεχόμεθα, καλό θα ήταν να γίνουμε και με έλλη. Αλλά αυτό δεν συζητείται, γιατί είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει πολιτική συνένεση το επόμενο διάστημα για να ε, υποβληθεί και πάλι αίτηση, ξέρετε ότι δύο φορές έχουμε υποβάλει αίτηση. Ξέρετε ότι είμαστε και υποψήφια χώρα και έχουμε μακρά εμπειρία υποψήφιας χώρας γιατί δύο φορές ζητήσαμε να μπούμε και δεν μπήκαμε. Το 72 και το 94 και θα χρειαστεί και κάποιος χρόνος ακόμα. Αυτή είναι η πλατφόρμα και εκεί θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και με χαρά βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο στις εκθέσεις τους είναι ε, ευνοϊκές. Μας επικρίνουν για ένα πράγμα που νομίζω είναι δίκαιο σε επίκριση και θέλω να είμαι και ειλικρινής. Θα μπορούσαμε να είμαστε ταχύτεροι στην ενσωμάτωση ε, της κοινοτικής νομοθεσίας, στην υιοθέτηση ε, στον ΕΟΧ. Τι κάνουμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή το αποφασίσουμε, το μεταφέρουμε πολύ καλά στο νομικό μας σύστημα. Εκεί είμαστε άριστοι στην εφαρμογή. Αλλά για να ληφθεί η απόφαση χρειάζεται πολύ χρόνος. Και τι λέμε ως κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας εκεί. Να ξεκαθαρίζουμε πρώτα τα μη προβληματικά ζητήματα και μετά να κάνουμε σοβαρή συζήτηση για τα λίγα καθόδια, πούμε, που θέλουμε κάπου να επιμείνουμε. Ε, λοιπόν, ανασυνταχθούμε. Και έρχομαι στο τρίτο και τελευταίο τώρα, πριν ε, γίνει η συζήτηση. Είναι η Αρκτική. Γι' αυτό που καμιά φορά λέμε στα αγγλικά high north, το, το, το, το απότατο βορρά. Τώρα high north είναι από εδώ. Ε, άμα τα βλέπεις από εδώ, όλα στην Νορβηγία είναι high north, είναι μακριά και βορράς. Αλλά ας πούμε αρκτική για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και ποιο είναι εδώ το μήνυμα. Μία από τις μεγαλύτερες φυσικές αλλαγές που συμβαίνουν αυτό τον καιρό στον κόσμο, για καλό ή για κακό δεν ξέρω, είναι το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι προειδοποίηση του πλανήτη. Βεβαίως θα πρέπει παγκοσμίως να το αντιμετωπίσουμε με καταπολέμηση του της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δεν είναι κάτι που προκαλείται επιτόπου εκεί. Είναι λόγω της υπερθέρμανσης γενικώ. Λιώνουν οι πάγοι. Ε, ε, αλλά στους πόλους και στο βόρειο και στο νότιο πόλο ε, είναι διπλάσια η αύξηση της θερμοκρασίας. Αν παγκοσμίω, ας πούμε είναι 2 βαθμοί Κελσίου, στους πόλους είναι 4 βαθμοί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πόσο δραματικές είναι οι συνέπειες. Και μία από αυτές τις επιπτώσεις είναι ότι μειώνεται ο πάγος και ε, εν μέρη και εν μέρη μετατοπίζεται από Ανατολά προς Δυσμάς και προς την Ευρώπη δηλαδή ε, βόρειες περιοχές λιώνουν οι πάγοι, οι μόνιμοι, εκεί που υπήρχαν πάγοι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί κανείς να πλέει στις θάλασσες πιο βόρεια πλέον. Και αυτό το βλέπουμε και στις ε, διπυρωτικές μεταφορές προς Κίνα και Ιαπωνία, από τη Βόρεια Νορβηγία. Το καλοκαίρι μπορεί κανείς να πλέει ε, φορτηγά πλοία ή κρουαζιερόπλοια, ξέρω εγώ, από τη Βόρεια Ευρώπη μπορούν να διασχίσουν από εκεί και να πάνε στην Ασία και Τούμπαλιν. Και ο χρόνος που χρειάζεται, ας πούμε, η Ρότερνταμ Γιοκοχάμα μειώνεται κατά 40% από το αν πας γύρω-γύρω από τις νότιες θάλασσες κτλ. Δηλαδή έχει σημαντική αλλαγή αυτό ε, ε, και γεωπολιτική. Είναι μια αλλαγή πολύ αξιοσημείωτη. Βέβαια πολλά ε, χρόνια θα περάσουν πριν από κτίσει μεγάλες διαστάσεις αυτό το φαινόμενο. Η ναυσιπλοή είναι δυνατή εκεί μόνο το καλοκαίρι. αλλά τώρα το καλοκαίρι είναι σχετική έννοια. Το τελευταίο πλοίο που πήγε στην Ιαπωνία ήταν το Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έρχεται πιο κοντά η Ασία ε, σε εμά γεωγραφικά, ε, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε το γύρο του κόσμου για να φτάσουμε στην Ασία, μπορούμε να πάμε και από βορρά. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Φανταστείτε μια υδρόγειο σφαίρα και κοιτάξτε την Αρκτική. Δεν είναι τόσο μακριά. Δηλαδή η Κίνα και η Νορβηγία είναι γείτονε. Μια χώρα μα χωρίζει, η Ρωσία. Τώρα, α μην το κάνουμε και θέμα. Δεν είναι τόσο μακριά. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και για αυτούς τους λόγους πολλές ασιατικές χώρες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να γίνουν παρατηρητές στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Και εγώ υποστηρίζω η Νορβηγία να υποστηρίξει σαφέστατα ε, την αίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει όντως παρατηρητής στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Όταν ανέλαβε η δική μας κυβέρνηση το 2005 είπαμε ότι η Αρκτική και ο Πότατος Βορράς, όπως λέγαμε τότε, είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητα εξωτερικής πολιτικής για την Νορβηγία. Να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί, το κάναμε και καταφέραμε να φτιάξουμε και μια πλατφόρμα για πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών της Αρκτικής. Ότι ισχύει η UNCLOS ε, που είναι ε, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης. Αυτό διέπει ε, Έχουμε μια διένεξη με τη Ρωσική Ομοσπονδία για τις οικονομικές μας ζώνες, αλλά το 2010-2011 μετά διαπραγματευτήκαμε. Διαπραγματευόμαστε 40 χρόνια, 40 και συμφωνήσαμε και μετά και ο Καναδάς και η Δανία συμφώνησαν και εκείνες για τις ε, ε, διαφιλονικούμενες περιοχές ε, στην Ακτική και είναι όλο λιγότερες οι αφισβητούμενες περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό. Κάθε φορά που διαβάζετε ένα άρθρο για την, η κούρσα για την Ακτική δεν είναι κούρσα, είναι λάθος. Είναι σημαντικό βεβαίως, αλλά το διαχειριζόμαστε. Είναι λίγοι οι ωκεανοί ή τα μέρη του κόσμου, οι θάλασσες που συμφωνούν όλοι για τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένες και της Ρωσίας, για το τι ανήκει σε ποιον δεν είναι αμφισβητούμενες περιοχές, δηλαδή δεν θα ε, διαπληκτιστούν εκεί χώρες για περιοχές. Και αυτό είναι σημαντικό και για τη θάλασσα της Νότιας Κίνας και άλλες θάλασσες. Το θέμα Λοιπόν, δεν είναι μόνο αποφασίσει τι ανήκει σε ποιον, αλλά και τι κανόνες ισχύουν. Ενεργειακά, περιβαλλοντικά κτλ. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και τα ειδικά όργανα που υπάρχουν, όπως είναι το Συμβούλιο της Αρκτικής, ε, είναι σημαντικό αυτό το όργανο και θέλουμε να επεκταθεί, αλλά και άλλα όργανα που υπάρχουν, αλλά όχι μόνο αυτό, ε, είναι μεγάλες οι προκλήσεις. Ε, λοιπόν, οι φορείς είναι ο IMO, Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, ας πούμε που αφορά εκεί την αυσιπλοεία στην Αρκτική και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον αυτός ο τομέας και εσάς θα πρέπει να σας ενδιαφέρει, ακόμα και αν δεν είστε βόρειοι, διότι είναι μεγάλες αλλαγές αυτές και έχουν σημασία για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, όχι μόνο τα βόρεια. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με τους Ευρωπαίους γειτονές μας της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά και έχουμε κοινή οπτική σε μεγάλο βαθμό. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε κάποια ζητήματα που τέμνονται, που είναι η αλληλεία, η ενέργεια, το περιβάλλον, νέες διμεταφορών, ασφάλεια ενεργητική και παθητική. Αυτά προσπαθούμε να ρυθμίσουμε με εταιρικό τρόπο. Αυτά ήταν μια γενική επισκόπηση και τώρα να κάνουμε και συζήτηση. Ε, αλλά είστε ελεύθεροι να με ρωτήσετε ότι άλλο θέλετε, προφανώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να ακούσουμε τον κύριο Γκάλακερ ο οποίος είναι συμπρόεδρος της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εκ μέρους της ε, αντιπροσωπείας της Μεκτής Κοινοβουλευτικής ε, Επιτροπής για τις σχέσεις με την Οβηγία, ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι ήταν ε, πολύ επικοδομητικός ε, ο διάλογος με την νορβηγική πλευρά ανέκαθεν και είναι και πολύ συστηματικός. Η συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής της 26 Φεβρουαρίου επικεντρώθηκε κυρίως στην ενεξελίξη αναθεώρηση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συμφωνία αυτή ήταν μακρογωνιαίος λήθος των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας και είναι όντως από τις πιο σφαιρικές ε, διεθνείς συμφωνίες ε, στις οποίες έχει προσχωρήσει η Νορβηγία. Όντως, Πολλές φορές η Νορβηγία ε, έχει συμμετάσχει σε αυτού του είδους τις συναντήσεις και γνωρίζουμε τα νορβηγικά συμφέροντα πολύ καλά, διότι πολλές φορές συμπιέπτουν με τα δικά μας. Είναι αμφίδρομες λοιπόν αυτές οι σχέσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Καλωσορίζω το γεγονός ότι η συμφωνία του ΕΟΧ θα παραμείνει βάση για την ευρωπαϊκή πολιτική και την ευρωπαϊκή κατεύθυνση της Νορβηγίας, κάτι που το εξέφρασε και η νορβηγική κυβέρνηση με μια λευκή δίβλο πρόσφατα. Φαίνεται να υπάρχει πάντως κοινή κατανόηση για το πολύ καλό ιστορικό που έχουμε καταγράψει στο, στη συμφωνία αυτή. Κάτι που βεβαίως δεν πρέπει να μας κάνει να πάυσουμε, να επαγρυπνούμε και να είμαστε σε επιφυλακή. Θα πρέπει η συμφωνία αυτή να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και για τα μηδέα ωφέλη και στο μέλλον. Για τα μηδέα ωφέλη των δύο πλευρών. Βεβαίω συνεργαζόμαστε στενά, γιατί αυτό έχει νόημα. Και προ αυτό το σκοπό πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινό κάποιε προκλήσει. Να αναφέρω δύο ω παραδείγματα. Κάτι που συζητήσαμε και στι συναντήσει μα στι Βρυξέλλε. Πρώτον, θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να επιταχυνθεί η ενσωμάτωση της σχετικής ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συμφωνία ΕΟΧ. Η ομοιογενοποίηση της ε, νέας αγοράς είναι σημαντική και για την εύρυθμη λειτουργία της Συμφωνίας και για τις ε, διμερείς αυτές σχέσεις. Και ως προς τα εποπτικά ιδρύματα για τις συμφωνίες αυτές θα πρέπει να βρούμε μια κοινώς αποδεκτή λύση που να επιτρέπει να συμπεριληφθούν οι απαραίτητοι άξονες στη συμφωνία αυτή, γιατί υπάρχουν και συνταγματικές ε, προκλήσεις από την νορβηγική πλευρά. Εννοείται βεβαίω ότι οι συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση και Νορβηγία ξεπερνούν τα όρια των όσων ορίζει αυστηρό η συμφωνία Στην τελευταία συνάντησή μα, στην Μεκτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή, συζητήσαμε και για την Αλία, εξαιρετικά σημαντικό κλάδο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Νορβηγία, και για εμπορικά ζητήματα στον τομέα του εμπορίου και της Γεωργίας έχουμε διαφορετικές απόψεις λόγω της ε, απόφασης της νορβηγικής κυβέρνησης να αλλάξει το σύστημα ενίσχυσης κάποιων γεωργικών προϊόντων. Ακόμα και αν καταλήξουμε σε συνένεση για το πώς θα πρέπει να αποτιμηθεί αυτή η απόφαση, στην τελευταία μας συνάντηση με τους ε, νορβηγούς βουλευτές είχαμε επικοδομητικό διάλογο και αποσαφηνίσαμε την συλλογιστική των μεν και των δε και για το γιατί οι απόψεις μας είναι αποκλίνουσες. Τέλος, η συνεργασία με τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας είναι ένα από τα θέματα προτεραιότητας στις διακοινοβουλευτικής μας συναντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία είναι στενά συνεργαζόμενοι, στενά, στενοί συνεργάτες στην τομέα αυτό. Και η όλη συνεργασία εξυπηρετείται από τα κοινά μας συμφέροντα και τις κοινέ μας αξίες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε βεβαίως και στην Αρκτική και είναι πρόεδρος ε, της... Ε, μάλλον ο, πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής ε, επισκέφθηκε επανειλημμένος την περιοχή. Ο πρόεδρος της ΕΖΕΣ συζητώντας με συναδέλφους από την περιοχή της Αρκτικής συνεργασία αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ακτικής είναι ε, αρμονική. Δεν έχουν προκύψει συγκρούσεις. Και βάσει της σύμβασης UNCLOS η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει ε, την όλη αυτή προσπάθεια και θέλει να είναι και μόνιμος παρατηρητής στο Αρκτικό Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι με τη στήριξη και τη Νορβηγία θα μπορέσουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Ακτικής. Στη γεωγραφική αυτή περιοχή υπάρχουν σοβαροί σημαντικότατοι πόροι πετρελαίου και αερίου που κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τρόπο βιώσιμο. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας σε άλλες περιοχές της Ιδρογείου κατά την αξιοποίηση τέτοιων πόρων και εν είδη συμπεράσματος να ζητήσω σχόλια για την κοινή διπουργική συνάντηση τον Μάιο φέτος για τα θέματα της Αρκτικής. Εκεί θα εξεταστεί το καθεστώς παρατηρητή και εδώ αναγνωρίζουμε βέβαια τη στήριξη τη Νορβηγία, αλλά θα θέλαμε να εντείνετε λίγο την επιρροή σα στου υπόλοιπου συνομιλητέ και συμμετέχοντε εκεί, που μπορεί για άλλους λόγους να αντιτίθενται στην δική μας συμμετοχή ως παρατηρητών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό που μας παρουσίασε τις απόψεις του. Ευχαριστώ. Ο κύριος, επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ελεφράγκα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε Υπουργέ. Χαίρομαι ε, που βλέπω ότι καταλαβαίνετε ισπανικά. Ε, Ανήκεται στο εργατικό κόμμα ε, της Νορβηγίας, αλλά θέλω πάρα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι θετικός και ενεργός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Νορβηγία και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την εξαιρετική συμφωνία αλλά και για τη συνεργασία με τη χώρα σας σε πολλούς τομείς. Και ιδιαίτερα στην Ευρωπόλ που είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Επίση, έχουμε και κάποιες δυσκολίες πρέπει να πούμε, όπως η καταγγελία που καταθέσετε στον ΠΟΕ, αλλά ε, είναι λογικό ότι σε κάποιες φιλικές σχέσεις καμιά φορά υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε. Δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχουμε όν μας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς από την προνομιούχα θέση σας ε, του Υπουργού Εξωτερικών μιας τόσο κοντινής χώρας ε, προς την Ένωση. Πώς βλέπετε τις δύο διαστάσεις της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και την εσωτερική, ε, εσωτερική αγορά, οικονομική και νομισματική ένωση, την κρίση που ζούμε τώρα μετά τη χθεσινή απόφαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου και επίσης πώς βλέπετε αυτή την κρίση, όχι μόνο την οικονομική κρίση χρέους, αλλά και αυτή την κρίση εμπιστοσύνης ε, που βλέπουμε στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ερώτηση δεύτερη. Έχει να κάνει με την εξωτερική προβολή μας. Μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας, δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς αξιολογείτε εσείς τη λειτουργία αυτού του νέου ε, σχήματος του ε, Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, όπου προεδρεύει είπατε πρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ποιο βαθμό αυτό ε, βοηθάει τη συνεργασία, τη συνεννόηση και πώς το βλέπετε εσείς ε, ως υπουργό Εξωτερικών. Και ένα τελευταίο. Είδα στο βιογραφικό σας ότι έχετε περάσει από τα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρω ότι υποστηρίζετε και βοηθάτε και ανθρωπιστικά την Συριακή αντιπολίτευση, η αντίσταση. Πώς βλέπετε εκεί την έκβαση. Θεωρείται όπως και κάποια κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να αρθεί μερικό το εμπάργο για να μπορέσει να υποστηριχθεί πιο άμεσα η αντιπολίτευση. Ή θεωρείτε ότι η πολιτική λύση μετά από διαπραγμάτευση ε, που υποστηρίζει ο πρόσωπος ε, του Αραβικού Συνδέσμου και του ΟΗΕ είναι η σωστή λύση. Και πώς βλέπετε και την υπόθεση μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά το βέτο της ε, Κίνας και της Ρωσίας για να λαμβάνουμε αποφάσεις πιο πρακτικές και πιο κατηγορηματικές για την επίλυση συγκεκριμένα του Συριακού. Καλά, δεν θα σας βομβαρδίσω με άλλες ερωτήσεις. Τελευταία, πώς βλέπετε τις επικείμενες εκλογές που είναι περιφερειακές και τοπικές στη Ρωσία, της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Σεπτέμβριο. Αυτά, Πρόεδρε, τα ολίγα. Ευχαριστώ. Next speaker, Mr. Watson. Ο κύριος Βότσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Κύριε Υπουργέ, όταν πήγατε στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, την περασμένη εβδομάδα, είπατε ότι ο σημαντικότερος εταίρος τη Νορβηγία είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εμεί είμαστε ο δεύτερο σημαντικότερο εταίρος σα ή υπάρχει κάποιο άλλο ε, μεταξύ μα. Χαίρομαι πολύ που έχουμε πάντως την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα και θα ήθελα να καταγραφεί η στήριξη της δικής μας ομάδας, της πολιτικής μας ομάδας για το έργο της Νορβηγίας κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις συμφωνίες του Όσλο μια σημαντική διαδικασία που, βλέπουμε, όπου ελπίζουμε να έχετε κάθε επιτυχία. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα περισσότερα για το πώς πήγαν οι συζητήσεις με τον Τζον Κέρι όταν ήσασταν στη Washington κατά την προετοιμασία της δικής του επίσκεψης ε, στη Μέση Ανατολή και της τρέχουσας επίσκεψης του Πρόεδρου Ομπάμα. Είπατε, νομίζω σωστά, ότι η Παλαιστινιακή πλευρά πιστεύει στη λύση των δύο κρατών. Και δεν μπορεί να συνεχίσει για πάντα το να μην υπάρχει ένα τέτοιο κράτος. Οι Αμερικανοί βλέπετε να θέλουν οι Παλαιστίνοι να επιμείνουν σε αυτή την ε, λύση. Θα πιέσουν τον Νετανιάχου. Γιατί είχαμε στο Στρασβούργο τον κύριο Περέ την περασμένη εβδομάδα, ο οποίο και πάλι δεσμεύτηκε υπέρ τη λύση αυτή των δύο κρατών. Αλλά βλέπουμε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη λύση αυτή. Εσείς λάβατε κάποια διαβεβαίωση από τον Τζον Κέρι προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύετε ότι με την νέα Ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί να υπάρχει κάποια καινούργια ευκαιρία ώστε να επιτευχθεί πρόοδος και να πάυσει παράνομος ε, επικισμός για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας. Από πολλές απόψεις φαίνεται να είναι καλύτερος ε, ε, Ευρωπαίος στις επιδόσεις η χώρα σας από ότι πολλοί, πολλές ευρωπαϊκές χώρες που εγώ γνωρίζω παίζεται ενεργό ρόλο στο χώρο του Σέγγεν και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε υποσχεθεί να κάνει το ίδιο κάποτε. Θα μου άρεσε αυτό, αλλά... Γνωρίζετε όμως και τις δυσκολίες που προκύπτουν από την έλλειψη δημοκρατίας. Με απογοήτευσε λίγο αυτό που είπατε ότι η πλήρης προσχώρηση της Νορβηγίας δεν είναι θέμα υπό εξέταση. Κατά την δική σας άποψη τα ερχόμενα χρόνια δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα να υπάρξει μια μεγαλύτερη στήριξη από την χώρα σας προς την κατεύθυνση της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε τη συμβολή σας, όχι μόνο στην οικονομία μας, αλλά και στη δημοκρατία μας. Και πραγματικά και την πολιτιστική σας την ε, συνεισφορά τη χρειαζόμαστε, για να οικοδομηθεί μια Ευρώπη ε, πιο σφαιρική. Δεν είναι μόνο οικονομική ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και πολιτικού χαρακτήρα έχετε και πολιτικά, πολιτιστικά στοιχεία να συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια. Και η Νορβηγία και η Ισλανδία λοιπόν ελπίζω στο εγγύ μέλλον να στραφούν περισσότερο προς την ε, πλήρη προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα για τον απότατο βορρά όπως τον ονομάζεται. Πολλοί εδώ ανησυχούμε γιατί δεν καταφέραμε να επιτύχουμε ταχύτερη πρόοδο προς μια οικονομία που να, να κινείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρά από τις παραδοσιακές. Πιστεύουμε ότι εν μέρει είμαστε υπεύθυνοι για το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής. Και μας ενδιαφέρει το τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην όλη συλλογιστική και μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Οδικό Χάρτη για το 2050 και το πέρασμα, τη μετάβαση στην πράσινη, την οικολογική ενέργεια. Ευχαριστούμε κυρία Γιακονσάρη, Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω όλοι στο Ευρωκοινοβούλιο εκτιμούμε την ε, ενεργή διπλωματική δράση της χώρας σας σε πολλούς τομείς, αλλά ιδιαίτερος στην προσπάθεια να βρεθεί λύση στην, ε, στο θέμα της, στο στην Παλαιστίνη. Επίσης μας απασχολεί το καθεστώς μόνιμο παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο. Η συνάντηση αυτή προβλέπεται για το Μάιο. Ήδη έχουμε κινητοποιηθεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ρωσία και ο Καναδάς ακόμη αντιτίθενται στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μόνιμο παρατηρητή. Όμως ζητώ κι εγώ από σας να τους μιλήσετε. Μιλήστε σε αυτούς τους διπλωμάτες, γιατί είναι σημαντικό και για μα να μπορούμε να έχουμε μια άποψη για τον από το βορρά. Τώρα, ο ρόλος της Κίνας στην πολιτική για την Αρκτική. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει, διότι μόλις διάβασα ότι στην Ισλανδία η μεγαλύτερη πρεσβεία είναι της Κίνας. Η Κίνα έχει τη δική της στρατηγική για μια Αρκτική απαλλαγμένη από τους ε, πάγους. Εσείς τι ε, σχέσεις έχετε με την Κίνα. Μας ενδιαφέρει πολύ από την πλευρά αυτής της πολιτικής. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι θα είναι το Ελντοράντο του μέλλοντος η Αρκτική. Είναι μια περιοχή με φοβερές δυσκολίες. Μόλις ε, διάβασα, λόγω χάρη, ότι η ΣΕΛ σταμάτησε να κάνει γεωτρήσεις στην περιοχή της Αρκτικής. Είναι δύσκολο λοιπόν σε αυτή την ειρηνική περιοχή να αποφύγουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και να διασφαλίσουμε μια ειρηνική λύση. Πώς λοιπόν θα εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα και των ντόπιων εκεί, των ε, ηθαγενών και ποιος θα είναι ο δικός σας ρόλος στην όλη αυτή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Mr. Gallen. Sir, thank you very much and... Ευχαριστώ πολύ και καλωσορίσατε, Υπουργέ. Ε, ο ΕΟΧ ε, μαζί με το Σέγγεν σημαίνει σχεδόν είσαι μέλος χωρίς να συμμετέχει στα θεσμικά όργανα. Δηλαδή δέχεστε ε, να ε, εφαρμόζετε αυτά που εμείς αποφασίζουμε χωρίς να συμμετέχετε στις αποφάσεις. Πάντως οι θύρες μας παραμένουν ανοιχτές, όποτε θέλετε. Για την Αρκτική και το λεγόμενο όποτε το Βορρά, εγώ είμαι εισηγητής του Κοινοβουλίου και το είπαν και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι παρόντες συνάδελφοι παρακολουθούν πολύ αυτά τα θέματα. Και ε, εκτιμούμε τα μάλα την υποστήριξη της Νορβηγίας για να δοθεί μόνιμο καθεστώς παρατηρητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αρκτικό Συμβούλιο. Ε, στην Ολομέλεια του Απριλίου μάλιστα έχουμε προφορική ερώτηση με συζήτηση και έτσι και το Κοινοβούλιο αλλά και είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει την ευκαιρία να μας πει πώς βλέπει τη μελλοντική συνεργασία. Αυτό ε, μπορούμε να το προσφέρουμε και η οικονομική συνεργασία μαζί μας. Είναι κάτι το ενδιαφέρον για όλα τα ενεχόμενα μέρη εκεί στην περιοχή της Αρκτικής. Ερώτηση λοιπόν. Η Λίζα Γιακονσάρη αναφέρθηκε σε αυτό και σας ζήτησε να, να πιέσετε τον Καναδά και τη Ρωσία να άρουν τις επιφυλάξεις τους. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, τι μηχανισμός υπάρχει για να καμφθούν αυτές οι αντιστάσεις ή οι δισταγμοί και από πλευρά των Ρώσων και των Καναδών. Μπορούμε κάπου εμείς να σας βοηθήσουμε και σε ποιο βαθμό. Ερώτηση τώρα που αφορά τη Μέση Ανατολή. Το Σαββατοκύριακο ήμουν στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα. Συζήτησα με πολλούς οι Παλαιστίνοι ε, νιώθουν μια ματέωση, ε, μια αγανάκτηση και σκέφτονται να μεταναστεύσουν κιόλας. ο πρώην υπουργός, ή πρώην υπουργός Εξωτερικών Τσίπη Λίβνη στο Ισραήλ τώρα ανέβαλε, ανέλαβε υπουργό δικαιοσύνης και θα είναι αρμόδια ε, για αυτά τα θέματα τώρα. Αλλά από αυτή την κυβέρνηση τη νέα κυβέρνηση του Ισραήλ διαβλέπετε καμία πρόθεση να επανέλθουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Γιατί ο, ο κόσμος λέει ότι μάλλον θα στραφεί στο εσωτερικό του Ισραήλ, θα ε, ομφαλοσκοπεί κάπως αυτή η κυβέρνηση γιατί τους πιέζουν ζητήματα δικά τους. Σήμερα ο Μπαράκ Ομπάμα φτάνει στο Ισραήλ τι πιστεύετε ότι θα είναι το δικό του μήνυμα σε σχέση με την ενευτική διαδικασία. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εξηγήσουμε εμεί στην νέα Ισραηλινή κυβέρνηση ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε. Σταματήστε τους επικισμούς. Σταματήστε τις απαλωτριώσεις των περιουσιών των Παλαιστινίων και επανέλθετε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων των ενευτικών. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Ο κύριος Σας παρακαλώ να είστε σύντομος στην ερώτησή σας. Ναι. Για εσά το λέω, όχι για μένα. Είναι απαντήσει ο Υπουργό. Ε, ευχαριστώ. Καλωσορίσατε ε, ε, Υπουργέ ε, θα σας μιλήσω γερμανικά και γερμανικά καταλαβαίνετε. Ε, τότε δεν σας φαίνονται ισπανικά αυτά που θα σας λέω, δηλαδή αλαμπουρνέζικα, το λέμε έτσι στη Γερμανία. Θέλω να σας ρωτήσω για τις κυπριακές τράπεζες. Ε, ρώτησε ο κύριος Σαλαφράνκα αλλά και στην Ισπανία παίρνουν χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ε, γιατί υπήρχε μια τεράστια φούσκα ακινήτων. Ε, τώρα γίνεται μια συζήτηση για τις τράπεζες, για τα ακίνητα κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Ο κύριος Γκάλερ αναφέρθηκε σε αυτό για την Παλαιστίνη και τη λωρίδα της ε, Γάζας και τη νέα Ισραηλινή κυβέρνηση. Εσείς ε, περιγράψατε κάποια βήματα, τι θα κάνετε για να βοηθήσετε τη διαδικασία, γιατί όλο και περισσότερο έχουμε την εντύπωση ότι η Ισραηλή κυβέρνηση τώρα θα ασχοληθεί με τα δικά της θέματα, τα εσωτερικά, τα κοινωνικά στη χώρα. Και δεύτερον, εκατέρωθεν και από πλευράς Παλαιστινίων αλλά και από πλευράς Ισραηλινών, Υπάρχουν ομάδες που έχουν μεγάλο συμφέρον να διατηρηθεί το status quo, γιατί ζουν από αυτό και κερδίζουν και δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. για την ένταξή σας, το είπε και ο κύριος Γουότσον, θα ήταν πολύ πιο απλό να μπείτε στην Ένωση και από πολλές πλευρές θα ήταν εμπλουτιστικό. Λέτε ότι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία καλείστε να δεχτείτε χωρίς να έχετε συναποφασίσει. Δεν το ξαναβάζετε αυτό στην ημερήσια διάταξη. Παρόλο που φαίνονται σκοτεινά και δύσκολα τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς σας περιμένουμε με αυτές τις αγκάλες. Ευχαριστώ. Ήσασταν ταχύτατος, ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ. Είμαι εισηγητής για τις σχέσεις Κοινοβουλίου Ισλανδίας. Και έχω μια ερώτηση για την Ισλανδία. Πώς γνωρίζετε, είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται το ενδεχόμενο ένταξή τη. Είναι εξαιρετικό ε, υποψήφιο. Όχι μόνο από τη σκοπιά της ε, πολιτικής της ακτικής για μας, αλλά επειδή ήδη είναι μέλος του ΕΟΧ και του Σέγγεν και ούτω καθεξής. Η ερώτησή μου αφορά το πώς βλέπετε εσείς την υποψηφιότητα της Ισλανδίας οι διαπραγματεύσεις ως σήμερα πώς γίνονται αντιληπτές στη χώρα σας. Και το ρωτώ, γιατί όπως φαντάζεστε, η προοπτική της Ισλανδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως ε, προσκύπτει, έρχεται να με τον ε, σκόπλο της Νορβηγίας. Είναι το πρώτο που αναφέρουν ε, ως όνομα οι, αντίμα, οι αντίπαλοι της ε, προοπτικής ένταξης της Ισλανδίας. Πώς βλέπετε εσείς λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, μήπως είναι ένα σφάλμα, μήπως θα έπρεπε να συζητηθεί και πριν τι εκλογέ το τι μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην Ισλανδία. Δεν είναι άδικο να επικρατηθεί η διαδικασία πριν τοποθετηθεί ο ίδιο ο λαό τη Ισλανδία. Ευχαριστούμε ο κύριος Βένσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Έιντε, κύριε Υπουργέ, που είσαστε τόσο σαφείς στην σχέση σας. Νομίζω ότι όλοι οι Σκανδιναβοί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για όσα είπατε σήμερα. Μιλήσατε για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγία σε αυτό το πλαίσιο. Μας ενδιαφέρουν βεβαίως οι εξελίξεις ούτως ή άλλως σε όλο τον κόσμο, αλλά ξέρουμε ότι η Νορβηγία έχει αναλάβει ενεργό δράση και για άλλα θέματα, όπως για την ε, Γερμανία. Θα ήθελα λοιπόν, Υπουργέ, να μας σχολιάσετε τη δική σας ε, την άποψη για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Γερμανία και για το τι μπορούμε να κάνουμε, όχι ε, η Νορβηγία, εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι εξελίξεις στο μέλλον θα συνεχίσουν ε, με τρόπο ειρηνικό, ε, ίσως και περισσότερο από ό,τι σήμερα. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε 10 με 15 λεπτά για να απαντήσετε. Έχετε πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα καλά σας λόγια και τις καλές και σημαντικές σας ερωτήσεις. Στα Ισπανικά, κύριε Σαλαφράγκα, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Όπως γνωρίζετε, έχω εργαστεί πολλά χρόνια ε, στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ε, για μας που είμαστε κοντά στην Ευρώπη, αλλά εκτός αυτής είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ε, για τη συμμετοχή μας στην Ένωση, γιατί ε, η συζήτηση αλλάζει από χώρα σε χώρα ανάλογα και με τα πολιτικά κόμματα και είναι σημαντικό και ενδιαφέρον να συμμετέχουμε σε τέτοιους πολιτικούς σχηματισμούς ε, στην ευρύτερη ένταξη στην Ευρώπη. Θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί δεν καταλαβαίνετε όλοι ισπανικά. Ε, πολύ σημαντικό αυτό που με ρωτήσατε για ε, πώς βλέπουμε εμείς τις εσωτερικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η Νορβηγία έχει το όφελος λόγω των ε, συνθήκων αλλά και της χρηστής διακυβέρνησης θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει μας πλήττει λιγότερο σήμερα η οικονομική κρίση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη επίγνωση και ε, πάρα πολύ στενερά λέμε στους ε, Νορβηγούς πολίτες ότι αν συνεχιστεί η ευρωπαϊκή κρίση θα μας πλήξει και μας γιατί είναι τόσο μεγάλη η ε, ολοκλήρωσή μας και τόσο μεγάλη η σχέση μας με την ευρωπαϊκή οικονομία και ε, το ΑΕΠ μας ε, δημιουργείται σε μεγάλο βαθμό από εξαγωγές, εισαγωγέ και συμμετοχή στην οικονομία σας. Ε, είναι πολύ μεγάλο το μερίδιο με την Ευρώπη. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να δείξουμε αλληλεγγύη και πολύ σοβαρά να τα πάρουμε όλα αυτά υπόψη. Η δική μου αίσθηση ποια είναι, που το βλέπω από την εγγύης αλλοδαπή ας πούμε η αποδόμηση είναι λάθος. Αυτό θα πυροδοτήσει πολύ μεγάλη αρνητική κλιμάκωση και οικονομικά και πολιτικά θα είναι δραματικό κάτι τέτοιο. Και παρόλε τι προκλήσει, πρέπει να σα πω ότι εμένα με έχει εντυπωσιάσει η ικανότητα να επιμείνετε, να προσπαθείτε να λύσετε ε, από κοινού την κατάσταση. Είδαμε τη δεκαετία του 30 τι σήμαινε όταν κάθε χώρα προσπαθούσε να λύσει τα προβλήματά τη από μόνη τη. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό δίδαγμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για εμά, που είμαστε από του πιο στενού γείτονέ σα και τέρου. Και πραγματικά ελπίζουμε η Ευρώπη γρήγορα να βγει από την παρούσα κατάσταση για να μπορέσουμε από κοινού να πάρουμε ένα καλύτερο εγώ παραμένω μακροπρόθεσμα αισιόδοξο, αλλά κάποια σκληρά χρόνια θα χρειαστούν για να φτάσουμε εκεί. Αυτό συνδέεται τώρα με το θέμα της εξωτερικής ε, προβολής και προοπτικής. Κάθε φορά ε, που βλέπω την κοινή εξωτερική πολιτική της Ένωσης, χαίρομαι. Ε, συμφωνούμε και με τη Βαρόνια Άστο την είπατε εκπρόσωπο, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά. Η, επόμενη συνεδρίασή μου θα είναι στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, όχι συγγνώμη, στο πίεση, στο, στην Επιτροπή Ασφαλείας. Το τελευταίο θέμα που συζητήσαμε ήταν για τη Βερμανία, όπως με ρωτήσατε κιόλας. Είναι λογικό όταν έχεις την ανάγκη να ασχολείσαι με τα εσωτερικά σου, χαλαρώνει η προσοχή στα εξωτερικά. Ε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον τόσο ορατή εκτός αυτής. Αυτό δεν είναι κριτική, είναι κατανοητό. Αλλά ε, σήμερα μια σύνοδος κορυφής ας πούμε έχει τόσα πολλά να ασχοληθεί με το εσωτερικό της Ένωσης ώστε η εξωτερική παραγωγή ας πούμε δεν είναι τόσο αντιληπτή. Το λέω πραγματικά με κάθε φιλικότητα και καλοπροαίρετα ότι χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό, Μέση Ανατολή, Αρκτική, Βυρμανία, Σουδάν, Βόρειο, Νότιο, αλλά ε, ακόμα και η ιδέα της ολοκλήρωσης μπορεί να δουλέψει και να μεταφερθεί πώς συνεργαζόμαστε. Μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και για τους Αφρικανούς, τους Νότιο Ασιάτες, Ασίας, Αμερική κτλ. Ε, είναι έμπνευση αυτό για τις δημοκρατικές χώρες να συνενώνονται και να συνεργάζονται πιο στενά και αλλού στον κόσμο. Και το υποστηρίζουμε θερμότατα. Για την ερώτηση που μου κάνατε τώρα για τη Συρία. Είναι η μεγαλύτερη τραγωδία στο σημερινό παγκόσμιο σκηνικό. Ουδής και ε, ε, εγώ έχω απάντηση πώς μπορεί να λυθεί αυτό. αλλά ένα σημαντικό τμήμα της απάντησης είναι να συνεννοηθεί το Συμβούλιο ασφαλεία και να καταλήξει σε ένα κοινό σχέδιο. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιο σχέδιο θα είναι αυτό. Το πρόβλημα σήμερα είναι ο διχασμός ο ίδιο στο εσωτερικό του Συμβούλιο Ασφαλείας και αυτό στέλνει μηνύματα και προ το καθεστώ του Άσαντ. Ότι έχει φίλου, έτσι υψηλά ισταμένου. και επίσης ε, ε, και στην αντιπολίτευση στέλνει μηνύματα ότι έχει φίλου υψηλά ισταμένου και συνεχίζεται η σύγκρουση. Με έναν τρόπο που δεν θα σταματούσε μένα, αλλά θα μειωνόταν, εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε μία φωνή από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Χθε το βράδυ κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά. Εγώ δεν έχω επιβεβαίωση γι' αυτό, για τα χημικά όπλα, αλλά αν αρχίζουν να χρησιμοποιούν χημικά όπλα, αυτό αλλάζει η άρδιν την κατάσταση. Ε, στο μεταξύ, εμείς έχουμε επικεντρωθεί και συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανθρωπιστική βοήθεια για ανακούφιση στο εσωτερικό της Συρίας και στις γειτονικέ χώρες, ε, τους άμεσους γειτονές της. Και ε, με το Λίβανο έχω μεγάλη συνεργασία, αλλά και το Ιράκ και τη η αλλά ο Λίβανος με ενισχύει πολύ. Κάτι άλλο ρωτήσετε για τη Ρωσία που μπορούμε να το συνδέσουμε με την ευρύτερη ιστορία της Αρτικής. Όπως είπαμε για τη Ρωσία θα ήθελα να πω τα εξής δύο γρήγορα. Οι σχέσεις γειτονίας με τη Ρωσία είναι καλές. Έχουμε διευθετήσει διαφορές, δεν έχουμε ενέξεις ε, για τα σύνορα, τις οικονομικές ζώνες. Στην Αλία συνεργαζόμαστε, συζητήματα της Αρκτικής γενικότερα και Έχουμε γενικά συναντήληψη για αυτά τα θέματα. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε σαφή αρνητική τάση στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ε, βλέπουμε αντιδημοκρατικές τάσεις. Ε, ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών, τον ελεύθερο τύπο ε, και γενικότερα συστηματικά καταστέλλεται, μειώνεται. Και ως γείτονας της Ρωσίας ε, ανησυχούμε πολύ. Γιατί η διμερή συνεργασία δεν είναι μόνο Όσλο Μόσχα. Είναι τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, επιχειρήσεις που συναντώνται στο βορρά. Και αν ε, στενεύει όλο και περισσότερο αυτός ο χώρος είναι πρόβλημα για μας και έχουμε δικαίωμα να αντισταθούμε και να υψώσουμε τη φωνή μας σε αυτό. Θα πρέπει να την παρακολουθούμε τη Ρωσία και κυρίως οι γείτονές της να παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη πολύ στενά. Σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Βότσον, Πρώτον, είπα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι οι πιο στενοί μα σύμμαχοι. Σύμμαχοι με την έννοια τη στρατιωτική συμμαχία, αφού είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει ε, σημαντικότερο μέλος του ΝΑΤΟ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά ε, οικονομικά και πολιτικά συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι πολύ πιο ε, ευρεία η συνεργασία μας από ό,τι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είστε κι εσείς πολύ κοντά μας. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε, γιατί θα πρέπει να ενταχθούμε. Να σας καλέσουμε στην Νορβηγία να τα πείτε αυτά και στους ψηφοφόρους, γιατί δεν εξαρτάται από μένα. Και εγώ χρησιμοποιούσα αυτά τα επιχειρήματα, αλλά στο περασμένο δημοψήφισμα τι έλεγα. Ότι δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή καμιά πολιτική τάση που να λέγει ότι θα ήταν πάρα πολύ σόφρον να υποβάλουμε νέα ε, αίτηση ένταξης γιατί και δημοψήφισμα να γίνει θα χαθεί αυτό και μάλλον θα αναβληθεί και πάλι η πιθανή ένταξη. Δεν είναι επιτάπητος, δεν λέω ότι διαπαντός έχει ε, εκλείψει αυτή η πιθανότητα αυτό το ενδεχόμενο, αλλά προς το παρόν δεν τίθεται. Και βεβαίω. έχει δίκιο και ο κύριος Γκάλε. Προσαρμοζόμαστε Μάλλον όχι. Υιοθετούμε, λέτε, αυτά που αποφασίζονται χωρί να συναποφασίζουμε. Δεν έχουμε επιρροή εδώ ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στο Συμβούλιο. Ε, ε, θέτουμε κάποια ζητήματα και η καλύτερη επιρροή μας ποια είναι. Όταν εντοπίζουμε πολύ νωρίς ένα θέμα ότι θα ανακύψει, το συζητούμε πολύ φιλικά. Ε, άμα μας ενοχλεί κάτι με ε, τεκμηρίωση, με πραγματογνωμοσύνη και τα άλλα που υιοθετούμε, και εδώ να είμαστε, δεν θα άλλαζε τίποτα γιατί συμφωνούμε. Ο ΕΟΧ έχει εξυγχρονιστεί τώρα ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και ε, δεν είναι μόνο ε, η οικονομία ε, που μας απασχολεί, συγχρονιζόμαστε και εμείς. Αυτό που με ρώτησε επίσης ο κύριος Βότσον για τον Τζον Κέρι. Ναι, πιστεύω ότι οι Αμερικανοί κάπως θα πιέσουν το Ισραήλ ε, για τη λύση δύο κρατών για να επανέλθουν σε αυτή. Αλλά θα είναι αρκετή αυτή η πίεση. Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι συμφωνούμε εμείς απολύτως με τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ε, στην Νορβηγία για τη λύση δύο κρατών. Ναι, αλλά πόσο ισχυρή είναι αυτή η βούληση για να επιβληθεί. Εγώ τι λέγω στο Ισραήλ. Δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των Παλαιστινίων, αλλά και του Ισραήλ του ιδίου να υπάρχουν δύο κράτη. Διότι η εναλλακτική λύση ποια είναι. Λύση του ενός κράτους λογικά. Και αυτό το κράτος πολύ γρήγορα θα κυριαρχείται από Άραβες. Οπότε οι Ισραηλινοί ε, θα αναγκαστούν να δεχτούν ότι δεν είναι εβραϊκό κράτος το Ισραήλ, είτε ε, θα κάνουν τους Άραβες κάπως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ε, και οι δυτικές ε, δημοκρατικές χώρες θα αντιδράσουν. Δηλαδή, αν τους λες μακροχρόνια ποιο είναι το όραμά σας, οι Ισραηλοί πάντα σου λένε δύο κράτη. Βέβαια, οι σημερινές πολιτικές δεν το δικαιολογούν αυτό. Και αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς στη Γερμανία, στην Νορβηγία δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτοί έχουν πρόβλημα, οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλοί και πρέπει να το λύσουν. Εμείς το βοηθούμε ε, και δικό τους θέμα να λυθεί όμως. Έγιναν κάποιες ακόμα ερωτήσεις, ε, την κυρία Γιάκοσαρη και άλλους, για την ακτική, τον απότατο βορρά. Είμαστε προσιλωμένοι στην υποστήριξη τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αρκτικό Συμβούλιο. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά, ε, πολύ εντατικά στο εσωτερικό του Συμβουλίου για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Και το καλύτερο επιχείρημα που έχουμε και εμείς και εσείς πιστεύω είναι ότι μια χώρα όταν γίνεται παρατηρητής υπογράφει και ενστερνίζεται και τους κανόνες του οργανισμού στον οποίο προσχωρεί. Και εκεί εμείς έχουμε βασικούς κανόνες ε, και το να το δεχτούμε τούν αυτό και οι παρατηρητές είναι και προς το δικό μας όφελος των μονίμων μελών. Παράδειγμα, η σήμαση για το δίκαιο της θάλασσας. Είναι καλό όταν ο άλλος το δέχεται και το υπογράφει. Α, έγιναν και κάποιες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι τις έχω καλύψει σε μεγάλο βαθμό και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα με ρώτησε για την Ισλανδία. από την Ισλανδία εξαρτάται να αποφασίσει. Αν θέλουν να κάνουν συζήτηση στην προεκλογική εκστρατεία δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτό είναι των Ισλανδών. Τους εύχομαι καλή τύχη. Δηλαδή, αν θέλει να ενταχθεί η Ισλανδία, είναι καλό πιστεύω για την Ισλανδία και δεν είναι κακό για μας. Γιατί θα παραμείνουν στον ΕΟΧ. Ε, ΕΟΧ, ξέρετε, είναι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρε ΕΖΕΣ. Ε, θα είναι λιγότερο στην πλευρά ΕΖΕΣ, περισσότερο στην Ένωση, αλλά δεν θα είναι καμιά ριζική αλλαγή. Γιατί το κεκτημένο το έχει θετήσει και η Ισλανδία και εμείς. Και οι περισσότερες διεθνείς σχέσεις που έχουμε με την Ισλανδία είναι του ΕΟΧ. Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, αλλά τώρα εγώ τι να σας πω. Δεν θα αναμειχθώ στα θέματα που κυριαρχούν στη συζήτηση και μάλιστα την προεκλογική στην Ισλανδία. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε απαντώντας στον κύριο Σβένσον για τη Βερμανία. Μιανμάρ, τώρα πρώην Μπούρμα. Έχουμε μεταβεί εκεί τρεις φορές. Ε, συναντήθηκα με την ηγεσία τους και εκεί και αλλού και με την Aung San Και ο πρόεδρος ήρθε στην Νορβηγία πριν από λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε στενά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπα και την τελευταία φορά που σας είπα ότι είδα το Συμβούλιο το εσείς στην Ευρώπη. Ξέρετε, η ελίτ της χώρας έχει αποφασίσει να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να περάσει σε ένα δημοκρατικό κράτος. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βόλης στην κορυφή. Θα πρέπει τώρα οι υπόλοιποι και οι στρατιωτικοί να τα στερνιστούν αυτά. Αυτό που χρειάστηκε είναι να καταργήσουμε το παλιό καθεστώς κυρώσεων και να ανοίξουμε τις επαφές και τις επενδύσεις. Εμείς, και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν το είχαμε κάνει, μάλλον θα ήταν αυτή η απόπειρα πολύ βραχία. Ε, αγκαλιάσαμε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταργηθούν οι κυρώσεις, να γίνει αυτό το άνοιγμα, αλλά να μην σταματήσουμε εκεί. Έχουν περάσει μόνο δύο χρόνια. Είναι πολλές ακόμα οι προκλήσεις και εθνικές συγκρούσεις που πρέπει να λυθούν χρειάζονται δημοκρατικά θεμέλια και μια διοικητική μηχανή για να γίνουν σύγχρονη χώρα. Αλλά θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε ενεργά. Και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και νομίζω ότι κάλυψα. Δέκα λεπτά μου δώσατε, εντάξει είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και κάνατε αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το μεσημέρι θα έρθει ε, ο Επίτροπος κ. για να συζητήσει τρία θέματα. Τη Βοσνία, και έχουμε τρία θέματα. Τη, τη, τη Βοσνία, την Τουρκία και την αρχή της ευθύνης για προστασία. Λοιπόν, σας παρακαλώ να τηρούμε τους χρόνους. Η έκθεση προόδου για την Βοσνία Ερζεγοβίνη λοιπόν. Περνάμε στην δεύτερη εξέταση της πρότασης. Η συγγήτρια η κυρία Ντόρις Πακ. Η κυρία Ντόρις Πακ έχει μελετήσει προσεκτικά τις 101 τροπολογίες που υποβλήθηκαν στο σχέδιό της και έχει συμφωνήσει με το σχεδιό εισηγητή επί 8 συμβαστικών. Έχετε κατευθείαν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ. Είχαμε 100 και, και τροπολογίες. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να συγκλίνουμε με συμβιβαστικές προτάσεις και οι συνάδελφοι Σκιώδης ήταν πάρα πολύ ευγενείς και πάρα πολύ συνεργάσιμοι και καταλήξαμε σε ένα καλό έγγραφο, τους ευχαριστώ γι' αυτό. Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι συμβιβαστικές λύσεις ε, που συζητήσαμε. Να το γυρίσω όμως στα γερμανικά, γιατί μιλάω αγγλικά. Να πω μερικά θετικά, δυστυχώς τα υπόλοιπα είναι αρνητικά. Ε, χαίρομαι που οι τοπικές εκλογές και οι περιφερειακές ήταν ελεύθερες και απρόσκοπτες, αλλά παραμένουν τα προβλήματα στο Μόσταρ. Ε, δεν έγιναν εκλογές εκεί και στη Σρεμπρένιτσα. Ε, αυτά που είδαμε πρέπει στο μέλλον να αποφευθούν. Βεβαίως χαίρομαι ε, που τελείωσε η Διεθνής Παρατήρηση της περιοχής του Πρίτσκο. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Ας πούμε το 2012 ε, εγκρίθηκαν κάποιοι νόμοι για την απογραφή ας πούμε και τις κρατικές ενισχύσεις και κάτι τέτοια Ωραία, καλή η έγκριση της νομοθεσίας, αλλά και η εφαρμογή τη είναι άλλη ιστορία. Αυτό μα ενδιαφέρει. Τώρα, οι λιμένες αποφάσεις να υλοποιηθούν κιόλα. Τώρα, γενικά, αν θέλετε να κάνω κάποια εκτίμηση για τη χώρα, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση των πολιτικών να προχωρήσει η χώρα. Η συμφωνία σύνδεσης και σταθεροποίησης ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ, παραμένουν ακόμα εκκρεμότητες. Γι' αυτό δεν μπορούν να κάνουν και αίτηση προσχώρησης. Υπάρχει ένας ύπατος εκπρόσωπος εκεί, όχι η δική μας η ύπατος, ε, ένας διεθνής. Δεν είναι η κυρία Άστον. Ένας που πήγε εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 90 για να βοηθήσει μετά τη δύσκολη κατάσταση ε, με τη συμφωνία του Ντέιτον, θυμάστε, αυτό ήταν χρήσιμο. Αλλά το γεγονός ότι είναι αυτός ο κύριος εκεί επηρεάζει και τους ε, ντόπιου πολιτικούς οι οποίοι νύπτουν τα σχήρα τους, θεωρούν ότι δεν είναι υπεύθυνοι και αδρανούν. Διότι είπαν ότι αν δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε, θα αποφασίσει ο ύπατος εκπρόσωπος και τέλειωσε η υπόθεση. Μα δεν λειτουργεί έτσι μια δημοκρατία. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε ο ύπατος εκεί εκπρόσωπος το συντομότερο να αποχωρήσει από τη χώρα, να είναι σε θέση να αποχωρήσει. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Οι πολιτικοί της Βοσνίας θα πρέπει να το καταλάβουν και να το καταφέρουν μόνοι τους αυτό. Υπάρχει και ανασφάλεια, εμπλοκή από την κατάσταση στην Ομοσπονδία, στη μία οντότητα της χώρας ας πούμε, όπου υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία παρετείται, μετά δεν έχει αναλάβει ακόμα, είναι μπλοκή, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Και γι' αυτό και η χώρα δεν πλησιάζει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εμποδίζει αυτό. Στο Μόσταρ δεν έγιναν, είπαμε, εκλογές τοπικές Υπάρχει το καθεστώς της πόλης που μέχρι σήμερα δεν συνάδει με την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου και αν θυμάμαι την εποχή τότε που ο, ο κύριος Κόσνικ, πρώην δήμαρχος της Βρέμης, πήγε στο Μόσταρ και προσπάθησε να συνενώσει αυτή τη διχοτομημένη πόλη, σήμερα είναι πιο διχοτομημένη από ποτέ. Και ε, αυτό χάρη εντό εισαγωγικών των τόπιων πολιτικών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Τι του ενώνει. Επίσης, άλλο πριν από τέσσερα χρόνια το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο εκάλεσε τους πολιτικούς να ε, δουν τα ζητήματα των μειονοτήτων. Ήταν η υπόθεση Βίντσι. Γνωρίζετε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί τίποτα και είναι αδύνατο. Επαναλαμβάνω, οι ντόπιοι πολιτικοί δεν έκαναν το σύνταγμα που έλεγε τον Ντέιτον. Και γι' αυτό τώρα τους ενοχοποιούμε ή τους λέμε να τα αλλάξουν. Αυτό το σύνταγμα, τη συμφωνία στον Dayton δεν την έκαναν οι ντόπιοι, την έκαναν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή έχουμε κι εμείς κάποια ευθύνη και κάποια ενοχή. Αλλά πώς θα βγουν από αυτή την κατάσταση, μόνοι τους πρέπει να βγουν. Επίσης ζητούμε να γίνει απογραφή τον Οκτώβριο. Είναι απολύτως απαραίτητο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο είναι μεγάλη δυσκολία και για τις επόμενες εκλογές. Κάτι άλλο που ζήτησα και το υποστηρίζουν και οι συνάδελφοι, η δομή της Ομοσπονδίας, η οποία δεν είναι κάτι που αποφάσισαν αυτοί, το αποφάσισαν στην Ουάσιγκτον και στον Τέιτον. Αλλά να μπορέσει να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η Ομοσπονδία στις δομές της. Δεν επιτρέπεται να έχουμε 13 πρωθυπουργού, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσους υπουργού, καμιά καμία 150ρια την έχουν σε ένα τόσο μικρό τμήμα της χώρας. Ε, δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα ως δομές. Εμείς έξωθεν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είναι η δική τους δουλειά των ντόπιων εκεί πολιτικών. Εμείς να τους βοηθήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία διακυβέρνησης της χώρας. Έγινε μια απόπειρα πριν από δύο χρόνια. Είναι καταδικασμένο αυτό να αποτύχει. Έχω κάνει και δύο προφορικές τροπολογίες, πάρα πολύ σημαντικές. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να μειωθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση σε αριθμό, αλλά να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί η διοικητική μηχανή, να κάνει τα καθήκοντά της. Το πρόβλημα ποιο είναι. Τεράστια διαφθορά στη χώρα και εντός της πολιτικής ελίτ λεγόμενης. Δίνει και παίρνει, είναι τεράστιο θέμα η διαφθορά και εμποδίζει την πρόοδο παντού. Στην εγκατάσταση επιχειρήσεων, την ανάθεση των διορισμού, τα πάντα. Είναι αλληλένδετα. Όλα είναι πολιτικοποιημένα και όλα είναι σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένα και με διαπλοκή μεγάλη. Ένα άλλο θέμα μεγάλο είναι η μόρφωση και η παιδεία. Χαιρόμαστε τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δημιουργήσει μια task force, μια ομάδα κρούσης για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η επαγγελματική κατάρτιση να ε, προσαρμοστεί για να μπορούν οι επενδυτές να βρουν και εργαζομένους καταρτισμένους που να ξέρουν να πιάσουν δουλειά. Χαιρόμαστε που ε, τα πανεπιστήμια έχουν μπει στη διαδικασία Μπολόνια, αλλά πολλά πράγματα πηγαίνουν στραβά ακόμα. Κάτι που με ενοχλεί εμένα ε, ένα τμήμα της Ομοσπονδίας είναι ο διαχωρισμός στα σχολεία. Δηλαδή, στο ίδιο κτίριο ε, ε, είναι δύο σχολεία, αριστερά οι μουσουλμάνοι, δεξιά οι Κροάτες ή το αντίθετο. Μα επιτρέπονται τέτοια πράγματα να τα διαχωρίζουν την ώρα που μπαίνουν στο κτίριο το ένα σχολείο δεξιά, το άλλο αριστερά και μετά πώς θα έρθει η συμφιλίωση, πώς θα τα ξαναβρούν αυτά τα παιδιά. Αν τα ε, διχάζεις από μικρά και τους εμφυσείς αυτό το θέμα του διαχωρισμού. Και εκεί απέτυχε και ο ΑΣΕ, διότι συμφώνησε να γίνει αυτή ο διαχωρισμό στο σχολείο. Άλλο θέμα, οι πρόσφυγες. Πολλοί επέστρεψαν, είναι γεγονός αυτό, αλλά ε, δεν έχουν συμβεί ότι θα μπορούσε να συμβεί. Υπάρχουν και μεγάλες δωρεές τώρα σε ειδικού τομεί για την επιστροφή και τον επαναπατρισμό των προσφύγων και εγώ ίδια ε, το έχω αναφέρει και αναφέρω μία περιοχή και παρακαλώ το καταλάβουν πολλοί οι συνάδελφοι. Πρέπει να σας πω ότι 23 χρόνια ασχολούμαι με την περιοχή αυτή και ξέρω περί τίνος πρόκειται. Όταν λέω να βοηθήσουμε τον επαναπατρισμό των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης και της βίνα. Γιατί το λέω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν την ξέρετε την Ποσεβίνα. Είναι ένα κατεστραμμένο μέρος ε, στο βορρά της Ρεπούμπλικα Σέρψκα που παλιά μένανε μόνο Κροάτες. Ε, είναι μια πολύ έφορη περιοχή και τώρα ερημωμένη διότι οι Κροάτες έχουν φύγει, έχουν πάει στην Κροατία και δεν θέλει κανείς να επιστρέψει. Ε, μάλλον ακόμα και αν θέλει τους εμποδίζουν. Και για να χτίσουν σπίτι που έχουν μαζέψει λεφτά δεν έχουν φως, νερό, τηλέφωνο γιατί δεν τους βοηθάνε να ε, μπουν στις υποδομές. Οι Κροατές είναι στην Ερζεγοβίνη, ε, στη θάλασσα και δεν ενδιαφέρονται για αυτούς εκεί, ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους περιοχή. Εμείς θα πρέπει να ε, φροντίσουμε η να αναζωογονηθεί, να ξαναγυρίσει ο κόσμος και είναι και προσώφορο των ε, ε, Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Και αν ακούσετε τον κύριο Ντόντιτς, πρώην Πρωθυπουργό και τώρα Πρόεδρο, σε όλες τις συνεντεύξεις τύπου καλεί τους Κροάτες να επιστρέψουν. Αλλά δεν τους βοηθάει όμως και οι δήμαρχοί του, ας πούμε, τους μπλοκάρουν δεν δέχονται την εγκατάσταση, την ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κτλ. Λοιπόν, και εκεί υπάρχουν πράγματα που πάνε στραβά και θα πρέπει να βοηθήσουμε και τον κύριο Ντόντιτ και όλου όσοι είναι καλοπροαίρετοι να βοηθήσουν. Και είναι και προ το όφελο τη Κροατία να επιστρέψουν οι άνθρωποι στι ιστίε του. Ένα άλλο πρόβλημα που με απασχολεί πάρα πολύ και με στεναχωρεί είναι στο τέλος το θέμα ότι η Βοσνία ζεγοβινη είναι η μόνη χώρα που δεν αφήνει τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου ε, να μπουν με ταυτότητες ε, του Κωσόβου ε, στη Βοσνία. Ακόμα και οι Σέρβοι τους αφήνουν, οι Βόσνοι όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό και λυπηρό γιατί υπάρχουν πολλές βοσνιακές οικογένειες που ζουν στο Κόσοβο, που έχουν στενούς δεσμούς με τη Βοσνία, οικογένειες και δεν μπορούν να του δουν. Πρέπει να πάνε σε τρίτη χώρα να συνδάσουν του γενεί του. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει πραγματικά η Βοσνία τουλάχιστον να ακολουθήσει τη Σερβία σε αυτό. Να του αφήνουν να μπαίνουν με έγγραφα του Κωσόβου. Μέχρι και οι Σέρβοι είπαμε του δέχονται. Και ένα τελευταίο. Η Βοσνία, Ερζεγοβίνη, λόγω του γεγονότος ότι από την 1η Ιουλίου η Κροατία θα γίνει το 28ο μέλος της Ένωσης, πρέπει να αναλάβει μεγάλη προσπάθεια στα σύνορα για να είναι πιο απλή η διάβαση στους μεθοριακούς σταθμούς και τα εμπορεύματα που παράγονται στη Βοσνία πιο εύκολα να πηγαίνουν στις υπόλοιπες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειάζονται και δομές και υγειονομικές που προσπαθούν να τις φτιάξουν. Λοιπόν, συμπέρασμα. Απομένει τεράστια δουλειά, αλλά α μην αποθαρρυνθούμε. Μην αφήσουν να μας αποκαρδιώσουν και να μας απογοητεύσουν. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Η κυρία, Σα... Ε, η κυρία Μπάσκουρτ είναι ε, σκιώδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Πάρκ καταρχήν για τη συνεργασία για να εξευρεθούν συμβιβασμοί εκ, εκ μέρους ομάδας ε, σοσιαλιστών και δημοκρατών. Θέλω να πω ότι και εμείς λυπούμαστε για την έλλειψη πρόοδου στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τις αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να φτιάξουν αποτελεσματικούς ε, μηχανισμούς συντονισμού ώστε να μπορούν να μιλούν με μια φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας ποια είναι σημαντικά το θέμα της πρόσβασης της Κροατίας, της ένταξης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευπρόσδεκτες οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ε, αυτό βεβαίως αφορά έκθεση Βοσνία-Ερσεγοβίνης. Είναι σημαντικό όμως και οι δύο πλευρές ε, να προσεγγίσουν με οικοδομητικό τρόπο για τη βελτίωση, τη βελτίωση του μηχανισμού για να βελτιωθούν οι επαφές και να βρεθεί ένας τρόπος να, να βαθμίσει τις προσπάθειές της και η Βοσνία Ερζεγοβίνη και να επιληθούν οι, οι εναπομένουσες διαφομίες. Όσον αφορά το νόμο για, ε, για την απογραφή, θέλουμε να γίνει απογραφή και να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Εδώ πρέπει να υπάρχουν ε, αντικειμενικές καταγραφές του πληθυσμού, το οποίο προβλέπεται για τον Οκτώβριο. Η ανεργία των νέων ε, στη Βοσνία Αρζεγοβή είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Ζητήσαμε από τις αρχές να αναβαθμίσουν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, κυρίως με κατάρτιση, εκπαίδευση και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα εν γέννη. Τώρα, όσον αφορά το, την ύπατη ε, αρμοστία, θεωρούμε ότι όλα ε, τα, ε, όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να, να εκπληρωθούν μέχρι ότου μπορέσει να κλείσει το γραφείο. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σεβόμαστε τις αποφάσεις της Κεντρικής ε, Εκλογικής Επιτροπής για τη Σρεπρένιτσα, αυτό πρέπει να γίνει απολύτω σαφές, ότι οι αποφάσεις είναι σεβαστές. Δύο ερωτήσεις προς την κυρία Πακ. Είδαμε στον κατάλογο ψηφοφοριών ότι κάποιες ε, τροπολογίες δεν υποστηρίζονται από την εισηγήτρια. Αυτό είναι δικαίωμά τη. Όπως μία από αυτέ είναι η 71 που αναφέρει στατιστικά στοιχεία για τους πρόσφυγες στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά προέρχονται από, κατευθείαν από την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ρωτάμε λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα με την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει πρόβλημα με τις συγκεκριμένες στατιστικές κατά την άποψή μας ε, είναι, δεν είναι ξεκάθαρο γιατί δεν ε, τις υποστηρίζετε αυτές, γιατί αποτελούν απλώς πληροφορίες εξ όσων γνωρίζουμε. Και η άλλη ερώτηση αφορά την τροπολογία παριθμών 25. Υπάρχει ξεκάθαρη έκκληση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από πολλές ομάδες. Θέλαμε η Βοσνία Τζεγοβίνη να επισπεύσει την ε, διαδικασία ένταξης. Στην τροπολογία αυτή ζητάμε έναν ε, μηχανισμό fast track για την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν καλό για την, να επισπευστεί όλη η διαδικασία ένταξης. Άρα είναι μια αντίφαση εδώ ανάμεσα σε αυτό το οποίο ζητάμε και αυτό το οποίο υποστηρίζουμε ή δεν υποστηρίζουμε υποστηρίζει ή δεν υποστηρίζει η εισηγήτρια. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την εισηγήτρια να υποστηρίξει, να βάλει συν σε αυτές τις τροπολογίες. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριος Κάτσιν, λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η Σάρα Λάτφορτ δεν είναι εδώ δυστυχώς και έτσι θα, πω, θα μιλήσω εκ μέρους της ομάδας μου και θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ντόρις Πακ, για τα χρόνια με τα οποία έχει ασχοληθεί με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Βοσνία Ερζεγοβίνη επί, επί έναν αριθμό θητιών έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πολύ δύσκολα θα βρούμε κάποιον άλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να έχει καταβάλει τέτοια προσπάθεια και μάλιστα να έχει θετικά επιδιώξει να, να βοηθήσει τη Βοσνία να κάνει βήματα πρόοδου. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει επαρκής ανταπόκριση. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια γενικά είναι διαφορετική. Υπάρχει η Τρόικα, Κωσυφοπεδίου, Σερβίας και Μαυροβουνίου που πάει καλά και αν το Κωσυφοπέδιο ξεπερνάει τη Βοσνία Ζεγοβίνη, αυτό λέει πολλά. Πραγματι ο έβδομος κύκλος του διαλόγου μεταξύ των πρωθυπουργών, τον κύριο Ντάτσιτς και τον κύριο Τάτσιν, ε, πράγματι γίνεται. Και σήμερα Μπορεί, να επισυμβεί μια ιστορική πρόοδος. Όμως στα μέσα ενημέρωση της Βοσνίας διαβάζουμε ότι στις 23 του μήνα οι εκπρόσωποι των έξι ε, ισχυρότερων πολιτικών κομμάτων της Βοσνίας θα πάνε στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για το ελάχιστο των ελαχίστων που είναι η εφαρμογή της απόφασης της υπόθεσης Σέντιτς Βίντσι που αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του ε, δικαιώματος να είναι κανείς υποψήφιος στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έτσι λοιπόν η πολιτική μου ομάδα θέλει να επαναλάβει ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη πρέπει από μόνη της να βρει μια λύση. Αλλά τέτοια λύση δεν θα βρεθεί για πολύ καιρό ακόμα χωρίς τη βοήθειά μας. Η διοργάνωση μιας ειδική διάσκεψης για τη Βοσνία ριζεγοβινη θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι θετικό. Αν δεν τροποποιηθεί όμως το σύνταγμά της, η Βοσνία ριζεγοβινη δεν θα γίνει πλήρες κράτος. Βεβαίως, φτάσαμε στο σημείο που θα πω κάτι που θα σα ανησυχήσει, πολλού από εσά θα σα ανησυχήσει. όμω την Κυριακή επέστρεψα από τη Λιβύη. Εκεί εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το Σύνταγμα, το οποίο ανεστάλλει το 69 από τον Κατάφη, έτσι ώστε να γίνει λειτουργικό το κράτος τους. Ενδεχομένως λοιπόν η Βοσνία Ζεγοβίνη θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης της εποχής που ήταν κομμάτι της Ιουγκοσλαβίας και ενδεχομένως ε, μέρη αυτού του συντάγματος να μπορέσουν να επιτρέψουν στη Βοσνία Ζεγοβίνη να γίνει και πάλι λειτουργικό κράτος. Φυσικά τα πράγματα και στις δύο οντότητε είναι πολύ ε, περίπλοκα, ιδίως ως Ομοσπονδία, αλλά το γεγονός παραμένει ότι το κόστος ε, Μια τόσο σύνθετης και μη λειτουργική διοίκηση στραγγαλίζει την οικονομία της χώρας. Η οικονομία της χώρας δεν θα μπορέσει να επιζήσει. Φυσικά το θέμα της οικονομικής επιβίωσης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απαντηθεί γιατί οι νέοι θα αρχίσουν να διαρωτώνται αν αξίζει τον κόπο να παραμείνουν στη χώρα ή όχι. Το 90% του, πληθυσμού, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, πιστεύει ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη δεν προχωρεί προς την ε, σωστή κατεύθυνση με το σημερινό πολιτικό προσωπικό της. κυρία Κοπά για δύο λεπτά παρακαλώ είστε πολύ ικανοί στο να τηρείτε το χρόνο σας. Ε, Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Πακ για το σχέδιο έκθεσής της και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για κάποιες επικοδομητικές ε, τροπολογίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη αποτελεί το μεγαλύτερο ε, κριτήριο αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ε, πράγματι γεγονός ότι έχει καθυστερήσει στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κατόπιν αυτού η κριτική στάση της έκθεσης είναι απολύτως κατανοητή. Θεωρώ όμως εξαιρετικά σημαντικό να επαναλάβουμε ξεκάθαρα την αφοσίωσή μας στην ε, ολοκλήρωση της Βοσνίας Εζεγοβίνης πράγμα που, την ένταξή της, πράγμα που θα ωφελήσει όλους. Έχω ζητήσει να, ενταχθούν, να ενταχθεί μια ξεκάθαρη δήλωση στην αρχή της έκθεσης και ελπίζω ότι αυτό θα το υποστηρίξετε. Η υποστήριξή μας προς τη χώρα είναι σημαντική, ιδίω για αυτούς οι οποίοι βλέπουν το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας ως μία ή και τη μοναδική λύση για πολλά από τα εσωτερικά της προβλήματα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα προβλήματα αυτά ε, επιδεινώνονται από την οικονομική κρίση και σχετικά με αυτό θέλω να καλωσορίσω την πρόσφατη απόφαση της ε, παροχής βοήθειας 100 εκατομμυρίων ε, ε, ευρώ στην Ευρωπαϊκή, στην Βοσνία Ερτζεγοβίνη τη στιγμή που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με ανεργία. Πρέπει να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια για να μπορέσει η χώρα να μιλάει με μια φωνή απέναντι στο, στην Ευρώπη για το ευρωπαϊκό της μέλλον, να φτιάξει ένα λειτουργικό κράτος και να μπορέσει να διαπραγματευτεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ένταξης. Αυτή ήταν η λογική πριν, πίσω από την τροπολογία υπαριθμών που υπέβαλα. Θέλω να δείξω ότι χρειάζονται οι συνταγματικές αλλαγές και προσαρμογές, όχι μόνο συνολικά, αλλά σε τοπικό επίπεδο και επίπεδο οντοτήτων. Αυτό δεν φάνηκε στο αρχικό κείμενο. Τώρα έχει ξεκαθαριστεί με το συμβιβασμό και τον υποστηρίζω πλήρως. Η, μια συμφωνία για τη δημιουργία ενός συντονιστικού μηχανισμού είναι επίσης απαραίτητος. Θέλουμε να έχουμε ένα συνομιλητή που να μιλά εκ μέρους του ενιαίου κράτους της Βοσνίας Ερσεγοβίνης και δεν μπορούμε πλέον να επιτρέπουμε να γινόμαστε μέρος της εσωτερικής διαμάχης. Τέλος, επειδή έχουμε μια, να αντιμετωπίσουμε μια κοινωνία που έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην συμφιλίωση και στα εγκλήματα ε, ε, μίσους. Θα πρέπει να καταδικαστούν τέτοιου είδους εγκλήματα και να γίνει έρευνα και να τιμωρηθούν οι δράστες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. With your permission I will speak in Greek. Ε, θα μιλήσω ελληνικά. Εγώ την κυρία Πακ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, να τη συγχαρώ για την πολύ καλή γνώση, την εξαιρετική γνώση που έχει όσον αφορά την Βοσνία ζεγοβινη Να σας πω ότι έχω και εγώ μια σημαντική εμπειρία, γιατί πέρασα αρκετό καιρό σε θελοντής γιατρός κατά τη διάρκεια του πολέμου και ξέρω πάρα πολύ καλά την τραγωδία σε όλη τη την διάσταση. Επισημένω από αυτά που είπε η κυρία Πακ όχι μόνο μια φορά, ότι αυτό το σύνταγμα της τριζωνικής περίπου ομοσπονδίας που έχει σήμερα η ε, Βοσνία και που βασίζεται σε εθνοτικό, θρησκευτικό και γλωσσικό διαχωρισμό έχει επιβληθεί στη χώρα από κάποιους άλλους που αποφάσισαν αλλού στις ΗΠΑ, εμάς, δεν ξέρω από ποιους. Έχει επιβληθεί το Σύνταγμα αυτό και φαίνεται πόσο μη λειτουργικό είναι, πόσο αντιπαραγωγικό, πόσο αδύνατο ε, να βοηθήσει τον λαό να προκόψει. Και από την άλλη η κυρία Πακ μας είπε ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην ε, διόρθωση αυτού του κακού. Αυτό το επισημαίνω γιατί είμαστε επιρρεπείς να κάνουμε τα ίδια λάθη συνέχεια. Ευχαριστώ. Mr. Ε, ο κύριος Βεβαίως, θέλω και εγώ, καταρχήν, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και θέλω να ευχαριστήσω ότι πραγματικά έχει εκτεταμένη γνώση. Όπως επίσης ότι γνωρίζει συναισθηματικά να εμπλέκεται με την υπόθεση. Η, διαχείριση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης σε μια τέτοια στιγμή συνεπάγεται το βάρος των μη πολύ επιτυχημένων παρεμβάσεων της διεθνούς κοινότητας στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτό αποτελεί συνέπεια του ότι χρησιμοποιήθηκαν προαποφασισμένες λύσεις για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Οι βοσνιακές αρχές πρέπει τώρα να καταλήξουν σε νέο σύνταγμα. Παλιά χρειαζόταν, τώρα δεν είναι λύση πλέον αυτό το θέμα για τη βοσνια Ζεγοβίνη είναι ότι πρέπει να οικοδομηθεί ένα κράτος της βοσνιας Ζεγοβίνης. Όμως το κράτος δεν μπορεί να οικοδομηθεί με βάση ένα μη λειτουργικό σύστημα διοίκησης. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το πρόβλημα του αυξανόμενου εθνικισμού και σε κάποια από τα γειτονικά κράτη της Βοσνίας Ερσεγοβίνης. Θέλω να αναφέρω τους γείτονες που έχουν κάποιους, κάποια μέρη του πληθυσμού στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Ο εθνικισμός επιστρέφει στη Βοσνία Ερσεγοβίνη και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Πρέπει η ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση να παραμείνει ανοιχτή για τη χώρα αυτή. Αλλά βεβαίως πρέπει να πούμε και το εξής θα πρέπει να είμαστε πιο γενναιόδοροι απέναντι σε, όλους, σε όλα τα πρώην κράτη της Ιουγκοσλαβίας. Δεν θα πρέπει να ακολουθούμε κάποια τακτική. Θα πρέπει να αποδεχτούμε χώρες με σοβαρά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας έχουν και αυτές προβλήματα. Αν τις αποδεχτούμε αύριο θα λυθούν πολλά από αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κυρία Πακ. Και όντως η έκθεση αυτή είναι κάτι, και το γνωρίζει και η ίδια, που λέγει ότι η λύση για τη Βοσνία Ζεγοβίνη περνά από την ανάκτηση της κυριαρχίας της και η ομάδα μου αυτό τονίζει. Έχει φτάσει η ώρα η κυριαρχία του βοσνιακού λαού να επικρατήσει και ελεύθερα ο λαός της Βοσνίας να ορίζει το μέλλον του. Η ομάδα μου λοιπόν κατέληξε στο συμπέρασμα και επιμένουμε ότι θα πρέπει να σταματήσει να τερματιστεί το Διεθνές Προτεκτοράτο, να κλείσει το γραφείο του ΙΠΑ του εκπροσώπου της, ε, του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις του συντάγματος για να μπορέσει ο λαός της Βοσνίας να αποφασίσει για το μέλλον του χωρίς καμία εξωτερική ανάμειξη, κανενός είδους και να γίνουν και όλες οι μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία των μειονοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανηλίκων. Και στις τροπολογίες μας η ομάδα μας θα τα υπογραμμίσει αυτά ε, τα τελικά θα ψηφίσουμε αποχή στην έκθεση γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχει εξεταστεί αυτή η ανάγκη να εγκαταλειφθεί, να τερματιστεί το προτεκτοράτο και να αποφασίσει ο λαός της Βοσνίας για την αυτοδιάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γέρκοβιτς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ως παρατηρητής από την Κροατία, θα ήθελα εν συντομία να προσθέσω κάποια σχόλια. Καταρχήν, κυρία εισηγήτρια, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά σας. Είναι απολύτως σαφές ότι γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σύνθετο είναι το θέμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση της Κροατίας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ε, για την περιφερειακή συνεργασία και στηρίζει πλήρως την πρόοδο και τις μεταρρυθμίσεις των χωρών της περιοχής εν ώψη της ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη Βοσνία-Ερσεγοβίνη, η Κροατία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα όχι μόνο υπό την έννοια του καλού γείτονα, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι Κροάτες είναι ένας από τους τρεις λαούς που αποτελούν τη Βοσνία σεγοβινη Θα ήθελα να κάνω λίγα σχόλια για την, επί της παραγράφου 17. Το περιεχόμενο της παραγράφου αυτής αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση της ε, περιοχής της Ποσαβίνα. Και όπως επεσήμανε και η κυρία Πακ, η επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισμένων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι οι βραδύτερη στην περιοχή και κυρίως αυτό αφορά τα μέλη της κροατικής κοινότητας. Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού του 1991, η κοινότητα των Κροατών ήταν η πιο πολυάριθμη της περιοχής και είχε πάνω από 130.000 μέλη. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία, το λιγότερο από 5% των Κροατών προσφύγων έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Υπό την έννοια αυτή, για το θέμα αυτό μάλλον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυβέρνηση της Κροατίας συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση της Βοσνίας και η Κροατία είναι ο μεγαλύτερος δωρητής της ανοικοδόμησης σπιτιών στην περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί, θα έλεγα, η επιστροφή, δεδομένου ότι το 70% των ε, προσφύγων από την Ποσαβίνα της Βοσνίας εξακολουθούν να ζουν στην Κροατία. Ελπίζω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα υποστηρίξετε την αρχική παράγραφο 17 της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία εισηγήτρια. Θα είμαι πολύ σύντομη, μην ανησυχείτε. Ήθελα να καθησυχάσω την κυρία Μπάσκοφ ότι είμαι υπέρ της 25 και της 72 όπως είπατε. Τις πάντων δύο αυτές που είπατε κυρία Μπόσκουρτ. Έκανα λάθος εγώ. Επίσης θέλω να σας πω, να πω στους πρασίνους, νομίζω τους, στους πρασίνους, δεν ξέρω, που είπαν ότι δεν θέλουν να το ψηφίσουν θέλουν να, να βγουν οι δύο εκπρόσωποι. Ακούστε, ο Ευρωπαίος είναι ο πρέσβης μας ε, και δεν έχει εξουσία ως ε, υπατος εκπρόσωπος σας παρακαλώ να κάνετε διάκριση ανάμεσα στους δύο. Θα χαρώ πολύ να φύγει ο διεθνής, αλλά ο άλλος πρέπει να μείνει γιατί εμάς μας ενδιαφέρει αυτή η χώρα και πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, έστω στέλνοντας έναν βαθμό πρέσβη. Και επίσης θέλω να ζητήσω από τους συναδέρφους να καταλάβουν ότι η ψηφοφορία θα γίνει μόνο το Μάιο. Δεν είναι κατεπήγον, δεν μπόρεσα να ενημερώσω νωρίτερα του Σκιώδης. Όχι τον Απρίλιο, το Μάιο θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, στην Ολομέλεια του Μαΐου. Ζητώ συγγνώμη, το καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Όλοι νομίζω είμαστε υπέρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο σύνολό της. Thank you. I would remind you that the vote will be tomorrow. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε αύριο στις 9 ακριβώς όμως αυστηρά. So, the second... Λοιπόν, έκθεση προόδου για την Τουρκία. δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης για το 2012 για την Τουρκία. Εξέταση των σοβιβαστικών τροπολογιών. 415 τροπολογίες κατατέθησαν. Δίνω ευθύ αμέσως το λόγο την κυρία Ρία Όμεν Ρούιτεν λεπτά. Ε, ε, και Στα αγγλικά. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους κοιόδης συγητές μου για τις ώρες ολόκληρες που συνεργαστήκαμε για τη δέσμευσή του και την πολύ επικοδομητική τους στάση και συνεισφορά. Είχαμε όντως πολύ εντατικές συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να πω ότι είναι ευρεία η συναντήληψη για το περιεχόμενο του ψηφίσματος αυτού. Έχω πει και στο παρελθόν ότι το 2013... Κύριε Πρέντα, Λοιπόν, έλεγα, έχω ξαναπεί ότι το 2013 θα αποδειχθεί σημαντική χρονιά στη σχεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα διατηρήσουμε και θα μετεξελίξουμε την περαιτέρω της επικοδομητικής μας ε, σχέσης σε αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. Και πιστεύω ότι η εκ νέου δέσμευση στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγματεύσεων είναι κάτι που χρειάζεται για να φτάσουμε σε μια νέα αμοιβαία ε, δέσμευση ε, χρειάζονται προσπάθειες εκατέρωθεν. Πραγματικά το λέω αυτό και το τονίζω. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, τονίζουμε τη σημασία ε, μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύγχρονο δικαστικό σύστημα τελείως αμερόληπτο και απολύτως ανεξάρτητο. Το τρίτο ε, πακέτο για τη δικαιοσύνη ήταν ένα σημαντικό βήμα, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο να συνεχιστεί. Υπάρχει ένα τέταρτο πακέτο που πάει τώρα στη Βουλή, στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και προσβλέπω στην τελική έκφαση της τέταρτης δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Τι λέει λοιπόν αυτή η δέσμη. Είναι βασική προτεραιότητα Ε, υπάρχει ένας ευρύτατος ορισμός για τις αξιόπινες πράξεις, για την τρομοκρατία στον αντιτρομοκρατικό νόμο και στον ποινικό κώδικα. Το ψήφισμα λοιπόν, αλλά και οι συμβιβασμοί τονίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης των περιορισμών ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ευρύτερη έννοια του κράτους δικαίου δεν είναι μόνο η νομοθεσία, η έγκρισή της, αλλά και η εφαρμογή της. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειες που καταβάλει. Αλλά και η δική μας πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Τουρκία στην προσπάθεια αυτή. Επίσης πιστεύω ότι αν μιλούμε για τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρειάζονται επίσημη ε, γνώμονες, ε, benchmark, ε, δείκτε συγκριτικοί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Αυτό είναι σημαντικό για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ας πούμε, Επίσης υπάρχουν και προθέσεις αλλά και διαβουλεύσεις, για, διαπραγματεύσεις για να λυθεί το κουρδικό αλλά και κάτι άλλο πάρα σημαντικό πάρα πολύ σημαντικό, συγγνώμη, που είναι το νέο σύνταγμα. Συνδέονται αυτά τα θέματα και στο ψήφισμα. Για το κουρδικό. Γίνονται κάποιες συνομιλίες που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ιστορική συμφωνία για να λυθεί το κουρδικό ζήτημα με τρόπο ειρηνικό και δημοκρατικό. Τι γίνεται με τη συντακτική διαδικασία επενούμε ε, τη διακομματική συμφωνία για την αναθεώρηση του συντάγματος και επίσης επενούμε το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια και την πρωτοβουλία. Αλλά όλα αυτά δεν αρκούν. Δεν προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Έχουν κάνει τροπολογίες και οι φιλελεύθεροι συνάδελφοι που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να υποστηριχθεί η συντακτική ε, διαδικασία. Ποιος είναι ο ρόλος τώρα της Τουρκίας στην περιοχή είναι σημαντικός ε, πρωταγωνιστής στην περιοχή και έχει και στρατηγικό ρόλο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ο υφιστάμενος πολιτικός διάλογος θα πρέπει να ενισχυθεί και εγώ ενθαρρύνω, ενθαρρύνουμε την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στα πλαίσια του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του συντονισμού. Ταυτόχρονα όμως το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την υποστήριξη ε, στη δέσμευση της Τουρκίας για την υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων στη Συρία. Λυπούμε βαθύτατα, και το λέω εδώ ξανά, για την απόφαση της Τουρκίας να μην συμμετέχει στις επαφές και συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το παρελθόν εξάμεινο. Νομίζω είναι μια χαμένη ευκαιρία να ξεκινήσει η διαδικασία ε, εξομάλυνσης, σε πάση περιπτώσει, των σχέσεων ε, Τουρκίας-Κύπρου αρνήθηκε η Τουρκία να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της πλήρους εφαρμογής του συμπληρωματικού πρωτοκόλου της Άγκυρας. Και αυτό ε, επηρεάζει σε βάθος τις διαπραγματεύσεις. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία. Πρέπει να σταματήσω. Ναι. Συμπέρασμα. Ε, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τις ιδέες τους που έκαναν στις προτάσεις, στις απολογίες προφανώς δεν μπορούσα να υιοθετήσω τα πάντα. Δεν θέλω να φτιάξω χριστουγεννιάτικο δέντρο τελικά, έκθεση θέλω που να μπορεί να διαβαστεί. Και ελπίζω πραγματικά το παρόν ψήφισμα να είναι δίκαιο, αντικειμενικό και να δίνει μια ισόρροπη προσέγγιση. Λυπούμε. Δεν βλέπω τον συνάδελφο Βαν Μπάλεν εδώ, γιατί διάβασα στις εφημερίδες ότι θα ερχόταν. Τον είδα και στην τηλεόραση που έλεγε ότι θα έρθει για να συζητήσει μαζί μου. Γιατί θέλει να σταματήσει τι διαπραγματεύσεις που δεν θέλω εγώ. Αλλά δεν τον βλέπω. Τι να κάνουμε και άλλη χαμένη ευκαιρία του κυρίου Φαντάλ. Γελάνε οι Ολλανδοί συνάδελφοι, αλλά πρέπει να το πω εδώ κάποια φορά αυτό δημόσια και στο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους υπολείπους συναδέλφους παρόλα αυτά που είναι παρόντες. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφοι. 14 εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των ε, αγροτών. Οι σκιώδεις εισηγητές θα έχουν 3 λεπτά ο καθένας. Όλοι οι υπόλοιποι από 1,5 λεπτό. Πρώτα απ' όλα η κυρία Φλότρο, της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε την έκθεση της ΡΙΑ, της κυρίας Φαμανρόιτεν, μετά από πολυάριθμες συζητήσεις και πραγματικά την ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κατέβαλε. Χωρίς ε, να διστάσει, να κοπιάσει για να καταλήξουμε σε πολιτικούς συμβασμούς. Έχουμε λοιπόν ένα κείμενο και ένα ε, και πλήρες για ένα σύνολο ζητημάτων. Ήταν ισόρροπη η διατύπωση. Δεν ήταν απλό γιατί τα ζητήματα που θίγονται σε αυτή την έκθεση είναι τα περισσότερα ευαίσθητα και θα μπορούσαν εύκολα να δώσουν αφορμές για διαφιλονικίες. Οι διατυπώσεις λοιπόν των περισσότερων τροπολογιών που αφορούν το άνοιγμα κεφαλαίων, που αφορούν το θέμα των Κούρδων, την ελευθερία έκφραση, το θέμα των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων, την καταπολέμηση τη διακριτική μεταχείριση, ιδίω βάσει του σεξουαλικού πρωτοστατολισμού, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η κατάσταση των γυναικών, όλα αυτά είναι ευαίσθητα ζητήματα. Ζητήματα που νομίζω ότι αναφέρονται με πολύ συνέπεια και ακρίβεια στο έγγραφο. Ε, είναι σημαντικό το κείμενο αυτό να αποτελέσει εργαλείο εύχριστο και για την Τουρκία και χρήσιμο και για τις χώρες μας. Χρήσιμο λοιπόν για όσους θέλουν να προωθήσουν τη δημοκρατία στην Τουρκία και οι οποίοι θέλουν να έχει δυναμικό χαρακτήρα η διαδικασία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πραγματικά η έκθεση αυτή του Κοινοβουλίου δίνει τη δυνατότητα να αναφερθούμε τις εθνοτικές, ε, τις εθνικιστικές και τις αυταρχικές, απολυταρχικές τάσεις που μπορεί να εκδηλωθούν από καιρούς καιρών. Η Τουρκία σήμερα ζει μια πολιτική περίοδο καθοριστικής σημασίας για την ε, δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και αυτό γιατί η συνταγματική διαδικασία είναι σημαντική, εδώ πραγματικά κάνει έκκληση η έκθεση στους ε, ενδιαφερόμενους και τους συμμετέχοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να δημιουργηθεί μια νοοτροπία, μια κουλτούρα συνένεσης, ε, συμφιλίωσης που πρέπει να υιοθετήσουν όλες οι παρατάξεις στην Τουρκία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην, ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να βρεθεί μια λύση στο κουρδικό ζήτημα. Πολύ σημαντικό λοιπόν και εδώ η έκθεση πραγματικά προσφέρει επιχειρήματα και στήριξη σε όσου θα ήθελαν να απαλλαγούν από τους εθνικιστικούς θύλακες ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και δημοκρατισμού της Τουρκίας. Πραγματικά λοιπόν εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις διάφορες διατυπώσεις που εξεπρέθησαν μέσω των συμβαστικών τροπολογιών, χάρη στις προσπάθειες της Ισγήτριας. Η έκθεση αυτή καταφέρνει Μάλλον έρχεται σε μια στιγμή όπου στην Γαλλία και στη Γερμανία τον περασμένο και μήνα είχε εκφραστεί βέτο και εδώ μπορεί να υπάρξει μια νέα όθηση στις δημοτεύσεις. Υπάρχουν και κάποια σημεία για τα οποία δεν είμαστε πλήρω ικανοποιημένοι, ιδίω ό,τι αφορά το κυπριακό ζήτημα. Νομίζω η Κύπρο σήμερα έχει έναν πρόεδρο που δείχνει εξαιρετικό κουράγιο, εξαιρετική τόλμη και έχει και έκτακτα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Βεβαίω πρέπει να εξηγιάνει την οικονομία, να διτηρήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να δώσει ανάκαμψη στη διαδικασία για την επανένωση του νήσου. Νομίζω λοιπόν ότι από αυτή τη σκοπιά το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αποστείλει μηνύματα ηχηρά, ηχηρά προς... με, για, για, με τη στήριξη που εκφράζει σε αυτή την πολιτική βούληση με τους παρατηρητές ε, της ε, τουρκικής κυπριακής δημοκρατίας. Αυτό θα, θα μπορούσε να είναι μια πρώτη έκφραση για να στηρίξουμε τη νέα πολιτική ομάδα που έχει αναλάβει τα Ινία στην Κύπρο. Και για την επανένωση, ολοκληρώνω εδώ, η επανένωση θα έχει σημαντικότατες οικονομικές ευεργετικές συνέπειες στην περίπλοκη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει την σήμερα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, δεν μπορώ να δεχτώ υπερβάσεις του χρόνου για κανέναν. Έχουμε και άλλο σημείο να συζητήσουμε και το μεσημέρι στις 12 θα έρθει ο Επίτροπος Φούλε. Δεν μου αρέσει να διακόπτω τους ομιλητές, δεν είναι κομψό, αλλά υποχρεούμε να το κάνω, γιατί πρέπει όλοι να προλάβουν να μιλήσουν. Σας παρακαλώ λοιπόν, παραμείνετε στα όρια του χρόνου σας. Ο κύριος Ομπιόλ. Για τρία λεπτά. Ελπίζω ε, να μην ξεπεράσω το χρόνο μου. Πρώτον, στην πρώτη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας είχα πει ότι ήταν καλό το προσχέδιο και δεν το έκανα αυτό για λόγους φιλοφρόνησης. Είναι ευφύς εγωισμός αυτό. Γιατί όταν κανείς διαφωνεί, ε, μπορεί τελικά συζητώντας να συνεννοηθεί για μια καλή βάση. Και αυτή τη βάση τη βρήκαμε. Λοιπόν, δίνεται μια όθηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στη διαδικασία διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εφτά χρόνια διαρκεί αυτό με σκαμπανεβάσματα και αντιφάσεις. Ε, βεβαίως, στην Τουρκία έχει υποστεί ε, πλήγμα υποστήριξη κοινή γνώμη, αλλά ε, είναι θετικές οι μεταρρυθμίσει και η διαδικασία στην Τουρκία. Επίσης έχουν διατηρήσει μια ευρωπαϊκή προσήλωση που μπορούμε ε, να τη θεωρήσουμε σημαντική. Η δική μας στόχη ποιοι ήταν. Να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τη σημερινή ευκαιρία. Όπως είπε και η Ελέν προηγουμένως, υπάρχει κάποια αλλαγή τώρα στη θεώρηση ορισμένων κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ένωσης είναι πιο ανοιχτή, πιο ρεαλιστική, πιο πραγματιστική η στάση τους. Από την άλλη υπάρχει μια τεράστια περιφερειακή κρίση στη χώρα που τους υποχρεώνει να εργάζονται πιο στενά για καλύτερες σχέσεις και καλύτερη συνεργασία. Στη συνέχεια, και δεν το λέω με λόγους κατά σειρά σπουδαιότητας, υπήρξε μια, μια περίπλοκη περίοδος, αλλά ενθαρρυντική ε, στις διαπραγματεύσεις με τους Κούρδους και προσπαθήσαμε να βρούμε όσο γίνεται μεγαλύτερη συνένεση και ευρύτερη υποστήριξη από το Κοινοβούλιο για την έκθεση. Πάντα σκεπτόμενοι τις επιπτώσεις και τις συνέπειες τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Να μην δίνουμε απλώς μαρτυρίες των απόψεών μας. Να ξέρουμε και το μετά. Θελήσαμε να υποστηρίξουμε τη διαδικασία χωρίς αναβολές. Υποστηρίζουμε το άνοιγμα νέων κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις ε, ε, θεωρούμε απαραίτητες ε, πρόοδους στην ελευθερία της έκφρασης του τύπου, του συνεταιρίζεστε και του συνέρχεστε. Επίσης, να παραμείνει η διάκριση των εξουσιών και ε, ποντάρουμε σε ένα σύστημα δικαιοσύνης ε, ανεξάρτητο με διαφάνεια ε, αμεροληψία. Υποστηρίζουμε ε, τις συνομιλίες της κυβέρνηση κυβέρνησης με τον Οτσαλάν για μια ειρηνική και μόνιμη λύση για να σταματήσει η βία και υποστηρίζουμε τη διαδικασία θεώρησης του συντάγματος. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Νομίζω ότι κάναμε δουλειά ίσως βαριά, μακροχρόνια, αλλά που στέφθηκε με καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταφ, παρακαλώ. Um, Πρόεδρε, η ομάδα Άλντε στηρίζει θερμά και ευρέως το σχέδιο έκθεσης. Λυπούμεθα που το 2012 η Τουρκία μοιάζει να έχει στραφεί πλήρως και να δίνει έμφαση στα εσωτερικά της προβλήματα. Χάνει το δυναμικό ε, των ευρωπαϊκών προοπτικών της και σχέσεων. Είναι καθοριστική περίοδος αυτή της κρίσης στην Μέση Ανατολή, στην ε, Αφρική Νοτίου της Σαχάρα, στο Σαχέλ και στην Μεσόγειο. Η Τουρκία θα μπορούσε να ευθυγραμμίσει την εξωτερική πολιτική της και την πολιτική ασφαλείας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία ο Πρωθυπουργός Ερντογάν να προσκληθεί στην ε, Σύνοδο του Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθεί η, ασφάλεια, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ως προς την συνταγματική μεταρρύθμιση, ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργό Ερντογάν ζητά προεδρική δημοκρατία, προεδρικό καθεστώς. Αυτό νομίζω ενέχει κινδύνους για την ε, καλλιέργεια της πολυφωνίας και της δημοκρατίας. Διότι θα οδηγήσει σε κατάρρευση τις διακομματικές συνομιλίες και θα δώσει ιδιαίτερα κεντρικό χαρακτήρα στην διοργάνωση της χώρας. Κάτι που δεν εξυπηρετεί την ε, εξέβρεση λύσης ούτε για το κουρδικό στο ίδιο πλαίσιο. Λυπούμαστε για τις απολυταρχικές τάσεις και τις ε, κοινωνικά συντηρητικές ε, εκφράσεις που ολένα και αυξάνονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Επίσης, ε, λυπούμεθα ιδιαιτέρως για την απουσία πρόοδου στο κυπριακό ζήτημα. Εάν υπάρχει κάποια κατάλληλη στιγμή για να δείξει μια καλύτερη στάση προς το κυπριακό ζήτημα και κοντύτερα στην εξέφραση λύση η Τουρκία, αυτή η στιγμή είναι τώρα. Ευχαριστώ. For the time. Ευχαριστώ που παρεμένατε στα όρια του χρόνου, κ. Φανόντε. Absent, Mr. Χατζηγεώργιου. Ο κ. Χατζηγεωργίου. Next time. Λυπούμε που η παρέμβασή μου δεν έπαιρνε της παρέμβαση του κυρίου Βανόρντεν. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσω από την γενική εικόνα του αν η Τουρκία έχει προοπτικές ένταξης ή όχι. Κατά την άποψη μου, για να μην γελιόμαστε ούτε εμείς ούτε να ξεγελούμε τους ίδιους τους Τούρκους και την τουρκική κυβέρνηση, δεν υπάρχουν πολλοί στην Ευρώπη κράτη ή και λαοί που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ένταξη της Τουρκίας και είναι γνωστό και ένα ρεύμα κατά της ένταξης και στην ίδια την Τουρκία. Όσοι λοιπόν κατά την άποψή μου έμειναν να υποστηρίζουν ουσιαστικά και ένθερμα την διαδικασία ένταξης της Τουρκίας πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτό περνά από τη Λευκοσία. Χωρίς λύση του Κυπριακού ή χωρίς ισχυρές ενδείξεις ότι η Τουρκία κινείται προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού οι ελπίδες για τη διαπραγματευτική διαδικασία εξανεμίζονται. Το δεύτερο που έχω να πω, επειδή ελέγχθη κάτι από την κυρία Φλότρ για παρατηρητές από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, να είμαστε ξεκάθαροι. Στα κατεχόμενα πλέον η πλειοψηφία είναι έπικη. Είναι Τούρκοι που κατοικούν παράνομα ε, στην, στην κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου και σε περίπτωση απόφασης να υπάρξουν εδώ παρατηρητές, δεν θα είναι παρατηρητές από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, θα είναι παρατηρητές της Τουρκίας. Και το τελευταίο, υπάρχουν πράγματι ενδείξεις ότι κάτι γίνεται σε σχέση με το κουρδικό. Ελπίζω και εύχομαι να προχωρήσει αυτό το πράγμα γιατί θα είναι προς όφελος και των Κούρδων και των Τούρκων. Υποψιάζομαι όμως ότι ο Πρωθυπουργός Εκτογάν παίζει και σε αυτό το θέμα ένα παιχνίδι να κερδίσει τις ψήφους των Τούρκων για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος σε ένα προεδρικό σύστημα στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Van Orden, you have minutes. Ευχαριστώ κύριος Βανόρντεν. Orden. Τρία λεπτά. Ε, και να τηρήσετε το χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, Είχα ε, επισκέψει από εκπροσώπου τη εκλογική μου περιφέρεια και ήταν σημαντικό να μιλήσω και μαζί του, αλλά και το θέμα σα εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κατά πρώτον, ανασυγχαρότηρια. Έχει κάνει εξαιρετική έκθεση, νομίζω. Ω συνήθω, βέβαια. Το περιμέναμε αυτό από τη ΡΙΑ. Εντάξει, δεν συμφωνούμε σε όλα. Αυτό δεν μα εκπλήσει. Αλλά συνολικά η έκθεση είναι καλή. Υπάρχει απλώ ένα ζήτημα που θέλω να θίξω το Κυπριακό. Ξέρω ότι θα μου πουνε οι περισσότεροι έκθεση αυτή αφορά την ένταξη της Τουρκίας και όχι την Κύπρο. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος είναι καθοριστική για το αν θα επιτελεστεί πρόοδος στη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας. Να είμαστε σαφείς. Ακόμη και αν δεν εκφράζεται ρητός πάντοτε, ισχύει. Και μια συγκεκριμένη παρατήρηση θέλω, στην οποία θέλω να, επιστήσω την προσοχή σας. Το θέμα της εκπροσώπησης των Τούρκο-Κυπρίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Βάσει των συνθήκων, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα της άμεσης αντιπροσώπησης εδώ στο Κοινοβούλιο. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υποσχεθεί και επαφές και εκπροσώπηση στους Τουρκοκυπρίους. Για κάποιο λόγο δεν έχουμε τηρήσει την ε, υπόσχεσή μας αυτή. Για λόγους που πολλοί από εμά προφανώς κατανοούν. Όμως έχει φτάσει η στιγμή να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες στο θέμα της εκπροσώπησης. Πρέπει να βρούμε μια λύση εδώ βεβαίως. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που εκκρεμούν. Όμως θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Διότι έχω μια συγκεκριμένη τροπολογία. 317. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε εδώ ένα καλό συμβιβασμό ώστε να, διατηρήσουμε τα βασικά στοιχεία αυτής της τροπολογίας και ελπίζω, Πρόεδρε, να υπάρξει στήριξη για την τροπολογία αυτή. Έστω και από συμμάχους που δεν έχω συνήθους. Θα ήλπιζα σε ευρύτερη στήριξη από την Επιτροπή αυτή για την τροπολογία αυτή και για μια τέτοια συμβαστική μάλιστα τροπολογία. Ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή της Ρίας αυτό και ήθελα επίσης να δείξει ευελιξία εδώ για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σαλαβράκος για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Όιμεν διότι κατάφερε παρά τη δυσκολία και ευαισθησία αυτού του θέματος να μας παρουσιάσει μια ισορροπημένη και σχεδόν πλήρη έκθεση. Μια έκθεση που εντοπίζει τις ατέλειες του συστήματος διακυβέρνησης στην Τουρκία και των κοινοτικών δομών στη χώρα αυτή. Ε, βεβαίως ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος το οποίο επί σειρά ετών είχε εμφανή και αμφανή κέντρα εξουσίες τα οποία ακόμη και σήμερα είναι ενεργά όπως δείχνει η υπόθεση Σεργένικων και η πρόταση του κεντρικού εισαγγελέου της Κωνσταντινούπολης χθε για επιβολή μεγάλων ποινών σε πολλούς στρατιωτικούς ηγέτες προηγουμένως. Ε, δεν θα συμφωνήσω βεβαίως ε, με την πρόταση του κυρίου Βανόλτεν. Το όλο πνεύμα της εκθέσεως είναι να φέρει μια ισορροπία και να σεβαστεί τόσο την Τουρκία σαν μεγάλο κράτος, όσο και τις παρενέργειες που έχουν ορισμένες ε, πολιτικές της Τουρκίας σε άλλα κράτη. Το παίρνει η έκθεση εξαπαλών ονείχων και με πολύ σύνεση και ε, πολλή σοφία. Εάν μπουν ρηματικές ε, τροπολογίες όπως η 317 του κυρίου Βανόρντεν δημιουργούν μείζον πρόβλημα από εκείνο που μπορούν να λύσουν ή επιχειρούν να λύσουν λαμβανωμένου υπόψη μάλιστα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε των τουρκοκυπρίων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Δεν το αποκρούει το θέμα είναι να εντοπιστούν ποιοι είναι οι τουρκοκύπριοι πολίτες και ποιοι είναι οι έπικοι οι οποίοι είναι αμυγός Τούρκοι πολίτες. Ε, βεβαίως η χώρα χρειάζεται πολύ δρόμο ακόμη και όσον αφορά τις ε, τροπολογίες θα ήθελα να επισημάνω και να συστήσω αν είναι δυνατόν στην κυρία Συγκήτρια στην συμβιβαστική τρία τη λέξη illegal, illegal immigration να την αντικαταστήσουν που αντικαθιστά με irregular immigration να την επαναφέρουν. Ε, στη Συμβαστική 8 ε, θεωρώ ότι η αναφορά που γίνεται στις επιθέσεις στην αρμανική κοινότητα θα μπορούσε να ενσωματεθεί στη Συμβαστική 21 και να παροτρύνουμε την Τουρκία να φέρει το θέμα στην δικαιοσύνη όπως αρμόζει. Χαιρετίζω ιδιαίτερως τη Συμβαστική 15 που αφορά το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, καθώς επίσης και τη σύμβαστική 18, που γίνεται αναφορά στη Σύμβαση του ΟΕΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και την ανάγκη για άμεση υπογραφή και κύρωση του πρωτοκόλου από πλευράς της Τουρκίας. Ε, παρατηρώ ωστόσο ότι σε σχέση με άλλες χρονίες δεν γίνεται αναφορά στις συνεχόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου καθώς και στο κάζους Μπέλι έναν της Ελλάδος που πλήττει την κατάσταση στην νότιο-ανατολική Μισόγειο και στη σχέση γειτονία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστούμε. Οι επόμενοι ομιλητές θα έχουν 1,5 λεπτό. Η κυρία Βοτκούρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, σύντομα σχόλια. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την κυρία Όμεν που κάθε χρόνο ασχολείται με αυτή την περίπλοκη έκθεση και νομίζω κάνει πολύ καλή δουλειά. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι και ελπίζω φέτος να μην συμβεί ότι αυτό που συζητάμε είναι έκθεση για την Τουρκία η Τουρκία από μόνη της είναι αρκετά περίπλοκη για να ασχοληθεί μαζί τη και δεν θα πρέπει να αποκατασταθεί η έκθεση και να γίνει έκθεση για την Κύπρο. Δεν είναι για την Κύπρο η έκθεση, είναι για την Τουρκία. Ε, να δούμε λοιπόν ποια είναι η αξία και ποια είναι τα προβλήματα της Τουρκίας. Το επόμενο πρόβλημα. Συμφωνώ με τη Ριόμεν Ρόιτεν ότι χρειάζεται ε, τα κεφάλαια 23 και 24 να ε, ξαναρχίσουν οι προσπάθειες. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολύ σημαντικό, τα δικαιώματα των ανηλίκων, των γυναικών, των ΛΟΑΔ, ε, ελευθεροτυπία. Θέλουμε πραγματικά να πιέσουμε την Τουρκία, ε, θα πρέπει να γίνει με διάλογο και ανοίγοντας αυτά τα κεφάλαια, 23 και 24. Και η Τουρκία αν δεχτεί, αν εγκρίνει και τη τέταρτη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, θα έχει προχωρήσει πολύ και βεβαίως και το θέμα του συντάγματος. Σταματώ εδώ, έχω να πω και άλλα, αλλά ευχαριστώ που μου δώσατε χρόνο γόρευση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σοφοκλέους παρακαλώ. Οφείλω να παρατηρήσω ότι γίνεται μια προσπάθεια από την εισηγήτρια να εκφράσει κατά τρόπο ισόρροπο τις θέσεις της για την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Οφείλω όμως επίσης να εκφράσω και τις διαφωνίες μου αναφορικά με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και αναφέρονται συγκεκριμένα. Στην άρση της λεγόμενης απομόνωσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, το αίτημα για συμμετοχή τουρκοκυπρίων παρατηρητών στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο απευθείας εμπόριο, στο ζήτημα της Επιτροπής Αγνωμένου και άλλες. Λόγω περιορισμένου χρόνου δεν μπορώ να κάνω εκτενή αναφορά σε όλες τις τροπολογίες, με τις οποίες διαφωνώ σεβόμενος τον χρόνο που μου δίδεται, θα ήθελα να τοποθετηθώ επιγραμματικά στα εξή. Το θέμα στο πευθείας εμπορίου εκκρεμεί και βρίσκεται παγωμένο με την απόρριψη τη προτινόμενη νομική βάση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Συνεπώ, δεν είναι δυνατό και συνετό να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Το ζήτημα των τουρκοκυπρίων παρατηρητών, πιθανών και επίκων, Στι εργασίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προωθεί την διαίρεση τη Κύπρου. Οι Τουρκοκύπροι έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε στι ευρωεκλογέ, άρα δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Επιτρέψτε μου απαντώ στον Βανόρτε που φαίνεται επιλεκτικά κατά καιρού ξεχνά αυτή την πάγια σταθερή θέση. Η λεγόμενη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να συνδέεται με την εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου, γιατί αυτό από μόνο το αποτελεί standalone προπόθεση για επίτευξη πρόοδου στι ενταξιακέ διαπραγματεύσει και δεν μπορεί να συνδέεται με άλλα ζητήματα. Αναφορικά με το ανοιχτό ζήτημα των αγνοωμένων, η Τουρκία πρέπει οφείλει να συνεργαστεί επικοδομητικά με την ΔΕΑ και να επιτρέψει πρόσβαση σε όλε τι στρατιωτικέ ζώνε. Τέλο και κλείνω, επιθυμώ να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με μία προπόθεση ότι περνά μέσα από τη λύση του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Mr. Watson, Ευχαριστούμε, κύριος Βότσον. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την ε, εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την έκθεση αυτή. Πρόεδρε, η εντύπωσή μας είναι ότι πρέπει να εξεύρουμε κάποια ισορροπία σε ορισμένα ζητήματα ακανθόδη. Ισορροπία που να αντικατοπτρίζει και το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην νήσο. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να βρει κάποια λύση για τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων της νήσου. Θα είναι απογοητευτικό. Αυτό θα γίνει πλέον ζήτημα μόνο των Ηνωμένων Εθνών. Η ομάδα μου στηρίζει τις τροπολογίες που προωθούν μια ισόρροπη στάση στα θέματα αυτά σε όλη την έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάποιοι από τους συναδέλφους καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να παρεμποδίσουν τόσο την επανένωση της Κύπρου όσο και την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμάς η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται ο κύριος Βανόρτεν και η κυρία Φλότρ να μιλάνε για εκπροσώπους της τουρκικής βόρειας δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό συνιστά τα φόπλακα στην προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία όταν θέλουν να εισαγάγουν εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσώπους ενός άλλου κράτους, της τουρκικής βόρειας δημοκρατίας. Ε, να, να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια για ένταξη τη Τουρκία από εκεί και πέρα. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταβάλει προσπάθειε για την ομαλοποίηση των σχέσεων τη με την Τουρκία και φάνηκε στη διάρκεια τη Προεδρία. Έχει κάνει ένταση, ε, αίτηση για ένταξη στο PFP και η Τουρκία αντιτίθεται. Κάτι που θα ομαλοποιούσε τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση-ΝΑΤΟ. Η Τουρκία και οι φίλοι της εδώ μέσα κάνουν κάθε προσπάθεια να καταστρέψουν την οποιαδήποτε πρόοδο καταβάλει η Τουρκία στο εσωτερικό της. Επισημαίνω ότι στην συμβιβαστική 18 και 24 υπάρχει μεγάλη αντίφαση γιατί από τη μια καλείται η Τουρκία να εφαρμόσει το δίκαιο της θάλασσας και να σταματήσει να παρενοχλεί οι γαλλικές εταιρείε στην τοτάδα Αμερικάνικες που κάνουν έρευνες στην θαλάσσια ε, ε αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και από την άλλη καλείται η Κύπρος να ανοίξει το, 15, μα, το κεφάλαιο 15. Γιατί να το ανοίξει το 15 όταν εμείς καλούμε την Τουρκία να συμμορφωθεί. Γιατί δεν βλέπουμε ότι η Τουρκία παρεμποδίζει την ένταξη τη Κύπρου και του Ισραήλ στην ε, Διεθνή Οργανισμό Ανανεωσίμων Πηγών Ενεργεία, να του ανοίξουμε εμεί το κεφάλαιο 15. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο και να σταθούμε πιστοί στο ευρωπαϊκό δίκαιο αν θέλουμε η Τουρκία να κάνει κάποιο βήμα. Διαφορετικά αυτό είναι η ταφόπλακα. Ευχαριστώ. Thank you, Ms. please. Στο κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Η... Συγχαίρω καταρχήν την κυρία Νόμενη για τη σκληρή δουλειά για αυτή την έκθεση. Η Τουρκία αντιμετωπίζει τρία καυτά προβλήματα, τρία αγκάθια στην ενταξιακή της πορεία. Το πρώτο είναι η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ίδια τη χώρα και εδώ χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και επιτάχυσή τους. Το δεύτερο είναι το κουρδικό και χαιρετίζω τη διεξαγωγή συνομιλιών. Το τρίτο είναι το κυπριακό. Η Τουρκία κάνει ένα μεγάλο λάθο δεν αναγνωρίζει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς δεν έχει εφαρμόσει το πρωτόκολλο που είναι συμβατική της υποχρέωση. Βλέπουμε εδώ το φιλοτουρκικό λόπι να προωθεί πολλές τροπολογίες και να επαναφέρει το μύθο περί απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, να ζητά άνοιγμα κεφαλαίων και μάλιστα τώρα μπαίνει κάτι καινούριο, ένα εμπόδιο να υπάρχουν δίθεν ε, Τουρκοκύπροι παρατηρητές. Σας λέω αυτά είναι εγκληματικά λάθη και αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην φέρει καινούργια εμπόδια. Η Τουρκία για να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρώπη είναι έχει δρόμο να διανύσει και πρέπει να συμβαστεί συμβατικές της υποχρεώσεις. Πέραν τούτου, θεωρώ ε, ότι το απευθείας... Έχω ανάμιση ή ένα λεπτό. Ε, Λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στο φιλοτουρκικό λόπι είναι, επαναφέρονται διαρκώ τα ίδια πράγματα για την απομόνωση, για τα απευθεία εμπόρια και τέτοια, ενώ η Κύπρο σέβεται τη συνθήκη τη Νίκαια και αν θέλουν οι Τουρκοκύπροι να συμμετέχουν στι ευρωεκλογέ, είναι ελεύθεροι να το πράξουν. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε και αν θέλουν στι επόμενε ευρωεκλογέ μπορούν να κατέλθουν ω υποψήφοι. Η κυρία Κοπά, παρακαλώ. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα σημεία. Ε, ξεκινώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ρία Ουμερόιτεν για μια εξαιρετική δουλειά για μια ακόμη χρονιά. Το πρώτο μου σημείο αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τραγική στην Τουρκία Δυστυχώς δεν έχουμε δει καμία βελτίωση το τελευταίο διάστημα, αλλά εξακολουθεί να παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης. Και είναι πολύ θετικό ότι τόσο σε τροπολογίες ε, όσο και στο ίδιο το κείμενο έχουμε ρητές αναφορές. Δεύτερο σημείο η Κύπρος. Η Κύπρος περνάει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδό της στην ιστορία της, ας μην βάλουμε νέα βάρη στους ώμους του νέου Προέδρου, του κύριου Αναστασιάδη, που προσπαθεί να κρατήσει τη χώρα του όρθια. Τροπολογίες οι οποίες μπαίνουν την τελευταία στιγμή, το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν. Το κάνουν δύσκολο, κάνουν αδύνατη οποιαδήποτε έναρξη διαλόγου για το Κυπριακό. Αποτελούν εμπόδια και δεν διευκολύνουν καθόλου τη διαδικασία. Τρίτο σημείο ελληνοτουρκικές ε, σχέσεις. Ο Πρωθυπουργό πήγε στην Τουρκία, τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και συνεχίζει να μην επικυρώνει και να ε, δέχεται την άγκλος το δίκαιο της θάλασσας. Μέχρι να λυθεί αυτό το ζήτημα, τα προβλήματα παραμένουν ανοιχτά. Ευχαριστώ. Thank you. Ms. Giannaco, one minute and Ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ήδη πολλοί συνάδελφοι Έλληνες έθεσαν τα προβλήματα. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η τροπολογία 355, η οποία αναφέρεται στο κάζους Μπέλη, δηλαδή στην απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ότι αν η Ελλάδα εφαρμόσει διεθνείς συμφωνίες όπως είναι η Άγκλος, η Τουρκία θα κηρύξει πόλεμο. Αυτά είναι πρωτοφανή. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει μια χώρα της Ένωσης και σε άλλη μια την απειλεί με πόλεμο. Και δεύτερον, οι συνεχείς υπερπτήσεις και παραβιάσεις του εναερού χώρου. Θέλω να παρακαλέσω την κυρία Όουμεν, της οποίας δυσκολέψαμε τη ζωή, κάνοντας τόσες πολλές τροπολογίες και την οποία αυτονοεί το συγχαίρω διότι είναι εξαιρετική επί πολλά χρόνια στην έκθεση για την Τουρκία, να τη δεχθεί. Και το δεύτερο είναι το θέμα της δίθεν εκπροσώπησης των τουρκοκυπρίων. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μπορούν κάλλιστα να εκπροσωπηθούν. Τι θα εκπροσωπούν αν έρθουν οι παρατηρητές. Ένα κράτος που δεν υπάρχει, που δεν αναγνωρίζεται από την Ένωση. Εγώ νομίζω ότι όσο εξερχόμεθα των κανόνων και των αρχών της Ένωσης ε, στην πολιτική μας συμπεριφορά, τόσο δυσκολεύουμε τις καταστάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Last speaker, Mr. Peterle, please. Ευχαριστούμε, ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την κυρία Όμεν Ρόιτεν για την έκτη έκθεση πρόοδου Έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι είναι και ρεαλιστικέ και πολύ ισορροπημένε στη διατύπωση οι εκθέσει τη. Αυτή η έκθεση έχει όμω και πολλά αισιόδοξα στοιχεία. Κάπου αναφέρεται ο όρο welcome, καλωσορίζουμε. Και μάλιστα αναφέρεται συχνότερα από ότι ο όρο we regret, λυπούμεθα. Εδώ θα συμμεριστώ την πίστη, την ε, ανάγκη που εκφράζει και η συγκήτρια να αναλυθούν νέες δεσμεύσεις από τις δύο πλευρές. Θέλουμε να πάρουν μια νέα τροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και θέλω, γι' αυτό παρακολουθούμε στενά τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Είναι σημαντικό η διαδικασία αυτή να συνεχίσει με του ρυθμού, αλλά επίσης σημαντικό είναι να συνεχίσουν και οι συνομιλίες με τους Κούρδους. Περιμένουμε να γίνει κάποια πρόοδο εδώ, εδώ και πολύ καιρό. Ως προς το Κυπριακό πιστεύω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο από τη σκοπιά τη διαδικασία τη προσχώρηση. Είναι ένα θέμα που πρέπει να επιληθεί ούτω ή άλλω ασχέτω από τη διαδικασία προσχώρηση. Και αυτό θα ελάφρυνε και πάρα πολύ την έκθεση, εάν βλέπουμε το θέμα ξεχωριστά. Επίση, και στο παρελθόν ε, είχαμε ταχθεί υπέρ του να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα που να οδηγήσει σε επίλυση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην εισηγήτρια που δέχτηκε και μια από τι τροπολογίε μου. Για την απελευθέρωση του Βορείου. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιαμόνι Ρόιτερ. Δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω, αν μου επιτρέπετε. Αυτό που προσπαθούμε ανέκαθεν είναι να γράφουμε μία έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας, αντικειμενική, ανοιχτή και δίκαιη. Και από το θέμα της δικαιοσύνης, αν το κοιτάξουμε, πρέπει να πούμε όντως ότι δεν είναι έκθεση για την Κύπρο. Αν κοιτάξετε τον κατάλογο ψηφοφορίας μου, θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότερες τροπολογίες που καλύπτουν πάρα πολύ ειδικά θέματα στις σχέσεις Τουρκίας-Κύπρου έχουν αρνητικό πρόσημο. Δεν θέλω να τις εγκρίνουμε, αλλά για να μιλάμε και για δικαιοσύνη. Πάντα θα πρέπει να κοιτάμε και τις τροπολογίες 3, 11, ε, ε, 17 και 19. Και όπως είδαμε και εδώ, είναι μεγάλη συζήτηση επί αυτών των θεμάτων. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπερψηφιστούν. Τι θα ήθελα να δω εγώ. Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία τώρα για τη νέα κυβέρνηση, για εξομάλυνση ε, των σχέσεων μεταξύ των δύο τμήματων της νήσου. Αυτό είναι νομίζω ο δικός μας στόχο. Προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Και πάλι δεν είναι έκθεση για την Κύπρο. Και το λέω αυτό προς τον συνάδελφο Βότσον. Για τα ενεργειακά, αν δούμε την παράγραφο που προτείνει, καλύπτονται όλα. Αλλά σας παρακαλώ, αφήστε τα αυτά τώρα και ακολουθήστε το δικό μου κατάλογο ψηφοφορία. Γιατί και η ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να είναι δίκαιη και η τουρκική πλευρά θα πρέπει να είναι δίκαιη. Αλλά αν δούμε το ζήτημα της Κύπρου, και εκεί χρειάζεται να επιδεικνύουμε δίκαιη στάση. Και καθόλου δεν συνιστώ να υποστηριχθούν οι τροπολογίες 3, 11, και 3, 19. Προτείνω καταψήφιση. Γιατί θα μπορούσαμε έτσι να παρεμποδίσουμε και να ενοχλήσουμε θετικές εξελίξεις. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, επόμενο σημείο είναι η έκθεση της κυρίας Φρανσίσκα Κατρίνα Μπραντνερ με τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή του ΙΕ για την ευθύνη προστασίας. Εκεί είστε, μάλιστα. Δεύτερη εξέταση της έκθεσης. 137 τροπολογίες και 18 συμβιβαστικέ τροπολογίε. Σα δίνω αμέσω το λόγο για την εισηγησή σα. Ίσως να περιμέναμε ένα λεπτάκι, Πρόεδρε. Okay, dear colleagues. Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, Όπως και ο Πρόεδρος είπε, είναι η δεύτερη φορά που συζητούμε εδώ στην Επιτροπή μας το θέμα αυτό. Και είχαμε έναν ε, σοβαρό αριθμό τροπολογιών, νομίζω οι περισσότερες πολύ καλές. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τους και όδης εισηγητές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και τις επικοδομητικές συνομιλίες χτες μόλις. Ε, ε, καταφέραμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες όπως είπατε. Είναι μακροσκελής ο κατάλογος των τροπολογιών μεν, αλλά φαίνεται να έχουμε κάποια κοινή ε, αντίληψη για τη σύσταση αυτή. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω την, τον εισηγητή της Επιτροπής Ντέβελ, τον κύριο Κάσμαν για την τοποθέτησή του και που οι δικέ του απόψει θα απηχηθούν με προφορικέ τροπολογίε, ε, των οποίων την έγκριση πραγματικά συστήνω Πολύ σύντομα επί τη ουσία. Βασικός στόχος ε, της σύστασης αυτής είναι να προωθήσει την διευκρίνηση των επιπτώσεων της ευθύνης αυτής για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, υλοποίηση της αρχής αυτής της ευθύνης για προστασία. Θέλω να βεβαιωθώ ότι ε, θα απηχηθεί σωστά η θέση του Κοινοβουλίου στην υλοποίηση της σύστασης αυτής, χωρίς όμως να ε, προδικάσουμε και να επηρεάσουμε το πώς θα διαμορφωθεί πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε επίπεδο ΟΗΕ η ερμηνεία της σύστασης. Στο επίπεδο του ΟΗΕ άλλωστε η διαδικασία βρίσκεται να εξελίξει. Υπάρχουν αρκετά καινοτόμα και ενδιαφέροντα στοιχεία που τα βλέπουμε και στις συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να τονίσω κάποια από αυτά. Θα πρέπει να ε, περιληφθούν κάποια από αυτά στο κεφάλαιο για την αρχή αυτή από την υπατική για την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ την υλοποίηση τη αρχή και την προστασία. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώ κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τηρήσει τι υποσχέσει τη ω προ την ε, ευθύνη προστασία. Επίση, πρέπει να συνεργαζόμαστε καλύτερα με του προέδρου αντιπροσωπιών, ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών, προκειμένου να εντοπίσουμε, να προλάβουμε, να εξηγήσουμε συγκεκριμένες ε, παραβιάσεις της ε, σύστασης αυτής. Επίση, η ειδική εντολή του Προσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, να συμπεριλάβει τέτοια r ε, σε στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην όλη δραστηριότητα της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Επίσης πρέπει να τονωθεί η συνιστόσα του πει στην προστασία δηλαδή σε όσα κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο κρεμή ζητήματα τα οποία ήθελα να τα θίξω προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Πρώτον, το θέμα των σχέσεων μεταξύ του RTP και των δράσεων για ανθρωπιστικούς λόγους. Στο διεθνές δίκαιο θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή εξισορρόπηση μεταξύ της σύστασης αυτής με την ερμηνεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανθρωπιστική δράση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να υλοποιήσουμε στόχους της ε, ευθύνη αυτής. Πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση των στόχων των δύο αυτών ε, σκοπιών, όπως το λέει και η έκθεση. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες μεταξύ μας ακόμη, δηλαδή πώς πρέπει να συσχετιστεί η σύστηση αυτή με τα όσα κάνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και εδώ θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι απόψει σα. Νομίζω ότι η ευθύνη για προστασία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στο διεθνές ποινικό δίκαιο, ακόμη και όταν ε, φτάνουν ενώπιον τη δικαιοσύνη, υπεύθυνοι για ανθρωπιστικές ε, εγκληματικέ ενέργειε και στο διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης. Θα ήθελα λοιπόν να λάβω τα σχόλιά σα Με μεγάλο ενδιαφέρον τα περιμένω και σα ευχαριστώ για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε για τη σύσταση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προκειμένου να μπορέσουμε και να είναι και εφικτό να ε, ακούσουμε τον Επίτροπο Φίλε στην ώρα του και για να μας δώσει και τις πληροφορίες που τόσο πολύ θέλουμε, ξέρω ότι έρχεται όπου να είναι, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για, το για την τεράστια δουλειά που έχει κάνει και να εκφράσω την ικανοποίησή μου. Διότι παρά κάποιε αποκλίνουσες απόψεις που και η ίδια τώρα μόλις μα θύμισε, κατάφερε να μας δώσει ε, ε, ικανοποιητικότατε συμβαστικές τροπολογίες. Έτσι, αποφεύγουμε και να διαταράξουμε την ε, επίσκεψη του κυρίου Φίλε. Θα υποβάλω κάποιε αποφορετικέ τοπολογίε, αυτό θέλω να το πω, για κάποια ζητήματα που τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Και ένα από αυτά έχει να κάνει με το ότι προτείνουμε και συστήνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνουν στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ να σκεφτούν τη δυνατότητα δημιουργία ενός κώδικα συμπεριφορά και τη, δική, τη χρήση του δικαιώματο ορνής κυρίας. Ένα από τα βασικά προβλήματα του ΟΗΕ. Για την περίπτωση γενοκτονιών ή εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά τη ανθρωπότητα, αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και επίση, μια δεύτερη τροπολογία, προκειμένου να ενισχυθεί η ιδέα ότι η αρχή ευθύνη για προστασία, η αρχή τη ευθύνη για προστασία μάλλον, θα πρέπει να ισχύει και για τις προσπάθειες εθνοκάθαρσης, τα εγκλήματα πολέτου και τις ανθρωπιστικές ε, εγκληματικές ενέργειες. για εθνοτικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, γεωστρατηγικούς λόγους όταν κάποια χώρα παραβιάζει την αρχή αυτή. Όταν αλλάζει το καθεστώς μιας χώρας λόγω χάρη. Το θέμα είναι αν εκεί γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές τις οποίες υπονοεί η ευθύνη για προστασία. Μαζί με το σημείο για τον κώδικα λοιπόν συμπεριφοράς, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σε περιπτώσεις όπως της Συρίας, αυτά οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Είναι πολύ μεγάλο όνειδος για την Ευρώπη να μην έχει αναλάβει εδώ καμία δράση και να μην κάνει τίποτα. Ε, τέλεια! Κυρία Μίνσκι, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Οι απόψει του ΕΛΚ για την έκθεση αυτή, για τη σύσταση τη ε, ευθύνη για προστασία. Να ευχαριστήσω κατά πρώτον την εισηγήτρια και του σκιώδει εισηγητέ ε, για την καλή συνεργασία που είχαμε για τη σύνταξη τη έκθεση. Νομίζω ότι φτάσαμε σε καλή συμβαστική λύση, καθώ στο κείμενο απηχεί τι θέσει των διαφόρων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Οπότε το ΕΛΚ θα στηρίξει το σύνολο τη έκθεση. Αυτό που εμείς ως βουλευτές επιδιώξαμε είναι να ξεκινήσει η συζήτηση για μια ευρωπαϊκή θέση ως προς την ευθύνη για την προστασία. Η έκθεση αυτή είναι ένα μόνο, ένα μόνο πρώτο βήμα στην όλη διαδικασία. Ελπίζω οι δικέ μα προτάσει να ληφθούν υπόψη και η σύσταση να υλοποιηθεί στο εγγύ μέλλον, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, λάβει ηγετική θέση στι διεθνεί συνομιλίε ω προ την αρχή τη ευθύνη για προστασία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σάκε. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι σύντομη, διότι έρχεται ο Επίτροπος. Και γιατί χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες δέχτηκαν ε, μέρος των τροπολογιών μας ε, τι συμβαστικέ τροπολογίε. Νομίζω ότι επιδιώκει η έκθεση αυτή να ενισχύσει τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναλαμβάνονται οι ευθύνε και πώ πρέπει να ασκείται το... η υποχρέωση αυτή. Η είναι σαφή η ανάγκη, νομίζω, εάν δούμε τι απειλέ υπάρχουν γύρω μα, τι απειλέ γενοκτονιών και εγκλημάτων κατά τη ανθρωπότητα. Είναι σαφέ ε, σε τόσε περιοχέ στον κόσμο τι συμβαίνει. Και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε την κατάλληλη και νομική βάση που πρέπει να είναι και σταθερή για να μπορέσει να υλοποιηθεί σωστά η σύσταση αυτή. Να τονίσω κάτι που το έθιξε και η ίδια η ότι σε πολλές από τις πρόσφατες συνομιλίες μας φάνηκε να υπάρχει σύγχυση, σύγχυση που ανέφεραν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και, και ανθρωπιστικών οργανώσεων και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ότι η χρήση τέτοιων προσχημάτων ε, αιτιολογιών στο ανθρωπιστικό έργο, μάλλον για ανθρωπιστικούς λόγους, μπορεί να βλάψει το έργο τους. Υπάρχει ε, ευθύνη και ε, βάση του ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, το Δίκαιο για τους Πρόσφυγες Οι νομικές βάσεις και αρχές που υπάρχουν ούτως ή άλλως ε, πρέπει να τονιστούν εδώ. Μην ξεχνάμε λοιπόν τι μερίμνες έχουν και αυτοί που εξέφρασαν τέτοιου είδους ανησυχίες. Πρόεδρος. Κάποιος άλλος. Άλλοι ομιλητές. Η Ευρωπαϊκή λοιπον τι μερημνες εχουν και αυτοι που Ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια που μας δίνει την ευκαιρία να σχολιάσουμε την έκθεση. Η συλλογιστική της ε, αρχής αυτής της ευθύνη για προστασία είναι φυσικά ευπρόσδεκτη και η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου το ίδιο. Στόχος είναι να προστατευτούν οι πολίτες από τα σοβαρά εγκλήματα ε, κατά της ανθρωπότητας ε, διεθνώς. Δύο ζητήματα μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε σχέση με την ε, ε, έννοια αυτή ως προς την βασική ανθρωπιστική δράση. Πρώτον, πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της αρχής R2P και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και τα πρωτογενή νομικά εργαλεία που είναι οι συμβάσεις της Γενέβης του 49. Ε, εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το R2P δεν έχει ακόμη το καθεστώς ε, διεθνούς ε, νόμου παρόλο που απηχείται σε διεθνείς κανόνες που ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνονται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ούτως ή άλλως υπάρχουν νομικές υποχρώσεις βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου διότι οι συμβάσεις της Γενέβης έχουν ακυρωθεί από όλα τα κράτη. Επιπλέον το πεδίο των υποχρεώσεων που προκύπτει από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι ευρύτερο από ότι τα εγκλήματα πολέμου που καλείται να αντιμετωπίσει η R2P. Επίσης η έννοια R2P θα πρέπει να μην επηρεάσει το ευρύτερο πεδίο υποχρεώσεων για τα κράτη, όπως προκύπτει από το Διεθνέ Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Και επίσης πρέπει να γίνει μια σαφής διάκριση μεταξύ της ε, σύσταση ευθύνη για την προστασία και της ε, μας μα δράση. Αυτό βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται σωστά στην γνωμοδότηση τη Επιτροπή ΔΕΒ δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως προσπάθεια για άσκηση ανθρωπιστικής δράσης η υλοποίηση της αρχής R2P. Θα πρέπει να είναι σαφής η διέξη ε, εντολών μεταξύ ανθρωπιστικών οργανώσεων και επίσης να υπάρχει σαφής πολιτική λογοδοσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πρέπει οι εργαζόμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις να μπορούν να εργάζονται αμερόληπτα βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των όσων αυτό προβλέπει και να μην διακυβεύεται η πραγματική προσφορά, η ανθρωπιστική προσφορά σε αυτούς που τη χρειάζονται, καθώς και η πρόσβαση του ανθρωπιστικού προσωπικού στις ε, υπηρεσίες που χρειάζονται. Είσαι για, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν θα χρησιμοποιήσω και τα τρία λεπτά. Νομίζω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή που διευκρίνησε τα σημεία αυτά και με την ευκαιρία θέλω να αναφέρω μια χωριστή ψηφοφορία που θα ήθελα να συμπεριληφθεί στην ε, ψηφοφορία της Πέμπτης, αύριο δηλαδή. Αφορά την τροπολογία 133. Εδώ μιλάμε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Εθνή. Το τελευταίο κομμάτι αναφέρεται το να αντιμετωπιστεί το θέμα της ενιαίας έδρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ξέρω ότι κάποιες ομάδες ή κάποια μέλη το θεωρούν δύσκολο. Γι' αυτό ζητώ ε, χωριστή ψηφοφορία για αυτό το μέρος σε σχέση με την υπόλοιπη τροπολογία η οποία δεν είναι τόσο δύσκολη για τους υπολείπους από εμά. Ε, το λέω γιατί ξέρω ότι θα βοηθήσει ότι αν είχε μία έδρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβουλίο Ασφαλείας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλω όλα τα υπόλοιπα να εξαρτηθούν από την απόφαση για αυτό το κομμάτι. Και επί των άλλων θεμάτων ε, ε, θα γίνουν κάποιες ε, ψηφοφορίες για τα θέματα που ήδη ανέφερα και να υπογραμμίσω αυτό που είπε η κυρία Νέντσκινη, το πρώτο βήμα σε μια συνολική πορεία και έτσι πρέπει να το εκλάβεται. Ε, δηλαδή πρέπει τα θεσμικά όργανα να καταφέρουμε να δουλέψουν επ' αυτού, να δραστηριοποιηθούν και να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση και την εφαρμογή της ευθύνης για προστασίας σε εποχές που φοβόμαστε ότι επιστρέφουμε και πάλι σε παλιές ιδέες για το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται να έρθει ο Επίτροπος κ. Φούλε και σας υπενθυμίζω, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο ακριβώς στις 9 το πρωί.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 Συνάδελφοι, θα έχουμε την ε, ομιλία του κυρίου Φίλε της ε, έκθεσης προ... και παροπτυσίας της έκθεσης πρόοδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε, που ήρθατε μετά την έγκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της εκθέσεις πρόοδου για τις γειτονικέ χώρες. Είναι σημαντική η έκθεση αυτή για την πολιτική μας, την ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και την ειρήνη ε, και πρόσφατα έχουν εκφραστεί ανησυχίε για τις πολιτικές εξελίξεις ιδίως προς Ανατολάς ε, κύριε Φίλε. Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας ε, πρέπει να καταμετρηθεί έναντι των εξελίξεων αυτών. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τη μόχλεψή μας και να προωθήσουμε τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να αποτιμήσουμε το κατά πόσο είναι εύστοχη η πολιτική μας και πόσο επιτυγχάνεται πρόοδο ω προ την επιδίωξη των στόχων που έχουμε από κοινού προσδιορίσει. Ιδιαιτέρω, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μα, στη λογική της περισσότερης Ευρώπης και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών μας για εξωτερικής, για δημοσιονομικά εργαλεία εξωτερικής δράσης, θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά εντελεχώς. Επίτροπε, σας δίνω το λόγο. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας την Επιτροπή σας. Να πω ευθύ εξ αρχή ότι είναι όχι μόνο χαρά μου, αλλά ότι το γεγονό ότι συνεχίζονται οι συζητήσει για την πολιτική γειτονία. Και ότι τέτοια ζητήματα τα εξετάζω όχι μόνο όταν έρχομαι να μιλήσω στο κοινοβούλιο, αλλά σε καθημερινή βάση. Να ξέρετε ότι κάνω ό,τι μπορώ, όσο πιο συχνά μπορώ και Μαζί σας επίσης συζητώ ε, όσο πιο συχνά γίνεται. Κύριε Πρόεδρε λοιπόν, ε, κύριοι βουλευτές, ε, χαίρομαι που έρχομαι απευθείας από τη συνάντηση της Επιτροπής που μόλις ολοκληρώθηκε στη δική σας συνεδρίαση. Ολοκληρώσαμε την εξέταση του συνόλου των εκθέσεων για την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεκινήσω αμέσως με τα συμπεράσματα τα οποία διεξήγαμε από τις εκθέσεις αυτές. Πρώτον, ακόμη βρισκόμαστε μόνο στην αρχή της όλης διαδικασίας. Είναι σαφές ότι η μετάβαση προς την δημοκρατία και η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας με μεταβατικές περιόδους θα πάρει καιρό. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει στην Αίγυπτο, την Τινησία, τη Λιβύη, όλα αυτά δείχνουν ότι ο δρόμος προς τον εκδημοκρατισμό δεν είναι ένας δρόμος ομαλός ούτε και σύντομος. Έπειτα, οι εκθέσεις μας δείχνουν ότι οι εκλογές είναι σημαντικό, αλλά παρόλα αυτά ένα πρώτο δηλοβήμα προς τον εκδημοκρατισμό. Πρέπει εδώ να διασφαλίσουμε το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών, ε, την, την ελευθερία του συνασπίζεστε και του ε, διαδηλώνει και την ελευθερία ε, έκφρασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης την ισότητα των γυναικών έναντι του νόμου και της κοινωνίας, καθώς και την ε, ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών. Κάτι που είναι ακόμα πρόβλημα σε πολλές χώρες, όπως και διαφθορά. Τρίτον, οι κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα, δώσουν, θα πάρουν ακόμη περισσότερο καιρό μέχρι να δώσουν απτά αποτελέσματα. Η έλλειψη αποτελεσμάτων όμως αυτή καθεαυτή απειλεί να υπονομεύσει ή να επιβραδύνει τη διαδικασία και δημοκρατισμού. Οι γείτονε μα και οι πολίτε και οι πολίτες των χωρών αυτών ε, περιμένουν τη δημοκρατία, αλλά χρειάζονται και δουλειέ. Μην ξεχνάμε ότι η Αραβική Άνοιξη αυτή η ίδια πυροδοτήθηκε από τις οικονομικές δυσκολίες και τις πολιτικές ελλείψεις. Τέταρτον, παρά τι ε, δυσκολίε, θα πρέπει να παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει στην πολιτική γειτονία μα. Πολλοί γειτονέ μα θέλουν να μα προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω λοιπόν η ειρήνη και η ευημερία στι περιοχέ αυτέ. Ενώ είμαι βέβαιο ότι το πολιτικό μας πλαίσιο είναι σωστό, θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του πλαισίου αυτού και την ενημέρωση των πληθυσμών των χωρών αυτών, ώστε να καταλάβουν ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί να τους προσφέρει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριοι Βουλευτές, οι προκλήσει είναι ακόμη σημαντικέ. Όμω και κάποιοι από του εταίρου μα έχουν ε, ε, καταβάλει προσπάθειες και έχουν επιτύχει αποτελέσματα στην ε, επιδίωξη των στόχων που είχαμε θέσει. Θα πρέπει να αλλάξει ο ρυθμός και κατεύθυνση κάποιων από τι μεταρρυθμίσεις κάνοντα εδώ διάκριση μεταξύ των διαφόρων εταίρων μας διαφοροποίηση μάλλον, ε, εφαρμόζοντα την αρχή more for more, περισσότερα για περισσότερα αποτελέσματα. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείξουν την ίδια διάθεση να μεταρρυθμίσουν, όπως αυτοί που ζητάτε από εκείνους Και εδώ θα πρέπει να διανοματίσει ένα ενεργό ρόλο και η κοινωνία των πολιτών. Είναι καθοριστικής σημασίας η μεταρρύθμιση αυτή για την πολιτική γειτονίας και θα συνεχίσει να είναι. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα κοινοβούλια των χωρών αυτών και άλλους σημαντικούς φορείς, όπως κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους του κόσμου των επιχειρήσεων. Με χαρά μου έμαθα ότι σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου η πολίτες από την περιοχή της πολιτικής γειτονίας και από την Ανατολική, από τον Νότο, σημειώνουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αλληλεγγύη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι καρπός και της διαρκούς και αμύωτης προσπάθειάς μας. Θέλουμε εδώ να έχουμε μεταρρυθμίσεις βάσει των στόχων που έχουμε συζητήσει με τις χώρες αυτές, καλύπτοντας τις ανησυχίες των πολιτών, ε, της κοινωνίας των πολιτών των χωρών αυτών και τις προσδοκίες τους. Αυτό είναι σημαντικό και για το Ευρωκοινοβούλιο και ε, εδώ είναι σημαντική η στάση του δικού μας κοινοβουλίου, στη Γεωργία, λόγω χάρη. Είδαμε ότι από την περασμένο Οκτώβριο και την αλλαγή εξουσίας υπήρξε μία έντονη συγκατοίκηση στην εξουσία. Όμως ε, ήταν επικοδομητικός ο διάλογος πλειοψηφίας και μεμψηφίας στο κοινοβούλιο της χώρας και έγιναν σημαντικά πρακτικά βήματα για να κατευναστούν οι εντάσεις ε, του διαστήματος μετά τις εκλογές στη χώρα αυτή. Αυτό πραγματικά είναι μια τάση που θα πρέπει να την αθαρρύνουμε. Το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο για την Δημοκρατία που δημιουργήθηκε πέρσι επίσης μπορεί να διαρματίσει σημαντικό ρόλο στηρίζοντας τις ε, δυνάμεις ειρήνευσης που εργάζονται υπέρ των δημοκρατικών αλλαγών και στηρίζοντας τους φορείς που φέρνουν τις πραγματικές αλλαγές στην γειτονιά της Ευρώπης αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια και προσφέροντας πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, να στραφώ τώρα στι ενεξελίξει διαπραγματεύσει μα για συμφωνίε προσχώρηση και στην συνολική, στην, σφαιρική, στην ευρύτερη περιοχή ελεύθερων ε, συναλλαγών. Έχουμε προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις με την ε, Γεωργία και την Αρμενία. Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν. και ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις και ε, συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία. Προτού υπογραφούν όμως οι συμφωνίες αυτές, θα πρέπει να υπάρχει αποφασιστική δράση και απτά αποτελέσματα στις προτεραιότητες μεταρρύθμισης, αλλά και στην αντιμετώπιση αναγκών και των ανεπαρκειών της δικαιοσύνης και των εκλογικών διαδικασιών. Ελπίζουμε ότι η σύνοδος της ε, ανατολικής ε, ζώνης στο Βίλνιους θα επιτρέψει να έχουμε στενότερη συνεργασία με τους ε, εταίρους μας εξανατολών και με σκοπούς πολιτικούς και οικονομικούς. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρύτερη περιοχή ελεύθερων συναλλαγών με το Μαρόκο και την ε, ενεργό του συμμετοχή. Επίσης, διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει με την Τινησία και στο εγγύς μέλλον θα συνεχίσει η προετοιμασία και η συνομιλίες με την Ιορδανία. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε την κινητικότητα των πολιτών. Υπάρχουν χώρες όπως η Μολδαβία που έχει προχωρήσει σε απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων πέρασε στη δεύτερη φάση και έχουμε συζητήσει την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και με τη Γεωργία. Οι διαπραγματεύσεις κινητικότητας και απελευθέρωσης έχουν, προχωρήσει, έχουν ολοκληρωθεί με το Μαρόκο και έχουν προχωρήσει με την Τινησία. Επίση, η μετανάστευση και η κινητικότητα είναι κάτι που μα απασχόλησε στις συζητήσεις μας με την Ιορδανία. Μα απασχολούν κινήσεις ερευνητών, φοιτητών, νέων και καθηγητών με προγράμματα όπως το Tempus, το Erasmus Mundus και το Youth in Action, νεολαία σε δράση. Η πρόοδος στα προγράμματα αυτά, τα ζητήματα που πολλές φορές είναι ευαίσθητα, είναι καθοριστική σημασίας. Όχι μόνο γιατί έτσι θα, θα καλύψουμε μια από τις βασικές προσδοκίες των γειτόνων μας, αλλά γιατί η κινητικότητα των πολιτών πάει χέρι-χέρι με την μετακίνηση και την κυκλοφορία ιδεών και κοινών αξιών. Θέλω να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή την ε, πτυχή της συνεργασίας μας στο προσεχέ μέλλον. ω προ την οικονομική συνεργασία και την στήριξη των μεταρρυθμίσεων στις γειτονικέ χώρες. Αξιοποιούμε όλο το φάσμα των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μα με προγράμματα όπως το Spring και το EPIC με κονδύλια που έχουν αποδοθεί σε όσους κατώτερες προσπάθειες για τον εκδημοκρατισμό και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δεύτερη φάση της διευκόλυνσης και την κοινωνία των πολιτών εγκρίθηκε με τον νέο προπολογισμό για 45 εκατομμύρια για το 2013 θα έχετε προσέξει ότι φέτος ε, το σύνολο των εκθέσεων δημοσιεύτηκαν και εγκρίθηκαν δύο μήνες νωρίτερα από ό,τι έγινε πέρσι. Αυτό μας επιτρέπει να αποτιμήσουμε τις εκθέσεις πρόοδου καλύτερα και λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο προγραμματισμό μας για την οικονομική ε, στήριξη των ε, γειτόνων μας βάσει της αρχής περισσότερες προσπάθειες για περισσότερα αποτελέσματα. More for more. Έχουμε ε, τονώσει την συνεργασία μας και με τις χώρες και των, της Ανατολής και του Νότου. Ιδίω προ τον Νότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιήθηκε για να δώσει μια, ένα προσανατολισμό στι χώρε αυτέ. Αναλάβαμε τη συμπροεδρία της Ένωσης, ε, της Ευρωμεσογειακής Ένωσης και προκειμένου να τονώσουμε την περιφερειακή συνεργασία στην Βόρεια Αφρική, στο Μαγκρέμ, με χειροπιαστές προτάσεις από την ανακοίνωσή μας ήδη του προηγούμενου Δεκεμβρίου και στις συναντήσεις του 5 συν 5. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια σφαιρική ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να ε, συμβαδίζει με ε, συστηματική δράση όλων των ευρωπαίων φορέων, των ευρωπαϊκών φορέων. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα, και τα δικά τους θεσμικά όργανα. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές από την πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η πολιτική αυτή, η πολιτική της γειτονίας είναι πλέον κατάλληλη και πλέον ευέλικτη ώστε να στηρίξουμε τους ε, γείτονές μας ε, και τις προσπαθίες τους τα ερχόμενα χρόνια. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, η διόγκωση της ανεργίας παραμένουν και ολοένα και επιδεινώνονται. Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ε, προβλημάτων, οι κοινωνικοί δείκτες που συνεχώς ε, είναι, μας απογοητεύουν δείχνουν πόσο χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και πόσο αναγκαίες είναι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Οι χώρες μας στα ανατολικά χρειάζονται ακόμα τη στήριξή μας για να πετύχουν τους στόχους τους. Είναι πεποίθησή μας ότι αξίζουν ένα μέλλον γεμάτο ελπίδες μιλώ για ένα από τα πλέον ισχυρά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξωτερικής της πολιτικής εδώ έκφραση της δυνατότητάς της να μεταβάλει τα πράγματα, την προοπτική μιας χώρας να προσχωρήσει βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μια χώρα συμμερίζεται τις αρχές ελευθερίας, δημοκρατίας και σεβασμού του κρατούς δικαίου, μπορεί να προσχωρήσει. Προς τον Νότο, προτείνουμε στη διευρυμένη ευρωπαϊκή ζώνη ε, την δυνατότητα ένταξης αναλόγως, μάλλον προκειμένου οι εταίροι μας να επωφεληθούν από, ε, ε, από την ένταξή τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δεχτούν τις αρχές και τις αξίες μας, αυτές που διέπουν την ενιαία αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο ελπίζουμε ότι η μετάβραση προς τη δημοκρατία θα συνεχίσει και στις χώρες του Νότου. Έτσι λοιπόν θα σας ευχαριστήσω για τον ενεργό σας ρόλο στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Διότι ο εκδημοκρατισμός δεν είναι απλή υπόθεση. Και τα κοινοβούλια και οι πολίτες των χωρών αυτών θα πρέπει να είναι κινητήριες δυνάμεις των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εν είδη συμπεράσματο, επιτρέψτε να τονίσω ότι οι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την κάθε μια από τι χώρε με τι οποίε υπάρχει συνεργασία είναι μοναδική. Πρέπει να διαφοροποιούμε βεβαίω τι πολιτικέ μα αποκρίσει ανάλογα με τι εξελίξει, τι φιλοδοξίε και τι ανάγκε του καθενό από του εταίρου μα αλλά η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία μας δίνει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των εταίρων και στο τι αυτοί περιμένουν από τι σχέσει που συνάπτουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα και στην αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει αμύωτε τις δεσμεύσει που έχει αναλάβει στα πλαίσια τη πολιτική Γειτονία. Έτσι λοιπόν περιμένω και από εσά την στήριξη, την έμπνευση και την όθηση που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε στις κοινέ μας προσπάθειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, για την ε, συζήτησή μας στους συντονιστές ή τους ε, αντικαταστάτες τους θα δώσω δύο λεπτά. Στους υπολείπους, ένα λεπτό. Δυστυχώς έχουμε πίεση χρόνου και θέλουμε να προλάβει ο Επίτροπος να απαντήσει. Πρώτος ο κύριος Αλαφράνκα. ΕΛΚ, δύο λεπτά. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε τόσο γρήγορα. Πρέπει να σας πω ότι φτάσατε ταυτόχρονα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περίπου και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και πραγματικά αυτή η δράση σας είναι υπόδειγμα καλής συνεργασίας με το Κοινοβούλιο. Στέκομαι στο τελευταίο που είπατε, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα και στις νέες συνθήκες μετά την τελευταία αναθεώρηση που έγινε πριν από μία διετία, ε, οφείλει να αποτελεί ένα μέσο που να προσαρμόζεται στις συνθήκες και στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας που είναι εταίροι μας. Όπως είπατε πολύ καλά, ε, είναι σημαντική οι πόροι που αφιερώνονται και σε χαλεπούς καιρούς οικονομικά και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με νέα μέσα όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Είναι σημαντικό και το είπατε και εσείς στην εισήγησή σας να έχουμε πιο στενές σχέσεις και καλύτερες με την κοινωνία των πολιτών και ένα δόγμα για να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε αυτή τη πολιτική. Το more for more που είχατε, περισσότερες προσπάθειες για περισσότερα αποτελέσματα. Δύο διαστάσεις έχει η πολιτική γειτονίας. Τη βόρεια διάσταση που θα ήθελα να ρωτήσω. Τι γίνεται με την Ουκρανία Πώς προχωρεί η δικαιοσύνη, ο ποινικό κώδικας και η μεταρρύθμιση του για να αποφευθούν καταστάσεις τύπου Ιούλιας Τιμοσέγκο ε, και άλλα ε, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία, Πρόεδρε, μας ανησυχούν τα επεισόδια που έχουν γίνει ε, οι δυσκολίες της συγκατοίκησης τα αντίπεινα που έχουν υποστεί ορισμένα μέλη του κόμματος του Προέδρου, καθώς επίσης και εφαρμογή κριτηρίων επιλεκτικής δικαιοσύνης. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε. Σε ό,τι αφορά τώρα την νότια διάσταση, μιλήσατε κύριε Πρόεδρε για μια συμφωνία που λανσάρατε με το Μαρόκο, την Τινησία και την Ιορδανία. Και τελειώνω Πρόεδρε για την Αίγυπτο. Το συνταγματικό δικαστήριο έχει διακόψει την εφαρμογή του εκλογικού νόμου. Ε, εσείς πώς αξιολογείτε όλα αυτά στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας Το Το Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Νέιτς. I'm sorry. Uh, President Commission. Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ που ξεκινήσατε, μια συχνή επικοινωνία μαζί μας, όπως προανέφεραν και άλλοι. Εκτιμάμε ιδιαίτερα το γεγονός. Η έκθεση αυτή προόδου, κύριε Επίτροπε, φτάνει σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup οι οποίες κατόπιν άλλαξαν, δεν έχουν ακριβώς ενισχύσει την ε, αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. Οπότε αυτό ε, δεν διευκολύνει τη σχέση μας με τις χώρες της ε, νότιας ακτής της Μεσογείου. Ε, γνωρίζετε ας πούμε για την περίπτωση του Μαρόκου ότι εγώ είμαι μέλος της ομάδας φιλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου όπως είπα και στους μαροκινούς μου φίλους, δεν υπάρχει σωστή φιλία αν δεν είναι δυνατή οι δυνατές επικρίσεις. Έτσι λυπούμαστε για τις ε, αποφάσεις των μαροκινών αρχών πριν από λίγες εβδομάδες να εμποδίσουν την πρόσβαση σε κάποιους συναδέλφους, παρότι δεν συμφωνώ με τις θέσεις των τεσσάρων αυτών συναδέλφων, ε, αλλά θα πρέπει ε, να πω ότι οι Μαροκινοί έχασαν μια ευκαιρία να παρουσιάσουν το θέμα και ε, αντίθετα ε, δεν προσπάθησαν να ε, αποδείξουν την εγκυρότητα των δικών τους ισχυρισμών. Παρά τα αυτά, αυτό δείχνει τις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν όταν ξεκινάμε μία σε βάθος και ολοκληρωμένη σχέση. Δεν εννοώ καθόλου ότι θα πρέπει να ανασταλούν οι συνομιλίες ή οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά αυτό πρέπει να περιμένουμε όταν ξεκινάμε ε, στενές και ολοκληρωμένες σχέσεις. on behalf of the Socialist Group. Εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Ξέρετε κύριε Επίτροπε ότι η Επιτροπή μας έχει επανειλημμένως εκφραστεί για το ρόλο και την πολιτική δράση που, και το, το πολιτικό αποτέλεσμα που δίνει η όλη αυτή ε, προσπάθεια και η παρουσία σας σήμερα εδώ το αποδεικνύει μια νέα πολιτική γειτονία. Δεν μπορεί βέβαια να λύσει σε συντομότατο χρονικό διάστημα όλα τα προβλήματα, ούτε και το περιμένει κανεί αυτό. Ωστόσο, πιστεύω ότι το να, να ελέγχουμε από καιρού καιρό την πολιτική αυτή είναι σημαντικό και για τι ενεξελίξει μετατροπές, αλλά και για να προσπαθήσουμε να τι δώσουμε μια νέα πνοή ε, όταν χρειάζεται. Να τονίσω απλώς ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντούμε σε αυτή τη διαδικασία έχουν να κάνουν με ένα πρώτο θέμα ότι οι πολιτικές γειτονία δεν, είναι, δεν θα πρέπει να είναι ένα δευτερογενές, ένα παραπροϊόν της εξωτερικής πολιτικής. Θα έπρεπε να είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής. Αν θέλουμε πρωταγωνιστικό πολιτικό ρόλο στις διαφορετικές περιοχές που μας ενδιαφέρουν, θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική αυτή. Εάν λοιπόν η εξωτερική μα πολιτική θέλουμε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλε αυτέ τι περιοχέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει εκεί και την πολιτική γειτονία, γιατί χωρί τη μια ή άλλη δεν μπορεί να προχωρήσει. Το δεύτερο στοιχείο που δημιουργεί δυσχέρειε είναι ότι σήμερα αυτό που κουράζει και δεν αυτό μάλλον που δεν προχωρά εύκολα είναι η κοινοβουλευτική διάσταση στα πλαίσια της πολιτικής γειτονία. Σκέφτομαι τις διάφορες νομοθετικές λύσεις που θα πρέπει να εξευρεθούν σε όλα αυτά τα κοινοβούλια που αναφέρατε κι εσείς. Δεν φαίνεται να υπάρχει σταθερή παρακολούθηση της κοινοβουλευτικής αυτής διαδικασίας διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν των συγκεκριμένων προβλημάτων που εντόπισε θα πρέπει διαρκώς να παρακολουθεί τις κοινοβουλευτικές εξέλιξεις στις χώρες αυτές και να προσφέρει στήριξη. Και μια τρίτη παρατήρηση και ολοκληρώνω. Τι συσχετισμό βλέπετε να υπάρχει μεταξύ ε, της πολιτικής γειτονίας πέραν του 5 συν και της ε, επικαιροποίησης της διαδικασίας υπομοκρατασμού. Η θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να διευκολυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Κυρία Λούνατσεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Φίλε. Εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την προθυμία που έχετε κάθε φορά που ε, βγαίνει μια έκθεση από εσά να έρθετε να εγκαίρως να τη συζητήσετε μαζί μου. Θα αναφερθώ για λίγο στον Νότιο Κάφκασο και μετά η συνάδελφος Σούλτς θα ασχοληθεί με την Ανατολή. Βεβαίως συμφωνώ μαζί σας με αυτό που λέτε, ότι χρειαζόμαστε και τα δύο. Και την δημοκρατία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και για όλες αυτές τις χώρες είναι δύσκολο για διαφορετικούς λόγους. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω που αναφερθήκατε στην κατάσταση του θέση των γυναικών. Σε όλες αυτές τις χώρες σηκώνει βελτίωση από βία εναντίον των γυναικών από τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή κτλ. Θα ήθελα να σχολιάσω σε δύο συγκεκριμένες χώρες. Κοίταξα τις περιλήψεις των ε, εκθέσεών σας, η Γεωργία πρώτον, όπου Πρόσφατα έγινε η κοινοβουλευτική συνάντηση με τους Γεωργιανούς. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε ψήφισμα. Αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, η δυσκολία της συγκατοίκησης εμφανίζεται και στην έκθεση την οποία θεωρώ σωστή και ισόρροπη. Οι δυσκολίες που υπήρχαν από το παρελθόν και άλλες που υπάρχουν τώρα. Αυτά είναι σωστό που πρέπει να τα λέμε για να φροντίζουμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Όσον αφορά το Αζερμπαϊτζάν τώρα, εκεί θεωρώ ότι, αν δεν κάνω λάθος, σας στείλαμε ε, μια επιστολή, η συνάδελφος Βεναζούλς και εγώ, ε, ε, στον πρόεδρο του Αζερμπατζάν, γιατί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλο και περισσότερο επιδεινώνεται. Ε, υπάρχουν καταστάσεις όπου όχι μόνο, λέτε στην εκθεσή σας, έχουν μπει στη φυλακή πολιτική της αντιπολίτευσης, αλλά και άνθρωποι που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και οι οποίοι ε, εκπαίδευαν πολίτες για την παρακολούθηση των εκλογών και συνελήφθησαν την ώρα που έκαναν αυτή την εκπαίδευση προσώπους ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έχουμε νομοθεσία που, ε, που περιορίζει τον έλεγχο, μάλλον αυξάνει τον έλεγχο για τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στην περίληψή σας θέτετε όλα αυτά τα θέματα, αλλά επ' αυτού πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι και επικριτικοί. Το ξέρω ότι το κάνετε κι εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να διαβιβαστεί πιο αποτελεσματικά αυτή η κριτική, γιατί όπως ξέρετε το Ζερμπατζάν δεν χρειάζεται τα χρήματα της Ευρώπης, έχουν πολλά, πολύ αέριο και πετρέλαιο, ε, από το οποίο εξαρτώμαστε είμαστε κι εμείς. Έτσι η προθυμία τους να προχωρήσουν ε, ε, στις μεταρρυθμίσεις η ελευθερία του συνέρχεται και μια σειρά από πολύ βασικά πράγματα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Ε, με τη δική μας βοήθεια πώς πιστεύετε ότι μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα εκεί. Mr. Kabrnoch. Κύριος Καμπερνόχ. Děkuji, vážený pane předsedo, pane komisaři. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να απευθυνθώ σε εσά ε, στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής της Επιτροπής, στην οποία δεν είμαι μέλος. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να ε, περιγράψω ε, την ε, διαφορά ανάμεσα σε μέλη της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Είμαι πρόεδρος αντιπροσωπείας για το Αζερβαϊτζάν και τη Γεωργία και την Αρμενία. Και θέλω να επισημάνω εδώ ότι κατά την άποψή μου πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ τις σχέσεις μας με το Κοινοβούλιο της Γεωργίας. Είχαμε ήδη πολλές προειδοποιητικές ενδείξεις που δείχνουν μια πόλωση ανάμεσα στο νέο κυβερνητικό συνασπισμό και τα πρώην κυβερνητικό κόμμα που τώρα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Είχαμε πολλά ανησυχητικά ε, σήματα πρέπει με την ευκαιρία αυτή να βοηθήσουμε την καλύτερη επικοινωνία, την ε, συγκατοίκηση, τη συνύπαρξη μεταξύ της αντιπολίτευσης και του συνασπισμού της Γεωργίας, να ε, εμποδίσουμε τη Γεωργία να απομακρυνθεί έτσι περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε Ιταλικά κύριε Πίτροπε. Ε, Ήθελα κι εγώ να ρωτήσω στην έκθεσή σας τι ε, γίνεται με τον Ραγκόρνο Καραμπάχ. Οι εντάσεις συνεχώς ε, ξύνονται και υπάρχουν συγκρούσεις. Αυτό δεν έχει επιπτώσει στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Διότι δημιουργεί μια διαρκώς αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, κάτι που είναι τελείως ασύμβατο με τη διαδικασία της εταιρικής σχέσης που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτή η εδαφική αναμέτρηση που έχει να κάνει με παραβίαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Μάνου Μιλιτάρη κιόλα, είναι κάτι που πρέπει να επιληθεί κάποια στιγμή. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ μπορεί να είναι καθοριστικός για την προοπτική αυτή ειρήνης στο μέλλον. Ο κύριος Λίζα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα μιλήσω για τη γεωργία, για αλλαγή. Παρόλο που γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Πίτρο, ποια είναι ε, η θεώρησή μου για τη γεωργία. Είμαι πιο αισιόδοξο από εσά. Θα ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας ένα γενικότερο σχόλιο. Όπου και να κοιτάξει κανείς, σε οποιαδήποτε χώρα της ανατολικής γειτονίας, υπάρχουν προβλήματα. Παντού. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως κατά τύχη δεν τους δίνουμε μια πραγματική προοπτική. Τι τους προσφέρουμε, γιατί προβληματίζονται, δεν ξέρουν τι προθέσεις έχουμε. Ε, μιλούμε για την ε, Σύνοδο Κορυφής για την Ανατολική Γειτονία στο Βίλνιους. Θα είναι καλή ευκαιρία να διατυπώσουμε στόχους. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία είναι ένα νέο μέσων, βεβαίως πολύτιμο, πλην ε, νεοσύστατο και δεν είναι ισχυρό εργαλείο και δεν έχει και μεγάλη πρικοδότηση. Για ε, αυτό που, λοιπόν χρειάζεται πολιτική βούληση για να χρηματοδοτηθεί αυτό το ταμείο από τα κράτη-μέλη. Σίβιτς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξής κύριε Επίτροπε. Αυτή η σύνοδο κορυφή στο Βίλνιου θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να πούμε την αλήθεια, όλη την αλήθεια όμως, ε, στου εταίρου μα, αλλά να την ομολογήσουμε και στον εαυτό μα για την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Οι καλέ ειδήσει ποιε είναι. Σε κάποιου τομεί έχουμε πρόοδο, κινητικότητα, η πολιτική θεωρήσεων διαβατήριων. Τρει συνθήκε έχουμε επιτάπητο, ε, συμφωνίε και οι τρει κινδυνεύουν. Η κατάσταση λοιπόν είναι περίπλοκη και το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Ένα άλλο σημαντικό ε, είναι ο κανόνας περισσότερες προσπάθειες για περισσότερα αποτελέσματα, αυτό το more for more. Αυτό ήρθε εκ των υστέρων. Ε, έχουμε κάποιους δείκτες για τη συγκριτική αξιολόγηση και να μπορέσουμε να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα και έναν απολογισμό. Τι έχει γίνει και τι απομένει ακόμα να γίνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τη συντομία. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου αφορά τη Συρία και την Ιορδανία. Αναφέρεται το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία ως νέο μέσον Υπάρχει όμω και το ίδρυμα, το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ρωτώ, υπάρχουν επίκαιρα μέτρα σημερινά για τη Συρία ε, που να βοηθά χωρίς γραφειοκρατία ε, δικηγόρου, ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ε, την ειρηνική αντιπολίτευση. Ή έχουμε μάλλον την πιο ανθρωπιστική προσέγγιση με γιατρού. Το δεύτερο για την Ιορδανία. Εκεί χρηματοδοτούμε καταβλισμού προσφύγων. Τα δύο τρίτα των προσφύγων όμω δεν ζουν στου αλλά στην Αποτέλεσμα, η Ορδανική κυβέρνηση πρέπει να δίνει πολύ περισσότερα χρήματα. Περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται αυτή η συνεισφορά για φέτο. Και ρωτώ, δεν θα μπορούσαμε κι εμεί με άλλου δωρητέ να βοηθήσουμε με δημοσιονομική βοήθεια επιπλέον τη χώρα αυτή, γιατί κινδυνεύει να καταρρεύσει. Γιατί Ουκρανία δεν έχω ε, ερώτηση. Ακόμα προσπαθώ να αποδικοποιήσω την απάντηση που μας δώσατε στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ απολύτως ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και η πρέπει να βρίσκονται στο προσκήνιο. Οι ερωτήσεις μου αφορούν την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική. Είπατε ότι ένα, μόνο, ένα και μόνο βήμα αποτελεί η σταγματική διαδικασία. Όμως σε χώρες όπως η Αίγυπτος και λοιπά ε, που ε, μπλέκονται μόνο οι άνδρες ενώ τα θέματα των γυναικών δεν τίθεται στην ημερήσια διάταξη τι είναι αυτό. Φοβάμαι ότι κλείνει το παράθυρο, η ευκαιρία που έχουμε πάει να εξαφανιστεί. Πρόκειται για μια αρχή η οποία φοβάμαι ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες αργότερα. Οπότε ρωτάω, αυτές οι γυναίκες που αντιτίθενται σε δικτάτορες και που τώρα διαπιστώνουν ότι τα δικαίωματα που είχαν υπό τις δικτατορίες αυτές εξαφανίζονται, τι μπορούμε να κάνουμε. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την οικονομική υποστήριξη. Πότε όταν βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κοινωνία των πολιτών υπάρχουν κανόνες για τις οργανώσεις που πρέπει να, υπάρχουν, να προϋπάρχουν οι οργανώσεις για κάποια χρόνια. Σε χώρες όπως η Λιβύη δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, δεν υπήρχαν ούτε καν οργανώσεις γυναικών. Πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή την υποστήριξη που είναι απολύτως απαραίτητη αυτή την εποχή. Τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σούλτς. Ich kann mich ναι. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία ε, και την ταχεία έλευσή σας εδώ. Πραγματικά δείξατε μεγάλη δέσμευση και δημιουργικότητα για να φέρετε πιο κοντά τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι είναι απογοητευτικές όσο και οπισθοδρομικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα στην Ουκρανία η επιλεκτική πολιτική δικαιοσύνη πέρα από τις ε, ε, Λουσέγκο και Τιμοσέγκο περιπτώσει. Τι γίνεται με τον Δημήτρη Κόσμαν και την υπόθεση Λασέγκο που είναι και άλλοι ε, κρατούμενοι. Συχνά μας κατηγορεί η Ουκρανία για ζητήματα ε, ενεργειακά και ότι δεν ασχολείται πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαπραγμάτευση της τιμής του αερίου με τη Ρωσία ή ότι την παρακάπτουμε την Ουκρανία με το South Stream η Λευκορωσία είναι ακόμα μέλος ανατολικής γειτονίας, αλλά δεν έχουμε επίσημες ακόμα πολιτικές επαφές. Τι κάνετε για να ξαναφέρετε πίσω ε, στο ευρωπαϊκό καράβι τη Λευκορωσία και τι γίνεται με τους πολιτικούς κρατούμενους, με την επικοινωνία μας μαζί τους. Ευχαριστώ. Κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο για την ε, δελεχή πληροφόρηση που μας έδωσε για την πολιτική γειτονία. Ήθελα να ρωτήσω κύριε Επίτροπε ε, πώς γίνεται ο συντονισμός με την πολιτική που ασκείται από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δηλαδή με τη δραστηριότητα της, ε, της της εκπροσώπου. Ε, επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα ή έχει βρεθεί ένας διάβλος μια καλή λειτουργικότητα μεταξύ των δύο τομέων που αποφέρει ωφέλη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε κυρία Αντρικένε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, μόλις ολοκληρώσαμε μια συνεδρίαση, την συνάντηση μάλλον της Μικτής Κοινοβουλευτικής ε, Συνέλευσης της Euronest. Και υπάρχουν εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Μολδαβίας που περιμένουν να ακούσουν ε, και τα δικά σας, τις δικές σας παρατηρήσεις και το τι πρόοδο έχουμε επιτύχει. Η πολιτική γειτονία είναι ένα καλό εργαλείο, αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς ταγκό, όπως λένε. Και θέλουμε να χορέψουμε με τις χώρες του Νότου, τους γείτονες ε, του Νότου, και αυτό είναι ο λόγος που το λέω, αλλά πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο και προς Ανατολάς. Η δική μου επιθυμία και βούληση είναι να υπογραφεί συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά είχε συμφωνίες με την Μολδαβία, είχε μονογράψει τις συμφωνίες με τη Μολδαβία, την ε, ο κύριος Μιλανμόν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε εδώ. Εγώ θα αναφερθώ στη Μεσόγειο και στη νότια γειτονία. Πρώτον, Υπάρχει ανάγκη να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε, να είμαστε παρόντες στην αλλαγή εκεί. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση για την Ευρώπη. Εκείνοι μπορούν να έχουν διαφορετικά μοντέλα. Εμείς θα πρέπει να είμαστε παρόντες, να τους βοηθήσουμε και να τους ενθαρρύνουμε. Και πιστεύω ότι το μήνυμα είναι συνένεση, συνένεση, διάλογο, συνένεση και τίποτα άλλο. Και ε, βλέπετε να υπάρχει καμιά δυνατότητα να υποστηρίξει χθούν οι δυνάμεις κοσμικές, οι μη θεοκρατικές στην Αίγυπτο. Για το Μαρόκο κάνει ε, μεταρρυθμίσεις, δεν ήταν βίαιη η μετατροπή και η μετάβαση, γίνεται μια ήπια, μια ήρεμη μετάβαση, θα τους βοηθήσουμε. Και ένα συγκεκριμένο, τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των, ελευθεριών. Για τα γεωργικά και τα αλλιευτικά προϊόντα έχετε τεθεί σε ισχύ. Βαθιά και συνολική συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο. 5-6 χρόνια όμως έχει αποτελματωθεί η ιστορία για τις υπηρεσίες. Τι γίνεται εκεί παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τέλος ο κύριος ε, Ντόρφερ. Κρέσλιντορφλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε Φίλε. Δεν θέλω να κάνω επιπλέον ερωτήσεις γιατί αλλιώς μέχρι το βράδυ θα μας απαντάτε όλα αυτά που σας ρωτήσαμε. Ε, είναι απολύτως απαραίτητο και επίγον εμείς και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο να τονίσουμε και προς τα έξω και δημόσια για την πολιτική γειτονία και να υποστηρίξουμε και την πολιτική γειτονία. Έχω την αίσθηση ότι το μόνο που μας απασχολεί πλέον η οικονομική κρίση και άλλα τεινά. Αλλά αυτά τα θέματα της γειτονίας δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε να χαλαρώσουν και με ψήφισμα ε, στην Ολομέλεια να τονίσουμε ότι σας υποστηρίζουμε και εσάς και τις απαιτήσει που θέτει σε όλους μας η πολιτική γειτονία και να το πούμε και προς τους γείτονες αυτό. Είναι μάλλον έκκληση αυτή και λιγότερο ερώτηση που σας απευθύνω. Τόσες ερωτήσεις σας έγιναν τώρα κύριε Πίτροπε. Mm-hmm. Απαντήστε. Χρόνο έχετε, μην ανησυχείτε. Till 1 p.m. Μέχρι τη μία εννοώ. Ευχαριστώ. Πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι την τελευταία φορά μου δίνετε. Είναι προσωπικό δώρο. Την περασμένη φορά μου δώσετε πέντε λεπτά λιγότερο. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, διότι δείχνουν πόσο ενδιαφέρεστε για τα θέματα αυτά και είναι βεβαίως και ένας τομέας των ειδικών σας γνώσεων. Φαίνεται πόσο ε, έχετε ενεργό ρόλο στην πρόθεση αυτών των ζητημάτων. Να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο κ. Παντζέρη. Ότι χρειαζόμαστε και κάποιο feedback, κάποια ε, αντίδραση. Θα ήθελα να βλέπω δύο πράγματα να συμβαδίζουν τη διαρκή δέσμευσή μας ως προς τις αρχές αυτές της νέας πολιτικής γειτονίας να πηγαίνει που βασίζεται όπως επεσήμανα στην αρχή του more for more και την ε, επικοινωνία, τη διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών και την οικοδόμηση των δικών τους δυνατοτήτων, ε, μια μακροπρόθεσμη επένδυση και ταυτόχρονα αυτά να πηγαίνουν παράλληλα με στρατηγική ε, με στρατηγικό σχεδιασμό, τον δημιουργία ενός συνόλου εργαλείων. Αυτή είναι η κατάλληλη πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες του ενός ή του άλλου εταίρου. Ταυτόχρονα, πραγματικά και εγώ αδειμονώ να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός για να γνωστοποιούνται οι αντιδράσεις και για να υπάρχουν διαρκείς διαπραγματεύσεις και συνομιλίες Άτυπε και επίσημέ και μαζί σας, αλλά και με τους εκπροσώπους των ε, συνεργατών, των τέρων μας. Πέρυσι μόλι, πολύ πρόσφατα, συμφωνήσαμε με τους εκπροσώπους γειτονικών χωρών ότι τουλάχιστον εξαμηνιαίως θα συναντώμαστε με τους ανώτερους αξιωματούχους για να συζητούμε τα σημαντικότερα ζητήματα της πολιτικής γειτονίας, ώστε και εμείς να μαθαίνουμε το τι συμβαίνει στις χώρες αυτές, αλλά ακόμη περισσότερο το πώς οι εταίροι μας αντιλαμβάνονται την ε, επιρροή και τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Να ξέρουμε από εκείνους τους ίδιους, από πρώτο χέρι, κατά πόσον δίνει αποτελέσματα η πολιτική μας. Δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο διάλογο μόνο με του ανώτερου αξιωματούχου, αλλά και με εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και με εκπροσώπου των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Πρώτη παρατήρηση και δεύτερη. Εάν δείτε όλη την περιοχή που έχουμε γύρω μας, τους γειτονές μας, οι προσδοκίες τους δεν είναι τόσο υψηλότερες από αυτές κάποιων άλλων. Μάλιστα, κάποιοι συνεχώς μας λένε δεν είμαστε ακόμα στην ε, περιοχή της διεύρυνσης. Ενώ βάσει της ε, εταιρική σχέσης υπάρχει έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, κάτι άλλο επίσης παραμένει προτεραιότητα. Όσο πιο στενά κοντά θέλει να συνεργαστεί μαζί μας ένας, ε, μια γείτον χώρα, τόσο περισσότερο θα πρέπει να έχει φιλοδοξίες και να πετύχει τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τόσο μεγαλύτερες είναι και δικές μας οι προσδοκίες. Αυτό είναι το καλό με την πολιτική μας, ότι οι εταιρικέ σχέσεις λαμβάνουν πραγματικά δυναμικό χαρακτήρα. Μια άλλη τρίτη γενική παρατήρηση. στις εταιρικέ σχέσεις. Δεν παραβλέπουμε την αντινάμωση των δημοκρατικών θεσμών. Κάποιοι από εσά σχολιάσατε το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βασιζόμενοι και στις δικές σας εκκλήσεις να κάνουμε κι άλλα και να ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς της ε, χώρας με τις οποίες υπάρχει συνεργασία, ιδιαίτερα στα κοινοβούλια τους. Αυτός είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να υπάρχει διάλογος για τις προτεραιότητες της κάθε χώρας. Και αυτό είναι πραγματικά ε, το σπίτι της δημοκρατίας. Εκεί πρέπει να διοργανώνονται ελεύθερες άμεσες εκλογές. Εκεί πρέπει να συζητώνται όλα τα θέματα, αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει και δημοκρατική ορίμανση. Τώρα, να πάω στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Την περασμένη εβδομάδα είχα έρθει στο Στρασβούργο. Νομίζω ωραία τα είπαμε για την Ουκρανία. Δεν θέλω να επαναλάβω όλη εκείνη τη συζήτηση. Είπατε πολλά και εσείς και εγώ εκ μέρους της είπατε εκπροσώπου, της κάθε άστον. Όμως είναι σαφές ποιες είναι οι προσδοκίες μας από την Ουκρανία. Καλωσορίζω το γεγονός ότι και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της χώρας έχουν δημοσιεύσει συστάσεις για να αντιμετωπίσουν τα τρία αυτά βασικά προβλήματα. Παραμένουν τα ζητήματα αυτά ανοιχτά στις σχέσεις με την Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και η επιλεκτική απόδοση δικαιοσύνης, κάτι που στηρίζει και η κάθε και εγώ και το τι κάνει ο πρόεδρος Κόξα και ο κ. Κοσνιεύσκη και νομίζω ότι υπάρχει σαφής κατανόηση των όσων βρίσκονται επιτάπητος, των όσων πρέπει να γίνουν και της απτής προόδου που χρειαζόμαστε για τα ζητήματα αυτά πριν τη Σύνοδο. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη Σύνοδο του Βίλνιους. Πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντική σύνοδος όχι μόνο γιατί υπάρχουν προσδοκίες από τη σύνοδο αυτή, αλλά γιατί μετά από χρόνια συνομιλιών, μελέτης, προσπάθειας ε, συνδυασμού των πολιτικών, προσπαθώντας να μεταμορφώσουμε την περιοχή αυτή που βρισκόταν από το Σοβιετικό καθεστώς, για πρώτη φορά καταφέραμε να εντοπιστούμε όχι μόνο σε λόγια, αλλά σε συγκεκριμένες ανάγκες. Ελπίζω ότι θα υπογραφεί η συμφωνία σύνδεσης και ότι θα πληρούνται, ότι θα δημιουργηθούν μάλλον οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε όλοι μας να αισθανθούμε ότι είμαστε σε θέση να υπογράψουμε τη συμφωνία με την Ουκρανία. Επίσης ελπίζω ότι στο Βίλνιους θα είμαστε σε θέση να βρούμε τρόπο ώστε να σηματοδοτήσουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης συμπεριλαμβανόμενη στη συμμετοχή στην ευρύτερη περιοχή ελεύθερων συναλλαγών με τους τρεις νέους εταίρους, Μολδοβία, Αρμενία και Γεωργία. Ελπίζουμε έτσι να υπάρχει υπογραφή τουλάχιστον αργότερα το 2014. Πολλές οι προσδοκίες λοιπόν από τη Σύνοδο του Βιλνίους. Μίλησα για την ευρωπαϊκή πρόπτικη. Από την άλλη, η ευρωπαϊκή πρόπτικη δεν είναι κάτι που τα κάτι μέλη θα έπρεπε να αισθάνονται ότι υποχρεούνται να το συζητήσουν να κάνουν κάποια βήματα προσέγγισης των ε, γειτόνων μας προς Ανατολές. Είναι σαφές. Όσο περισσότερα αποτελέσματα πετύχουν οι ανατολικοί μα γείτονε για τις μεταρρυθμίσεις, και βάσει των δεσμεύσεων που ανέλαβαν, τόσο περισσότερο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και στο δημοκρατικό καθεστώ θα ε, επιτευθούν και τόσο περισσότερο θα προχωρήσουν προς το μέρο του στα ευρωπαϊκά κράτη. Και τα κράτη-μέλη νομίζω και οι εταίροι μας κατανοούν τους κανόνες του παιχνιδιού. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο πριν το Βίλνιους. Πάντως, όπως και εσείς, σημειώνω ότι εξελίξεις υπάρχουν και στη Μολδαβία και στη Γεωργία. Αναφέρθηκε μια-δυο φορές. Για τη Γεωργία βλέπω να υπάρχει μια κίνηση και μάλιστα προς μια κατεύθυνση επικοδομητική. Αναφέρθηκα ήδη στο διάλογο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Θα πρέπει να δεχτούμε αυτή τη συγκατοίκηση στην εξουσία, αποδεχόμενη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ισχύοντος γεωργιανού συντάγματος και αυτό είναι πραγματικά μια τεράστια πρόκληση. Θα ήταν μια τεράστια πρόκληση ούτως ή άλλως για μια παλιά δημοκρατική χώρα. Ακόμη πιο πολύ για μια χώρα σαν την ε, Γεωργία σε διαδικασία μετάβασης προς τη δημοκρατία. Πριν λίγους μήνες, μαζί με την Κάθη Άστον, ζητήσαμε από τον Τόμας Χάμεμπεργκ, πρώην επίτροπο στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες, να πάει στη Γεωργία, να μιλήσει με τις αρχές, συγκεκριμένα με τον Πρωθυπουργό. Και έχει γίνει πλέον ειδικό σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νομικά και συνταγματικά δικαιο... Ε, ζητήματα συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρίσκεται λοιπόν εκεί ώστε να διευκολύνει τους Γεωργιανούς και την κυβέρνησή τους να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Όπως έκαναν και στην περίοδο πρώτων εκλογών με τις τότε υποσχέσεις τους. Θέλουμε να πετύχουν αποτελέσματα βάσει των κοινών προτύπων των κοινών αρχών που έχουμε καθορίσει. Να ενισχύσουν το κράτος δικαίου και όχι να το αποδυναμώσουν. Επίσης βρίσκεται εκεί ώστε να διευκολύνει και τον πρόεδρο της χώρας και τον πρωθυπουργό να έχουν καλύτερη επικοινωνία ήταν δυσχερέστερη προηγουμένως. Ελπίζω ότι ο κ. Χάμπεργκ θα έχει τη στήριξη του Κοινοβουλίου και εγώ θα καταφέρω να μιλήσω με τον πρόεδρο Μπροκ να δούμε πώς και εκείνος θα μπορούσε να σας μιλήσει για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα της Γεωργίας της γεωργίας που πλησιάζει διαρκώς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το αντίστροφο. Επίσης, ε, τέθηκαν μια σειρά από ερωτήσεις ως προς τον Νότο και τους γειτονέ μας στον Νότο. Να ξεκινήσω με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Αναλάβαμε τη δέσμευση να στηρίξουμε το Ίδρυμα. Και αυτό γίνεται δημοσιονομικός. Είμαστε αποφασισμένοι και εγώ και ο Έλμαρ Μπροκ ότι και στο μέλλον θα παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση αυτή. Δεν θα υπάρξουν προσχήματα από την πλευρά μας για να ανακοπεί η στήριξη προς το έλλειμμα αυτό. Καλείται να καλύψει και να στην περίπτωση μη κυβερνητικών οργανώσεων ή πολιτικών κομμάτων που για διαφορετικούς ε, υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή στήριξη. Μια από τις χώρες αυτές θα είναι η Λιβύη. Προανέφερα και το ίδιο έκανε και η κυρία Μπούθκουρτ ότι υπάρχουν προβλήματα στην πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ευρωπαϊκή στήριξη. Πάντω οι ίδιοι οργανώσεις κοινωνία των πολιτών στηρίζονται στη Λιβύη από εμάς. Υπάρχουν προγράμματα των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη τη κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Λιβύη. Αλλά περιμένουμε περισσότερα ακριβώ με την ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο για την Δημοκρατία. Ο κ. Μίλαν Μόρ ζήτησε για ρώτησε να μάθει τι γίνεται με το Μαρόκο και τις υπηρεσίες, το κατά πόσον προχωρήσαμε με το DCFTA. Επίσης για τη Συρία τέθηκαν ερωτήσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να στηρίξουμε την δημοκρατία στη Συρία αλλά και εκτός Συρίας. Μάλιστα, συγκεκριμένα τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει μια ειδική έκθεση για τους φοιτητέ και νέους. Θα τους φέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα σχολεία μας και στα πανεπιστήμια μας. Θέλουμε να σπουδάσουν. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην εξομάλυνση της κατάστασης στη Συρία. Η Συρία είναι ένα ζήτημα περίπλοκο. Το συζητήσαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Να αποκωδικοποιήσουμε λίγο αυτά που υπόθηκαν στο Στρασβούργο τώρα. Πρέπει να είμαστε κάπως πιο δημιουργικοί και εφάνταστοι στη, τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και επιπτώσεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Πρέπει να μεταφράζονται σε μια σαφή έκκληση προς τους πολιτικούς να βρουν ξεκάθαρες πολιτικές λύσεις, αλλά καλούν τα γεγονότα αυτά και μας να υπερβούμε την αρχή της απλής ανθρωπιστικής στήριξης. Αυτό ήδη φάνηκε με τα πρώτα βήματα που έγιναν στο Λίβανο πριν από 15 μέρες επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο για τις ανάγκες των προσφύγων, αλλά και τις ανάγκες της κοινότητας των ε, φιλοξενούντων, υποδοχής. Έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους τους ανθρώπους αυτούς. Και θα πρέπει και τα κρατη μέλη να αναλάβουν ένα μερίδιο της ευθύνης. του βάρους να βρουν λύσεις σε αυτό το σημαντικό άμεσο πρόβλημα των, των προσφύγων. Είναι παράγοντας πίεσης και χωρίς επιπλέον στήριξη από τη δική μας την πλευρά θα υπάρχουν επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή ως προς την ασφάλειά της. η συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπα αντιπρόεδρο της Επιτροπής και του αντιπρόεδρου μάλλον της Επιτροπής είναι εξαιρετική και σε προσωπικό επίπεδο και επαγγελματικά. Και με μένα συνεργάζεται στενά και όπως ξέρετε και με, τους, ε, με τον Πρωθυπουργό της Σερβίας του Κωσυφοπεδίου έχει συνομιλίε για να βρεθούν λύσει και στα προβλήματα τα πολύ συγκεκριμένα που υπάρχουν, όπω το βόρειο τμήμα τη χώρα. Συζητάμε για τι πολιτικέ προτεραιότητές μα, για τι απόψει μα για το πώ να αξιοποιούνται τα διάφορα εργαλεία. Δεν υπάρχει επικάλυψη στι δραστηριότητέ μα. Στηρίζουμε ο ένα τον άλλο, ώστε να γίνεται η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη. Σε άλλες περιπτώσεις είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα παραδείγματα της αρχής του More for More, του περισσότερες προσπάθειες για περισσότερα αποτελέσματα. Τώρα συζητούμε για το νέο αυτό εργαλείο στήριξης των γειτονικών μας χωρών. Ξέρετε ότι αυτό το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο θέλουμε να διέπεται από την αρχή more for more και αυτή η αρχή να ενσωματώνεται στην ε, ουσία της βοήθειας που προσφέρουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε δύο πράγματα. Να είμαστε πιο ευέλικτοι και να στηρίζουμε τις ε, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στις γειτονικές χώρες. Δεύτερον, έχασα τον ήρμό. Η ώρα έχει περάσει. Αυτός μπορεί να είναι ο λόγος. Θα επανέλθω. Προς το τέλος. Υπάρχουν σαφείς ε, δείκτες συγκριτικοί για το πώς μπορούμε εδώ να πετύχουμε αποτελέσματα. Ρωτήσατε για την αρχή More for More και το τι γίνεται με την Αίγυπτο. Το ρωτήσατε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και λάβατε σαφείς ε, δηλώσεις δέσμευσης από την πλευρά της ΥΠΑ εκπροσώπου. Εγώ θα συμφωνήσω με όσα είπε. αυτό που είπε η κυρία Νέτ για το Μαρόκο και τη Σαχάρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι καθώς εμβαθύνουμε και ενδυναμώνουμε τις σχέσεις συνεργασίας μας, ότι οι εταίροι μας μπορούν να είναι ειλικρινέστεροι στην επικοινωνία μας. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν ταμπού στις συνομιλίες. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι δεν θα υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχουν άτομα ή ομάδες ε, εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άλλων θεσμικών οργάνων, καλοπροαίρετες ε, αποστολές, επισκέψεις που πρέπει να επισκεφθούν ε, σημεία, διαφορετικά σημεία της χώρας από τους εταίρους μας. Τέτοια στάση περιμένουμε και από το Μαρόκο πιο συγκεκριμένα. Είναι μια χώρα με την οποία έχουμε προνομιακή εταιρική σχέση. Τώρα τις δικές μας τις μέρημνες πώς να τις περάσουμε και να τις κάνουμε κατανοητές στο Αζερμπαϊτζάν. η κυρία Λούνατσεκ το έθεσε αυτό. Στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Πακού, στον Πακού μάλλον, στις αρχές Μαΐου, θα είμαι πάλι εκεί, είχα μια σειρά από επαφές για να καταρτήσουμε με την είπατε εκπρόσωπο μια κοινή προσέγγιση και να δούμε a closer connection between uh, making sure that we have a number of the concerns and making sure that we have not only concerns but we have also uh, an ideas uh, how to uh, tackle